Dear colleagues, dear members. Συνάδελφοι, αγαπητοί, αγαπητά μέλη του Ευρωκοινοβουλίου, μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων, κύριε Βόλσλένερ, αγαπητή Αντιπρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κύριε Γενική Διευθυντά, αγαπητοί προσκεκλημένοι, είναι μεγάλη μου χαρά που κηρύσω την έναρξη της συνεδρίασης της Διευκοινοβουλευτικής Επιτροπής για το θέμα της κοινωνικής ένταξης των ε, Ρωμά και της καταπολέμησης αθηγανοφοβίας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συγκεκριμένα η Επιτροπή Θεμελιωδών Δικαιωμάτων αποδίδει μεγάλη σημασία στο ζήτημα αυτό, όπως αποδεικνύεται και από το ψήφισμα της 25ης Οκτωβρίου 2017 για τα θεμελιώδη δικαιώματα όσον αφορά την ένταξη των Ρωμά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την καταπολέμηση του αντιαθηγανισμού. Το ψήφισμα αυτό υπογραμμίζει ότι παρά τις προσπάθειες και τις χρηματοδοτικές ε, ενισχύσεις που έχουν επενδυθεί, καθώς και τα πολυάριθμα ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα και ταμεία που έχουν ε, προσπαθήσει να δώσουν απάντηση στα προβλήματα των κοινοτήτων των Ρωμά, οι συνθήκες διαβίωσης αυτών των κοινοτήτων δεν έχουν βελτιωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια και η ένταξη δεν έχει προχωρήσει με την απαραίτητη ταχύτητα. Προκειμένου να καταπολεμηθεί η περιφερειοποίηση... οι διακρίσει και οι αποκλήσεις εναντίον των Ρωμά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το ψήφισμα αυτό περιείχε συγκεκριμένε εστάσει που απευθύνονταν στα κράτη-μέλη, όπως είναι η πλήρης εφαρμογή των εθνικών στρατηγικών τους για την ένταξη των Ρωμά, καθώς και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να αναβαθμίσει το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις, στρατηγικές, για τις εθνικές στρατηγικές για την ένταξη των Ρωμά έπειτα από το 2020 προκειμένου να ε, μια βελτιωμένη, επικαιροποιημένη και πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση. Η σημερινή μας εκδήλωση λοιπόν αποτελεί ευκαιρία ένα χρόνο μετά να γίνει ένας απολογισμός σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο για αυτό το σημαντικό θέμα σε συνεργασία με τους συναδέλφους μας από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Όσον αφορά τη διερμηνία, σημειώστε ότι σήμερα έχουμε διερμηνία σε όλες τις επίσημες ε, γλώσσες Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός από τα δανέζικα, τα λετονικά, τα μαλτέζικα και τα ιρλανδικά. Το πρόγραμμα σήμερα περιλαμβάνει μια σειρά από πολύ σημαντικούς ομιλητές. Θέλω να καλωσορίσω εδώ την κυρία Γιάροκα, αντιπρόεδρο του Κοινοβουλίου, την κυρία Ντόρι Βόλφ-Λένερ, που είναι επικεφαλής του τμήματος της ε, καγκελαρία της, μόνιμη ε, μόνιμης τη της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και την Τίνα Άστολα, που είναι Γενική Διευθύντρια για ζητήματα δικαιοσύνης και καταναλωτών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήθελα να δώσω το λόγο τον, ε, στην κυρία Λίβια Γιάροκα, αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ως πρώτη ομιλήτρια της εναρκτήριας αυτής εκδήλωσης για τη σημερινή μας διακοινοβουλευτική συνάντηση. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστώ που ήρθατε σε αυτή τη συνεδρίαση. Είμαι πολύ ικανοποιημένη και σας καλωσορίζω όλους στο όνομα του κυρίου Ταγιάννη. Το Κοινοβούλιο σε ό,τι αφορά το θέμα των Ρωμά ήταν πρωτοπόρος. Ο κύριος Μπούζεκ πριν από λίγα χρόνια κατάλαβε ότι αν δεν ενωθούμε, η Κομισιόν δεν πρόκειται να μας πάρει στα σοβαρά. Γι' αυτό λοιπόν πήγε με τον κύριο Μπαρόζο σε μια άτυπη συνεδρίαση για να του εξηγήσει πόσο σημαντικό είναι το θέμα. Χάρη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στις προσπάθειές του, και στις προσπάθειες όλων των πολιτικών ομάδων που υποστήριξαν το ψήφισμα για τους Ρωμά, μπόρεσε και η Ουγγρική κυβέρνηση το 2011 για να μπόρεσε να περάσει το κείμενο αυτό στο Συμβούλιο. Λέω ότι μπόρεσε, ότι ήταν πιο εύκολο, γιατί υπήρχαν πολλά επιχειρήματα τότε το 2011 για την οικονομική ε, ένταξη ε, ήταν πέντε φορές πιο εύκολο να εντάξουμε τους στοχούς ε, στις κοινωνίες μας. Ε, γιατί καταλαβαίνουμε ότι αν δεν κάνουμε τίποτα για τους Ρωμά, αν δεν εντάξουμε τις φτωχές Ρωμά στην αγορά εργασίας, θα μας κοστίσει πολύ στο μέλλον, μέχρι το 2050. Ε, εάν δεν αντιμετωπίσουμε τα θέματα εργασίας και απασχόλησής τους, η, στρατηγική, η ευρωπαϊκή στρατηγική πλαίσιο δεν θα αρκέσει. Λίγα χρόνια μετά η κυρία Σοράγια Πόστ ξανά ενέκυψε επί του θέματος και κοίταξε ότι η εφαρμογή της οδηγίας για τα δικαιώματα δεν είναι ικανοποιητική και υποσκάπτει την επιτυχία και στους άλλους τομείς. Το 2010 οι, όσοι ζούσαν σε φτώχεια ε, σε όλη την Ευρώπη ε, ήταν 40 με 50 εκατομμύρια. Δημιουργήθηκε από την Κομισιόν μία task force για τους Ρωμά και ζητήσαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να χαρτογραφήσει την κατάσταση και τότε είδαμε ότι το 50% των φτωχών στην Ευρώπη είναι προέλευση Ρωμά και όλοι οι υπόλοιποι οι οποίοι ζουν γύρω-γύρω ε, και δεν είναι Ρωμά είναι στην ίδια κατάσταση. Το έγγραφο αυτό είπε ότι από τα 43 άτομα 10 εκατομμύρια είναι Ρωμά. Ε, σήμερα εξακολουθούμε να έχουμε 8 με 10 εκατομμύρια φτωχούς Ρωμά. Χάρη σε αυτό το πλαίσιο έχουμε περισσότερες δράσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλοι οι εθνικοί φορείς προσπαθούν να υλοποιήσουν τις υποσχέσεις της Κομισιόν, του Κοινοβουλίου και των, και των κρατών μελών που ανέρχονται στην ε, εποχή του 2011. Παρότι υπάρχουν πολλά κονδύλια, παρότι υπάρχει ένας τεράστιος μηχανισμός ε, στο εσωτερικό της Κομισιόν και στο εσωτερικό των ε, κρατών μελών για τη μείωση της στόχιας των Ρώμα, παρόλα αυτά οι χώρες αυτές δεν χρησιμοποιούν αρκετά τα διαφορετικά ταμεία και το κοινωνικό ταμείο αρκετά και η συμμετοχή των ιδίων των Ρωμά δεν ήταν ικανοποιητική. Ίσως γι' αυτό λοιπόν εξηγείται ότι η απομόνωσή τους τα τελευταία πέντε χρόνια ε, δεν έχει, το θέμα της απομόνωσής τους δεν έχει βελτιωθεί γιατί έχουμε ασχοληθεί κυρίως με τα οικονομικά θέματα. Δεν υπάρχει αρκετή πρόοδος. Το πρόβλημα δεν είναι ότι οι Ρώμα δεν εμπλέκονται στα προγράμματα, αλλά με βάση την έρευνα έχουμε καταλήξει ότι τα project, τα έργα αυτά, τα οποία ε, συμμετέχουν, στα οποία συμμετέχουν οι ίδιοι Ρωμά και κυρίως οι Ρωμά που ζουν στην περιοχή, είναι πολύ πιο βιώσιμα. Εκείνη την εποχή, λοιπόν, για, ε, με, μου είπαν στην συνάδελφοι γιατί να μην βάλει τον αθηγανισμό περισσότερο μέσα στα κείμενα. Έχουμε τελικά μία οδηγία η οποία λαμβάνει υπόψη της το θέμα της απομόνωσης των Ρωμά. Ε, το θέμα είναι να εφαρμοστεί αυτή η οδηγία. Η Σοράγια Πόστ έγραψε μία έκθεση που δείχνει ότι και στην οδηγία της Κομισιόν για τους Ρωμά θα πρέπει να γίνουν συγκεκριμένα πράγματα και να μπουν πολλά από τα στοιχεία της έκθεσης Σοράγια Post ε, για να αλλάξει η κατάσταση των Ρωμά. Οι γονεί μου, από την προσωπική μου εμπειρία, ε, σας λέω ότι έκαναν πολλά για να ε, εξασφαλίσουν ότι δεν καταπατώνται τα δικαιώματά μου, αλλά όταν πήγαινα στο σπίτι και τους έλεγα ότι πέφτω θύμα ε, διακρίσεων επειδή είμαι τσιγκάνα, ε, μου έλεγαν ότι θα το πολεμήσει αυτό πώς γίνεις, όταν γίνεις η καλύτερη. Πρέπει να αριστεύσεις. Εγώ τι κατάλαβα, ότι πρέπει να πολεμήσουμε. Ε, ο πατέρας μου μου εστάλαξε και η μητέρα μου μου εστάλαξε αυτές τις ιδέες. Ε, πολέμησε ο πατέρας μου και η μητέρα μου για να μπω σε κανονικό σχολείο, όχι ειδικό σχολείο. Επίσης και για την αγορά εργασία. εργασίας μου είπε ότι θα ανταγωνιστώ με τους άλλους αν έχω τα ίδια τουλάχιστον προσόντα. Ε, να το μήνυμα της για την ε, καταπολέμηση των διακρίσεων και είναι πολύ σημαντικό όλα αυτά που είχαμε πει τότε πριν από 7 χρόνια, ε, καλά σχολεία, παιδική σταθμή, νηπιαγωγία, ε, καλές δουλειέ, καλά εργοστάσια κτλ. Τίποτα από αυτά δεν έχει νόημα εάν δεν εξασφαλίσουμε την αποφυγή των διακρίσεων. Τίποτα δεν θα αλλάξει εάν δεν έχεις αυτά τα εργαλεία που θα σε βοηθήσουν για να αλλάξεις την εκπαίδευση, τις συνθήκες διαβίωσης, την εκπαίδευση. Όχι μόνο τα θεμελιώδη δικαιώματα, όχι μόνο να αποφύγεις τις διακρίσεις, αλλά να εξασφαλίσεις παράλληλα ότι τα project είναι αποτελεσματικά, τα λεφτά δεν εξασφαλίζονται, ότι οι ίδιοι οι Ρωμά εμπλέκονται σε αυτά τα έργα που τους αφορούν από την αρχή ως το τέλος. Όλοι οι ευρωβουλευτές ε, του Κοινοβουλίου ενωμένοι και κυρίως αυτοί που είναι προέλευσης Ρωμά ε, αποφάσισαν να βοηθήσουν την Κομισιόν για τον σχεδιασμό του επόμενου πουδουπού, του επόμενου πολυμερού δημοσιονομικού πλαισίου, πολίτου δημοσιονομικού πλαισίου. Η Σοράγια είναι υπεύθυνη για τα θέματα των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ο κ. Φανή Τελρόι εξετάζει τη χρηματοδότηση από τα διαρθωτικά ταμεία. Εγώ στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων προσπαθώ να δω τι γίνεται με τον επόμενο προπολογισμό. Τι βρήκαμε λοιπόν ε, ετοιμάζοντα την επόμενη έκθεση. Ότι τα λεφτά των τελευταίων 7 ετών δεν χρησιμοποιήθηκαν α, έτσι όπως πιστεύαμε όλοι ότι θα χρησιμοποιούνταν. Το καλό είναι ότι έχουμε πολλά λεφτά ακόμα που δεν έχουμε εξοδέψει, τα κράτη-μέλη δεν έχουν εξοδέψει για να τα χρησιμοποιήσουν για τους Ρωμά μέχρι το τέλος του 2020 η Κομισιόν θα πρέπει να πει στα κρατη που δεν έχουν ξοδέψει ε, λεφτά για να μην τα ξαναστείλουν πίσω στο γενικό προπολογισμό, να του πει χρησιμοποιήστε τα, ξοδέψτε τα και χρησιμοποιήστε τα για αυτό το σκοπό για τον οποίο σχεδιάστηκαν. Πριν περάσουμε στα επό... στην επόμενη εφταετία, τον επόμενο προγραμματισμό δηλαδή τη επόμενη εφταετία, σε αυτή τη φάση ήδη, τώρα που μπορούμε να εξασφαλίσουμε από την Κομισιόν ότι η οδηγία θα πάρει τη μορφή αυτή που πρέπει να πάρει για την ε, προάσπιση των πιο φτωχών. Θα πρέπει λοιπόν αυτή τη στιγμή να υποφεληθούμε και από την Αυστριακή Προεδρία και από τους μήνες που έχουμε μέχρι το τέλος της θητείας μας, ούτω ώστε να γίνει γνωστό ότι υπάρχουν πολλά λεφτά ακόμα που δεν έχουν δαπανηθεί και μπορούν να δαπανίσουν τα κράτη-μέλη υπέρ των Ρωμά. Θα πρέπει λοιπόν να βασιστούμε στις ε, εκθέσεις που αφορούν τα έξυπνα χωριά, την ψηφιοποίηση της Ευρώπης, τη γεωργία, την κοινή γεωργική πολιτική. Μόνο η έκθεση Σοράγια ε, είναι για τους Ρωμά. Ε, είναι, υπάρχει έκθεση για, τους, για τον καρκίνο. γιατί οι Ρωμά είναι τα χειρότερα θύματα έχουν περισσότερους καρκίνους από το μέσο ε, Ευρωπαίο, έχουν ε, τα περισσότερα δεινά γενικά, όλα αυτά είναι περίεργα. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να κάνουμε, να χρησιμοποιήσουμε τα λεφτά, έχουμε τα εργαλεία, ας χρησιμοποιήσουμε αυτή την έκθεση και τις άλλες αυτά εκθέσεις που υπερψηφίστηκαν από το Κοινοβούλιο ήδη. Για να πιέσουμε να περάσει ε, το ψήφισμα τον επόμενο βήμα, ούτω ώστε να βοηθήσουμε την Αυστριακή Προεδρία να κάνει αυτά που πρέπει για να βοηθήσει και η Αυστριακή Προεδρία την Κομισιόν να κάνει το έργο της. Έχουμε την ενδιάμεση αξιολόγηση τώρα. Πέρυσι είχαμε μια πλατιά διαβούλευση με όλους τους Ρωμά και με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών χάρη στην προετοιμασία αυτής της έκθεσης. Ξέρουμε τι θέλουν πλέον οι Ρωμά, ξέρουμε τι θέλει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όλοι είναι ενωμένοι. 90% των ευρωβουλευτών ψήφισαν υπέρ της έκθεσης ώρα για Post και υπέρ της δικής μου έκθεσης. Δεν υπάρχει θέμα πολιτικό. Ας υλοποιήσουμε τις προσπάθειές μας. Υπάρχουν και τα λεφτά. Είναι πολύ δύσκολο οι Ρουμάνοι τον επόμενο μισό χρόνο να κάνουν κάτι. Γιατί αν δεν, και επιπλέον, αν δεν κάνει κάτι η Ρουμανική Προεδρία, θα κάνει τίποτα κανένας ε, μέχρι την επόμενη επιτροπή. Εάν δεν κάνουμε κάτι λοιπόν του επόμενου δύο μήνε θα χάσουν μια τεράστια ευκαιρία, μια φοβερή χρονική στιγμή. Σα ζητώ όλου να βοηθήσετε το Κοινοβούλιο, τα δικά σα εθνικά κοινοβούλια να σταθούν στο πλευρό του Ευρωκοινοβουλίου, γιατί και στα εθνικά κοινοβούλια συμβαίνει, γράφεται η ιστορία. Εσεί θα πάτε πίσω στα κοινοβούλια σα. Όλοι έρχεστε, έρχεστε από διαφορετικέ περιφέρειες στη χώρα σα. Ξέρετε που είναι η φτωχή. Και ξέρετε ότι τα τελευταία 7 χρόνια γίνανε κάποια έργα Ξέρετε ποια είναι αυτά τα έργα. Ξέρετε τι λείπει επίσης στη δική σας περιοχή. Επομένως, ας επιστρέψουμε σε επίπεδο εθνικών κοινοβουλίων. Γιατί με αυτόν τον τρόπο ξέρουμε πολύ καλά ποια είναι η κατάσταση στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε μια μικρή χρονική περίοδο, αλλά την έχουμε στη διάθεσή μας. Τις επόμενες εβδομάδες ε, υποβάλλετε προτάσεις για αυτή τη νέα στρατηγική των Ρωμά μέσω των πρεσβειών σας, λέει η μιλήτρια. Σας ευχαριστώ πολύ. Μιλάμε για τη νέα περίοδο πάντα 2020-2027. Thank you very much to our... Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ που επισημάνατε πολλά και συγκεκριμένα πράγματα για το θέμα των ΟΡΜΑ και πάνω απ' όλα να δείξατε ότι είναι πολύ σημαντική συνεργασία ε, από το ευρωπαϊκό μέχρι το εθνικό επίπεδο, γιατί η πραγματική δουλειά γίνεται πάντα και σε εθνικό, αλλά ακόμα και σε τοπικό επίπεδο. Είναι απαραίτητη λοιπόν αυτή η συνεργασία. Θα δώσουμε λοιπόν απευθεία το λόγο στην δόκτωρα Ντόρι Βολσένερ από τη Γερμανική, συγγνώμη, Αυστριακή Προεδρία. Ευχαριστώ κυρίε και κύριοι, ευχαριστώ για την πρόσκληση που μου απευθύνεται. Η Αυστριακή Προεδρία χαιρετίζει την διακοινοβουλευτική, ε, συνάντηση τη Διακοινοβουλευτική Επιτροπή ε, για τι ε, πτυχέ θεμελιωδών δικαιωμάτων σε ό,τι αφορά τη συμπερίληψη των Ρωμά. Ε, ε, Ευχαριστούμε και την Επιτροπή για την ε, διοργάνωση αυτή τη συνεδρίαση. Όπω προτείνει και προκύπτει και από την ημερήσια διάταξη, η καταπολέμηση του αντιθεγενισμού ε, εντοπίζεται ω μία από τι βασικέ τη επιτυχίε για την συμπερίληψη των Ρωμά. Το Συμβούλιο ε, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην καταπολέμηση των διακρίσεων και των προκαταλήψεων κατά των Ρωμά. Ο αντιαθεγκανισμός είναι βασική αιτία του κοινωνικού αποκλεισμού των Ρωμά. Ήδη έχουν γίνει σημαντικές ε, προσπάθειες για την αναγνώριση του φαινομένου αυτού στην ενδιάμεση αναθεώρηση της στρατηγικής μέχρι το 2020. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντοπίζει την ανάγκη ενίσχυσης και ανάδειξη, ε, του σημείου Εστίαση κατά του αντιθεκανισμού και των διακρίσεων και σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο. Η καταπολέμηση του αντιαθηγανισμού είναι μία από τις βασικές προτεραιότητες της ε, ε, επικαιροποιημένης αυστριακής στρατηγικής για Το Συμβούλιο ΕΠΣΚΟ πρόσφατα υιοθέτησε συστάσεις για το ζήτημα αυτό με σκοπό την προώθηση Τη υλοποίηση των εθνικών στρατηγικών και της ε, υπερεθνικής συνεργασία. Επίσης, η σύσταση αναδεικνύει την ανάγκη καταπολέμησης του αντιαθηγανισμού και παροτρύνει τα κράτη-μέλη ε, να αναλάβουν και δράσεις ε, θετικών διακρίσεων, αν θέλετε. Από τη Βιέννη προέκυψε ότι ο αντιθυγανισμός είναι βασικός μοχλός κοινωνικού αποκλεισμού που υπονομεύει την κοινωνική ένταξη των Ρωμά. Υπάρχει και το πλαίσιο για μετά το 2020 και τα, συμβούλ... και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 8 Δεκεμβρίου 2016. Και σε αυτό το πλαίσιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πλαίσιο για την συμπερίληψη των Ρωμά μετά το 2020 θα διοργανώσουμε μία ε, διάσκεψη ε, στις 27 Νοεμβρίου ακριβώς για την υλοποίηση αυτής της στρατηγικής. Σκοπός της συνδιάσκεψη είναι να καταλήξει σε σαφείς συστάσεις για το πώς ε, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο του αντιαθυγενισμού. Με τη συνδιάσκεψη θα συγκεντρώσουμε διάφορα ενδιαφέροντα μέρη, εκπροσώπους ε, διεθνών οργανισμών, ευρωπαϊκών οργανισμών και φορέων, ε, εθνικών σημείων επαφής, εκπροσώπους και υποψηφίων χωρών που είναι κάτι σημαντικό, εκπροσώπους τοπικών και περιφερειακών αρχών αλλά και εκπροσώπου ε, οργανώσεων ε, τη κοινωνία των πολιτών και του ακαδημαϊκού χώρου. Η Αυστριακή Προεδρία θέλει να διευκολύνει ε, και να επιτρέψει μια ανοιχτή και ευρεία διαδικασία διαβουλεύσεων για την αντιμετώπιση του αντιαφηγανισμού. Και αυτό θα καθορίσει και την επιτυχία των μελλοντικών προσπαθειών συμπερίληψη κοινωνική ένταξη των Ρωμά και τη αποτελεσματικότητά του. Ευχαριστώ. Thank you very... Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα μπορούμε απευθεία να περάσουμε στην κυρία Τίνα Άστολα, Γενική Διευθύντρια Δικαιοσύνη και Καταναλωτών των την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρακαλώ, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι. Θα ήθελα και εγώ να ξεκινήσω ευχαριστώντα θερμότατα την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ που πήρε την πρωτοβουλία για αυτή την διακοινοβουλευτική συνάντηση για τα θεμελιώδη δικαιώματα, την ένταξη των Ρωμά και την καταπολέμηση του αντιαθηκανισμού. Εμείς ε, στην Κομισιόν θεωρούμε ότι είναι πολύ επίκαιρη η συνεδρίαση αυτή γιατί βρισκόμαστε στη φάση οριστικοποίησης της βάθος αξιολόγησης του πλαισίου για τους Ρωμά. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης την Αντιπρόεδρο Γιαρόκα για την συνολική συμβολή της στην ε, περαιτέρω ανάπτυξη της ευρωπαϊκής πολιτικής για τους Ρωμά και ιδίως στην ανάπτυξη των εθνικών και ευρωπαϊκών στρατηγικών. Και φυσικά να ευχαριστήσω και την κυρία Σοράγια Πόστ για την εξαιρετικά φιλόδοξη έκθεση που συνέτεξε για την καταπολέμηση του αντιαθηκανισμού. Αποτέλεσαν ε, όλα αυτά πολύ μεγάλη συμβολή και στην ενδιάμεση αξιολόγηση και στον προβληματισμό για την προσέγγιση που θα υιοθετηθεί μετά το 2020. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω όλους όσοι βρίσκεστε σήμερα εδώ και από τις θέσεις σας ε, έχετε συμβάλει στην ε, ανάπτυξη και τη βελτίωση των πολιτικών μας. Είμαστε όλοι σύμμαχοι σε αυτή την προσπάθεια για να καταστήσουμε πραγματικότητα την ένταξη των Ρωμά. Όπως γνωρίζετε οι περισσότεροι από εσάς, η αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Πλαισίου για, το, για τις Εθνικές Στρατηγικές ένταξεις των Ρωμά πρόκειται να αριστικοποιηθεί σύντομα. Η, η ανακοίνωση του 2018 αντικατοπτρίζει τις βασικές ε, ε, σκέψεις στις οποίες έχουμε καταλήξει και θα δημοσιευτεί το Νοέμβριο, στις αρχές Νοεμβρίου. Επίσης, ε, αναμένουμε την δημοσίευση της εξωτερικής έκθεσης που ανατέθηκε και που καλύπτει το 2011 με 2017 και αξιολογεί την, ε, τον οργανωμένο χαρακτήρα, την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα, τον δίκαιο χαρακτήρα, τον συντονισμό, τη βιωσιμότητα και την προστιθέμενη αξία του πλαισίου που εφαρμόστηκε. Αναλύει λοιπόν τις, ε, τα δυνατά και τα δύναμα σημεία του πλαισίου και θα καταλήξει σε συγκεκριμένες συστάσεις για το πλαίσιο μετά το 2020. Κάναμε πραγματικά πολύ μεγάλη προσπάθεια για να καταλήξουμε σε μια ειλικρινή και διαφανή αξιολόγηση ώστε πραγματικά να μπορέσουμε να συλλέξουμε στοιχεία και ενδείξεις και να προχωρήσουμε στο έργο μας παρατέρα. Η σημερινή μου τοποθέτηση θα βασιστεί σε αυτά τα προκαταρκτικά πορίσματα της μελέτης, τα οποία καταδεικνύουν την ανάγκη να υπάρχει ενισχυμένη προσπάθεια ε, στην καταπολέμηση του αντιαθηγανισμού που θα συμβαδίζει με κοινωνικο-οικονομική ένταξη των Ρωμά. Δυστυχώς πρέπει, ε, μάλλον, πρέπει η κοινωνική ένταξη να συμβαδίζει, από, ε, να συμβαδίζει με παρακολούθηση από θεσμικούς φορείς και ε, ε, με συνεργασία της κοινωνίας των πολιτών. Η αξιολόγηση καταλήγει ότι οι στόχοι θα μπορούσαν να είχαν, πιο, θα μπορούσαν να είχαν υπάρξει πιο ε, φιλόδοξοι. Πρέπει να καταπολεμηθούν οι διακρίσεις κατά τον ε, Ρωμά και να δοθούν καλύτερες, πιο εξειδικευμένε απαντήσεις εντός υποομάδων της κοινότητας των Ρωμά, των νέων Ρωμά, των παιδιών των Ρωμά, των γυναικών Ρωμά. Η αξιολόγηση καταδεικνύει ότι χρειάζεται πιο στοχευμένη προσέγγιση στην ε, μη διακριτική μεταχείριση και την καταπολέμηση του αντιαθηγανισμού. Και αυτό ανεδείχθηκε στις συζητήσεις που έγιναν την προηγούμενη εβδομάδα στην Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για την Ένταξη των Ρωμά, στην οποία ξέρω ότι κάποιοι από εσά συμμετείχατε, που επικεντρώθηκε στι αδικίες όσον αφορά την ε, πρόσβαση των Ρωμά στη στέγαση και τι υγειονομικέ υπηρεσίε. Ο αντιαθηκανισμός ε, ανεδείχθηκε ως βασικός ε, λόγος για τον οποίο πολλοί Ρωμά δεν έχουν πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες. Θεωρώ ότι οι συζητήσεις που έγιναν στην πλατφόρμα είναι πάρα πολύ σημαντικές και μας δείχνουν και πώς πρέπει να προχωρήσουμε από εδώ και πέρα ε, και πώς πρέπει βεβαίως και να συνεργαστούμε. Αυτά βοήθησαν και τροφοδότησαν και τις συζητήσεις μας για την περίοδο μετά το 2020, όπως και η σημερινή εκδήλωση, η οποία επίσης θα ληφθεί υπόψη στο σχεδιασμό μας για την περίοδο μετά το 2020 και βεβαίως βασιζόμαστε πάντοτε και στη δική συμβολή και υποστήριξη. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Κάποιες φορές όταν μιλάμε για τον αντιαθηγανισμό γνωρίζω ότι κάποιοι συμπολίτε μας μας λένε ναι αλλά ξέρετε υπάρχουν πολλά στρώματα που θεωρούν ότι δεν είναι τμήμα της κοινωνίας ή που αισθάνονται περιθωριοποιημένοι. Νομίζω όμως ότι οι Ρωμά είναι εκείνοι που όχι μόνο έχουν υποστεί διακρίσεις στη διάρκεια αιώνων, αλλά μιλάμε για διακρίσεις βία, περιθωριοποίηση, αποκλεισμό κοινωνικό, κάποιες φορές ακόμη και δολοφονίες. Και έχοντας υπόψη ότι οι διακρίσεις ε, συνεχίζονται μέχρι και σήμερα, στον 21ο αιώνα, νομίζω ότι αυτό από μόνο του δείχνει ότι πρέπει επιτέλους να αναλυφθεί ε, δράση, όχι μόνο με τη μορφή ε, ψηφισμάτων ή ακόμα και χρηματοδοτική στήριξη, αλλά να περάσουμε πραγματικά σε πραγματικές δράσεις. Γι' αυτό και θα ήθελα να ευχαριστήσω ευχαριστήσω τις, τις ε, τρεις ομιλήτριες μας για τις ομιλίες τους και για τις παρεμβάσεις τους και για την παρουσία τους. Λοιπόν, περνάμε στο επόμενο κομμάτι της ε, συνεδρίασής μας. Δεν βλέπω να υπάρχουν ερωτήσεις, οπότε περνάμε στο επόμενο πάνελ. Προτού το κάνω όμως αυτό, κανονικά θα πρέπει να με είχε αντικαταστήσει ένα συνάδελφο. Αυτό που μπορώ να κάνω εγώ τώρα είναι να ανακοινώσω ότι η συνεδρίασή μας θα διαρκέσει έως τις 6 το απόγευμα και θέλω να ξεκαθαρίσω ότι οι διερμηνείς θα μας εγκαταλείψουν ακριβώς στις 6, τελειώνει το ωράριό τους. Έχετε το αυτό υπόψη σας. Πρέπει να γίνονται σεβαστά και τα δικαιώματα των εργαζομένων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε τις συζητήσεις μας μετά τις 6. Λοιπόν, Τούτων λεχθέντων να ξαναευχαριστήσω βεβαίως όλε τι ομιλήτρε που είναι εδώ και περνάμε στο επόμενο πάνελ. Νομίζω λοιπόν ότι δεν χρειάζεται να ε, χάσουμε άλλο χρόνο. Ε, ξαναλέω ότι διερμηνία έχουμε στη διάθεσή μας έως τις 6 το απόγευμα. Προτού με αντικαταστήσει συνάδελφος, θα ήθελα να ξεκινήσω να κηρύξω την έναρξη της πρώτης συνεδρίασης που αφορά το θέμα της ένταξης των Ρωμά και τα κοινωνικά, τα θεμελιώδη δικαιώματα. Πρωτού λοιπόν δώσω το λόγο στους προσκεκλημένους ομιλητές μας, θα ήθελα να πω δύο λόγια για το πώς θα διαρθρωθεί η συζήτησή μας σήμερα. Και όσο εγώ θα μιλάω, μπορούν οι ομιλητές να έρθουν στο βήμα. Θα ακολουθηθεί λοιπόν η εξή διαδικασία. Ο λόγος θα δίνεται λάξ σε δύο μέλη Εθνικών Κοινοβουλίων και έναν Ευρωβουλευτή έως ότου εξαντληθεί ο κατάλογος των ομιλητών. Οι εθνικοί βουλευτές που θέλουν να παρέμβουν παρακαλούνται να συμπληρώσουν το έντυπο παρέμβασης και να το δώσουν στους κλητήρες, οι οποίοι με τη σειρά τους θα το φέρουν εδώ πάνω στο βήμα. Ο κατάλογος ομιλητών θα καταρτιστεί με βάση αυτές, με αυτά τα έντυπα, με τη σειρά που θα έχουν παραλυφθεί. Κάθε ευρωβουλευτής μπορεί να ζητήσει το λόγο κάνοντας απλώς ένα νεύμα προς τον Πρόεδρο, ως ήθιστε άλλωστε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Λοιπόν, αυτά και νομίζω ότι λίγο χάθηκα τώρα στις σημειώσεις μου. Όσον αφορά την πρώτη συζήτηση, θα ήθελα καταρχάς να προσκαλέσω την εισηγήτριά μας, την κυρία Πόστ, εισηγήτρια για την έκθεση 2017 για τα θεμελιώδη δικαιώματα όσον αφορά την ένταξη των Ρωμά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να μας κάνει μια γρήγορη παρουσίαση των πορισμάτων της έκθεσής της. Προτού της δώσω όμως το λόγο της Σοράγιας, θα ήθελα επίσης να ε, καλωσορίσω τον πρόεδρο της Επιτροπής μας, ο οποίος και, την πρόεδρο της Επιτροπής μας, η οποία και θα αναλάβει ε, τα καθήκοντά μου και θα με αντικαταστήσει. Thank you very much. And thank you, Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Μπίργκιτ, που προέδρευσες σε αυτή την εκδήλωση, την απογευματινή. Καλησπέρα, συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Χαίρομαι που σας βλέπω. Είναι σημαντική ημέρα. Ευχαριστώ όλους τους προσκεκλημένους ε, από τα Εθνικά Κοινοβούλια των Κρατών Μελών που αφιερώνουν το χρόνο τους για να συμμετάσχουν σε αυτή τη σημερινή συνεδρίαση της Διακοινοβουλευτικής Επιτροπής. Θα σας πω ποια είναι. Θα ακούσατε ότι το όνομά μου είναι Σοράγια Πόστ και είμαι μέλος της, ε, του, κόμματος, του Συνδικού Κόμματος ε, Φεμινιστικής Πρωτοβουλίας. Ήμουν εισηγήτρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την έκθεση θεμελιωδών δικαιωμάτων ε, και την ένταξη των Ρωμά, καθώς και την καταπολέμηση του αθηγανισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με αυτή την έκθεση ήθελα να σας δείξω ότι ο Ρώμα δεν απολαμβάνουν τα θεμελιώδη δικαιώματά τους λόγω αθηγανισμού. Ε, είναι μια συγκεκριμένη μορφή ρατσισμού εναντίον τους. Είναι αποτέλεσμα ε, δίωξης πολύχρονης γίνονται, είναι θύματα απόλυτης φτώχειας, απόλυτης ένδυας και είναι και από διοπομπέι τράγοι για πολλά δεινά. Θεωρούνται κατώτεροι, θεωρούνται τεμπέλιδες, δεν έχουν όρεξη να προσπαθήσουν, δεν είναι ικανοί και καλοί πολίτες στις χώρες που ζουν για χρόνια και δεν θέλουν να ενταχθούν. Ο αθηγανισμός βασίζεται σε αυτές τις πεπιθήσεις και οδηγεί σε συγκεκριμένες πράξεις, παίρνεται πολλές μορφές. Ε, ρητορίες μίσους, ε, στήρωση αναγκαστική των γυναικών, υπερβολική αστυνομική βία, απομόνωση στα σχολεία, στη στέγαση και τα λοιπά Υπάρχουν και άλλες πιο λεπτές μορφές ε, που οδηγούνται από μη ηθελημένη αμέλεια. Παραδείγματος χάρη, Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, υπάρχουν διάφορα προγράμματα για να βοηθήσουμε τα παιδιά των Ρωμά. Ε, τους του δίνουμε ας πούμε, δωρεάν ε, εισιτήρια για να συμμετάσχουν σε διάφορε εκδηλώσει. Ξεχνάνε όμω ότι δεν έχουν βασικά, ε, βασικές δυνατότητε για να καλύψουν άλλε ανάγκε του. δεν έχουν νερό. Ε, δεν έχουν τρεχούμενο νερό. Δεν έχουν ηλεκτρισμό στα σπίτια τους. Ε, τι να κάνουν όταν δεν ε, υπάρχουν ε, συγκοινωνίε στις περιοχέ που ζουν. Και υπάρχουν πάρα πολλοί καταβλισμοί Ρωμά που δεν έχουν αυτές τις βασικές υπηρεσίες, αυτές τις βασικές ευκολίες. το κενό ανάμεσα στους Ρωμά και στους μη Ρωμά είναι πολύ το, σημαντικό σε όλα τα πεδία ζωής. Ε, αν δείτε την τελευταία έκθεση της Δικαιοσύνης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ΦΡΑ, θα δείτε ότι 63% των νεαρών Ρωμά 16 ε, έως 24 χρονών είναι άνεργοι. Δεν πάνε σχολείο, δεν κάνουν κάποια κατάρτιση. Τη στιγμή που έγινε ας πούμε η πανευρωπαϊκή αυτή έκθεση, ενώ ο μέσος όρος για τους συνομιλικούς τους μη Ρωμά είναι 12%. 63 η Ρωμά, 12 η μη Ρωμά. Κάθε νοικοκυριό Ρωμά ζει ε, χωρίς τρεχούμενο νερό. Ένα στα δύο μάλλον. Ένα στα δύο δεν έχει κανονικό μπάνιο. Ένα στα πέντε σπίτια έχει στέγη που στάζει. Έχει σπασμένα ή σαπιά παράθυρα. Ένας από τους τρεις Ρωμά ε, έχει υποστεί παρενόχληση και πολλές γυναίκες έχουν υποστεί θύματα, έχουν πέσει θύματα φυσικής βίας. Συχνά ακούω να λένε ότι οι Ρωμά δεν θέλουν να ενταχθούν, δεν θέλουν να δουλέψουν. Φταίνε για την κατάστασή τους, λένε. Θα ήθελα να σας αναφέρω τον πρόεδρο Μιλοσέμα από την Τσεχική Δημοκρατία που πριν από λίγες εβδομάδες ότι οι Ρωμά είναι τεμπέλδες και ότι θα πρέπει να τους χαστουκίσουμε. Σας διαβεβαιώ τα εξής, για τα εξή όμως. Κανένα δεν θέλει να είναι φτωχό. δεν θέλει να είναι αποκλεισμένος. Και επίσης υπάρχει κάτι το καταστροφικό στο να ακούς μια ζωή να σου λένε ότι είσαι άχρηστος. Χειρότερος από τους άλλες, άλλους πολίτες, ότι είσαι πολίτης δεύτερης κατηγορίας. Και μην ξεχνάτε, μας το θυμίζουν αυτό καθημερινά. Πριν από λίγα χρόνια, εγώ μεγάλωνα για να ζήσω και να αναγνωρίσω τον εαυτό μου σαν ισότιμος πολίτης πρώτης κατηγορίας. Είμαι 62 χρονών. 50 χρόνια πέρασαν. Άντε, 55. Επί 55 χρόνια όμως έβλεπα τον εαυτό μου και έβλεπα στον καθρέφτη πολίτη δεύτερη κατηγορία. Γιατί έτσι με έβλεπε η κοινωνία. Συνεισέφερα στην κοινωνία. Επίση όρις. Όχι δεν μου επέτρεπαν. Γιατί δεν ήμουν πολύ τη πρώτη κατηγορία στην πραγματικότητα. Ήθελα να, συ, να συνεισφέρω σε αυτήν την κοινωνία. Σίγουρα. Όταν άρχισα λοιπόν να το κάνω, τότε άρχισα να εκτιμώ τη χώρα μου, τη δημοκρατία μου, να αισθάνομαι ότι αγαπώ τους συνανθρώπους μου. Εδώ στο Κοινοβούλιο αισθάνομαι ότι με σέβονται, αισθάνομαι ότι είμαι πολίτης πρώτης κατηγορίας αλλά έφτασα εδώ δύσκολα και δεν το πετυχαίνουν όλοι. Όχι ακόμα. Μη θεωρήσετε όμως σε καμία περίπτωση ότι δεν θέλουμε να δουλέψουμε, ότι δεν θέλουμε να συνεισφέρουμε. Σε καμία περίπτωση. Απλώς φοβόμαστε και δεν υπάρχει εμπιστοσύνη σε μας. Συχνά οι πιο ισχυροί και η πλειοψηφία θα πρέπει να κάνουν την χειρονομία και να φτάσουν στους πιο αδύναμους και, στους, και στη μειονότητα για να τη βοηθήσουν. Εγώ θέλω για τους Ρωμά ό,τι έχουν οι μη Ρωμά. Θέλω μια κοινωνία ίση για όλους. Όλοι να γεννιόμαστε ελεύθεροι και με την ίδια αξιοπρέπεια. Πρέπει να εξασφαλίσουμε την ισότητα ε, και την ισονομία. Δεν πρέπει να υπάρχει καμία διάκριση σε κανένα τομέα της ζωής. Και θα πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη. Να συνεργαστούμε γι' αυτό, γιατί χωρίς εμπιστοσύνη δεν υπάρχει μέλλον. Είμαι πεπισμένη ότι ο αθηγανισμός είναι η βασική αιτία αυτής της δυσπιστίας που υπάρχει στις κοινωνίες μας σήμερα, που θα καθυποτάξουμε μόνο εάν δημιουργήσουμε επιτροπές ε, συμφιλίωσης στις χώρες μας. Θα πρέπει να καταλάβουμε τι περνάνε οι Ρωμά τα, τις τελευταίες δεκαετίες και αιώνες τις φρικαλαιότητες που αντιμετωπίζουν ακόμα και σήμερα. Το να ζεις αποκλεισμένο σου καταρακώνει την εικόνα που είσαι τον εαυτό σου. Το πώς βλέπεις το γειτονά σου. Και το πώς εκτιμάς τον εαυτό σου και τις ικανότητές σου. Ήμασταν σκλάβοι, διωχθήκαμε, και μας διώξανε σχεδόν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες. Συστηματικά μας δολοφονούσαν κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι γυναίκες μας επί δεκαετία στηρώνονταν υποχρεωτικά. Τα παιδιά μας, μας τα παίρνανε και τα βάζανε σε ιδρύματα κρατικά. Και αυτό δεν είναι ιστορία. Αυτό συμβαίνει ακόμα και σήμερα και γίνεται όλο και χειρότερο. Τα παιδιά μας θεωρούνται κατώτερα πνευματικά και ότι θα πρέπει να πηγαίνουν σε χωριστά σχολεία επί αιώνες μας αρνούντα την ανθρωπιά μας. Πρέπει να υπάρξει μια ευαισθητοποίηση, ένας διάλογος και να σταματήσουν αυτές οι αντιλήψεις να κυκλοφορούν στα βιβλία και στα σχολεία κτλ. Γι' αυτό σας κάνω έκκληση να δημιουργήσετε γέφυρες, να δημιουργήσετε επιτροπές συμφιλίωσης στις χώρες σας. Και κάτι άλλο σημαντικό. Μετά από μεγάλη καθυστέρηση, οι πολιτικοί θα πρέπει να αναλάβουν τι ευθύνες τους και να αναλάβουν και τις ευθύνες για τους πολίτες Ρωμά που έχουν στις χώρες τους. Όταν πηγαίνω σε διάφορε αποστολέ, να δω ποια είναι η κατάσταση επιτόπου, πάω σε διάφορου Δήμου και κοινότητε. και βλέπω ότι οι αρχές Βλέπουμε τελείως διαφορετικό μάτι τους πολίτες Ρωμά από τους υπόλοιπου πολίτες. Δεν είναι σημαντικό για αυτού το γεγονό ότι τα παιδιά των Ρωμά δεν, έχουν, δεν πάνε στο σχολείο, ότι δεν έχουν τρεχούμενο νερό. Είναι συνηθισμένοι, λένε. Είναι στην κουλτούρα του. Φταίει η κοινότητα των Ρωμά, ε, λένε, για αυτή την ε, κατάσταση. Αλλά είναι ντροπή για την Ευρώπη ότι διαιωνίζεται αυτή η κατάσταση θα πρέπει οι πολιτικοί να αναλάβουν τι ευθύνε του για όλου όσου είμαστε εδώ σε αυτήν την αίθουσα. Για όλου του πολίτε. Και όχι μόνο κατά τη διάρκεια των εκλογών ε, βουλευτικών ή το, της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δεν θα πρέπει να γινόμαστε από δύο πομπέι τράγοι. Είναι ντροπή αυτό. Γιατί αλλιώς οι ρητορίες μίσους, ε, η θυματοποίησή μας θα ρηπάνουν ακόμα περισσότερο τις κοινωνίες μας. Θα πρέπει αντίθετα οι κοινωνίες μας βασίζονται στην ανεκτικότητα, σε ανοιχτό πνεύμα, σε αξίες, στις αξίες που διασφαλίζονται και μέσα από τις ευρωπαϊκές συνθήκες, τις συνθήκες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ όλους όσους είστε σήμερα εδώ και όταν επιστρέψετε στη χώρα σας, ελπίζω να αναλάβετε τις ευθύνες για όλους τους πολίτες, ανεξάρτητα από την ε, εθνική τους προέλευση, το φίλο τους, από τις διαφορές τους. Έχει σημασία. Και οι πολίτες Ρωμά μετράνε. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους που υποστήριξαν την έκθεση από την αρχή και ευχαριστώ όλους όσους δέχονται την ευθύνη για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες, όποιοι και να είναι αυτοί. Thank you, Soraya. Ευχαριστούμε, Σοράγια. Καταπληκτική η παρέμβασή σου. Να δώσουμε τώρα το λόγο στον κύριο Ιωάννη Δημητρακόπουλο, επικεφαλής ε, του Τμήματος ε, Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στον ε, Οργανισμό Θεμελιώδων Δικαιωμάτων, που θα μας παρουσιάσει τα βασικά ευρήματα του FRA για το αντιαθυγανισμό ως εμπόδιο στην κοινωνική συμπερίληψη των Ρωμά. Παρακαλώ, έχετε το λόγο για 10 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ που προσκαλέσατε τον οργανισμό μας ε, σε αυτή τη σε πάντα είναι πολύ σημαντικό να μοιραζόμαστε τις προτάσεις μας ε, με τα μέλη του Ευρωπαϊκού αλλά και των Εθνικών Κοινοβουλίων. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία καθώς, ε, όπως ανέφερε και η Γενική Διευθύντρια στο ΛΕΑ προηγουμένως, να δούμε τι έχει συμβεί και τι έχει επιτευχθεί από το 2011 υπάρχει το ενωσιακό πλαίσιο το οποίο έθεσε τη συμπερίληψη των Ρωμά πρώτη, για πρώτη φορά ε, σε ένα πλαίσιο θεμελιωδών δικαιωμάτων με άμεσε ε, παραπομπές στι ευρωπαϊκές Συνθήκε και στην χάρτα θεμελιωδών δικαιωμάτων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Άκουσα και από άλλου ομιλητέ για την ε, σύσταση του Συμβουλίου του Δεκεμβρίου του 2013 για αποτελεσματικά μέτρα ενσωμάτωσης και ένταξης των Ρωμά στα κράτη-μέλη. Αναφέρεται και συγκεκριμένα ότι πολλοί Ρωμά στην Ένωση έρχονται αντιμέτωποι με ε, ανέχεια, κοινωνικό αποκλεισμό, διακρίσει και ε, προσκόμματα προ την άσκηση των θεμελιωδών του δικαιωμάτων, το οποίο του εκθέτει στην εκμετάλλευση. Δεν είναι εξορισμού όμως ευάλωτη ομάδα η Ρωμά. Καθίστανται ευάλωτοι όταν έρχονται αντιμέτωποι με την ανέχεια, την, ε, τον κοινωνικό αποκλεισμό, ε, και την προκατάληψη και τον αντιθεγανισμό. Τα μέτρα πολιτικής ε, που συστήνονται από το Συμβούλιο περιλαμβάνουν μέτρα κατά των διακρίσεων και των προκαταλήψεων κατά τον Ρωμά και από τότε ο οργανισμός μας ε, εκπονεί ένα έργο συγκέντρωσης στοιχείων και δεδομένων και από τα γραφεία μας στη Βιέννη, αλλά και επιτόπου, στις τοπικές ε, κοινωνίες, πηγαίνουμε και βλέπουμε πώς ε, υλοποιούνται ή δεν υλοποιούνται τα μέτρα ε, για την κοινωνική ένταξη των Ρωμά. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, προσπαθούμε και σε τοπικό επίπεδο να δούμε πώς λειτουργούν οι αρχές τι πάει καλά και τι δεν πάει καλά, αλλά και από το επίπεδο της αρχής μας. Πέντε χρόνια αργότερα, λοιπόν, τα δεδομένα τα οποία συλλέγουμε συστηματικά δείχνουν ότι η Ένωσή μας, που να μην το ξεχνάμε και αυτό είναι από τις ε, πλουσιότερες περιοχές στον κόσμο ακόμα δεν μεταχειρίζεται με τον ίδιο τρόπο και ισότιμα τους πολίτες Ρωμά. Υποβαθμίζουν και υποσκάπτουν την κοινωνική, τους, ε, την κοινωνική συνοχή, την ανταγωνιστικότητα και γενικά ε, και τελικά δημιουργούν και κόστος για την ευρωπαϊκή κοινωνία στο σύνολό τη. Ε, έχουμε αποτρόπες μορφές αντι αδιαθυγανισμού, από ε, εγκλήματα με κίνητρο το μίσος, ε, παρενόχληση και βλέπουμε ότι κάθε φορά που οι κυβερνήσεις ε, λαμβάνουν μέτρα αποτυχάνουν εάν δεν υιοθετούνται και παράλληλα και άλλα μέτρα, γιατί από μόνο τους δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Δεν θέλω να επαναλάβω όλα τα στοιχεία που ανέφερε Σωράγια. Αυτό που θέλουμε πραγματικά παράδειγμα είναι το 4% ε, των ερωτηθέντων με δειγματοληπτικές διαδικασίες ε, στους Ρωμά σε νέα κρατημέλη βλέπουμε ε, ότι έχουν έρθει αντιμέτωποι με βία, με κίνητρο το μίσος. Αυτό μεταφράζεται σε εκατοντάδες περιπτώσεις που θα έπρεπε να έχουν φτάσει στην αστυνομία και στη δικαιοσύνη. Αλλά δεν συνέβη αυτό γιατί τα θύματα αυτή τη βία ε, δεν πηγαίνουν στην αστυνομία. Μόνο το 1 τρίτο έχει πάει στην αστυνομία. Πρέπει λοιπόν να ενισχύσουμε την υποστησύνη στι αρχέ επιβολή του νόμου, που θα βοηθήσει του Ρωμά ε, να αναφέρουν τέτοια περιστατικά. Οι προκαταλήψει όμω επηρεάζουν και τι ευκαιρίε που έχουν στη ζωή Ακούσαμε τα στοιχεία πριν ε, για, τις, ε, για την ανεργία στους νέους, όμως οι νέοι Ρωμά έχουν πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα σχέση με τον γενικό πληθυσμό και οι γυναίκες, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν σημαντικά ε, κονδύλια ευρωπαϊκά, αλλά δεν αξιοποιούνται πάντα στο βαθμό που πρέπει. Βλέπουμε ότι η στέγαση επίση είναι πολύ σημαντικό παράγοντα σε ό,τι αφορά τι ευκαιρίε που έχει κανεί στη ζωή. Το να ζει κανεί σε καθεστώς κοινωνικού διαχωρισμού και προκαταλήψεων με, σε ακατάλληλες συνθήκες συνδέεται με δύο μεταβλητές. Να, το να μην είναι κάποιος στο εκπαιδευτικό σύστημα και να μην ε, εργάζεται κανείς. Βλέπουμε ότι πολύ σημαντικό τμήμα των Ρωμά εξακολουθούν να ζουν υπό ε, πολύ άσχημες συνθήκες. Στη Ρουμανία, για παράδειγμα, 68% των Ρωμά δεν έχουν τρεχούμενο νερό στο σπίτι τους για δεκαετίες για εμάς εδώ ας πούμε στην αίθουσα είναι κάτι το δεδομένο. Ένα εξαιρετικά χαμηλό ποσοστό του γενικού πληθυσμού με βάση τα στοιχεία της Eurostat ε, ζει υπό τέτοιες συνθήκες. Του χρόνου το καλοκαίρι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις θα συζητήσουν με τους ομολόγους τους ε, του ΟΗΕ στην ε, Νέα Υόρκη σε ό,τι αφορά την πρόοδο που έχει σημειωθεί για την επίτευξη των του, στόχου υπαριθμών 10 ε, βιώσιμης ανάπτυξης υπό το θεματολόγιο για το 2030. Και πραγματικά θα είναι μεγάλη ντροπή να αναγνωρίσουμε ότι παγκοσμίω η αναλογία, το ποσοστό των ε, νέων Ρωμά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι και από τι πλουσιότερε περιοχέ στον κόσμο, των άνεργων λοιπόν νέων, ε, ή μάλλον αυτών που δεν βρίσκονται στην ε, απασχόληση, στην αγορά εργασία ή στην κατάρτιση, αντιστοιχεί στα επίπεδα που βλέπουμε στην Ονδούρα, στην Ιεμένη, στο Τρινιδά, τον Πάγκο και στη Σαμόα. Ε, εξίσου χαμηλά είναι τα ποσοστά όσων έχουν πρόσβαση ε, σε καθαρό νερό. Αντίστοιχα χωρών όπως το Μπουτάνι, Γκάνα και το Νεπάλ. Όλα αυτά δεν είναι τυχαία. Αποτελούν το αντικείμενο ε, διακρίσεων που χρονίζουν. Το 2019 συμπληρώνονται 50 χρόνια από τότε που η Κοινοβουλευτική Σύνοδος του Συμβουλίου της Ευρώπης εξέφρασε τη βαθιά του ανησυχία στη σύσταση 563 ε, για την αδυναμία του να βελτιώσουν την κατάσταση των Ρωμά στην Ευρώπη. 50 χρόνια πριν, έτσι. Και αναφέρεται ότι μάλιστα η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα, μπορούμε να πούμε ότι είναι εξαιρετικά λυπηρή κατάσταση, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρείται φάρος ε, ε, προαγωγής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θα περίμενα κανείς ότι θα μπορούσαμε να σημειώσουμε σημαντική βελτίωση στις ζωές των Ρωμά. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν, αυτό που λέω πάντα, πρέπει ε, να επιμείνουμε, πρέπει να επενθυμίζουμε στις κυβερνήσεις μας ότι είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος που πρέπει να αναλάβουν και ότι υπάρχει και σημαντική ευθύνη να υπενθυμίζουμε συνεχώς τις κυβερνήσεις σε τον αντίκτυπο του αντιαθηγανισμού που υποσκάπτει την ε, προσήλωσή του στη συμπερίληψη των Ρωμά. Να υπερθυμίζουμε τη σύσταση του Συμβουλίου. Πρώτα απ' όλα να διασφαλίσουμε ότι υπάρχει σωστό συντονισμό σε εθνικό επίπεδο και εδώ συγχαίρω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που από το 2012 και όλας ανέπτυξε ένα δίκτυο εθνικών σημείων επαφής Ρωμά που συναντούνται συχνά και ανταλλάσσουν πληροφορίες και δεδομένα. Ξέρω ότι η δική μου χώρα τώρα καταβάλει προσπάθειες ε, να αναπτύξει ένα τέτοιο δίκτυο σε περιφερειακό επίπεδο, ούτως ώστε ε, το, οι προσπάθειε αυτές σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, εκεί που πράγματι μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, να γίνονται με πιο αποτελεσματικό τρόπο. Πρέπει να πείσουμε τις κυβερνήσει μας ότι πρέπει ε, να υιοθετήσουν και να υλοποιήσουν πολιτικές μείωση τη ε, ανέχεια που θα αξιοποιούν ε, μέτρα κοινωνική προστασία και και εργατικών μεταρρυθμίσεων αξιοποιώντα το έπακρο, τα ευρωπαϊκά διαφορετικά και επενδυτικά ταμεία, ε, καθώς και το ταμείο για τους ε, πλέον μειονεκτούντες. Μετά, πρέπει να βελτιώσουμε τις συνθήκες ε, στέγασης των Ρωμά, να καταπολεμήσουμε τον διαχωρισμό τους από την υπόλοιπη κοινωνία και να διασφαλίσουμε ότι θα έχουν πλήρη πρόσβαση στις υπηρεσίες κοινή ωφελία και υποδομές. Κυρίε και κύριοι, έχουμε μια πολύ σημαντική ευκαιρία εφόσον ολοκληρώνεται ο κύκλο ε, του θεματολογίου 2011, κλείνει τον κύκλο του 2020 και τώρα θα περάσει στη φάση τη αναθεώρηση. Η ανάλυση μα δείχνει ότι η διαδικασία τη συμπερίληψη των Ρωμά ε, πρέπει να αλλάξει, δεν μπορεί να συνεχιστεί στην πεπατημένη. Ε, πρέπει να συζητήσουμε τι ανεπάρκειέ μα και να ανανεώσουμε την προσήλυσή μα για να πετύχουμε του βασικού στόχου μα που είναι να κάνουμε τη διαφορά στι ζωέ των Ρωμά. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστούμε πολύ. Επόμενος ομιλητής, ο κύριος Jonathan ε, Μακ από το Κεντρικό Συμβούλιο Ρωμά και Σύντη στη Γερμανία, ο οποίος ε, αντικαθιστά τον ε, κύριο Ρωμάνη τον πρόεδρο του Συμβουλίου. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Δυστυχώς ο κύριος Ροζ είχε ένα ατύχημα. Ζητά συγγνώμη, γι' αυτό και θα μιλήσω εκ μέρους του. Αγαπητοί Πρόεδρε, αγαπητά μέλη των Εθνικών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θέλω να ευχαριστήσω την ε, Επιτροπή ΛΥΜΠΕ για την ευκαιρία που μας δίνεται να συζητήσουμε σήμερα εδώ την κοινωνική ένταξη και τα θεμελιώδη δικαιώματα των Ρωμά. Το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την αντιμετώπιση του αντιαθηγανισμού είναι θεμελιώδου σημασία για του Ρώμα και του Σύντη σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και θέλω να ευχαριστήσω τη Σοράγια Πόστ για την εξαιρετική της δουλειά ε, και για όλο το έργο που έχει επιτελέσει γύρω από αυτό το θέμα. Για πρώτη φορά το θέμα του αντιαθηγανισμού αντιμετωπίζεται πλέον ως πηγή ε, βίας, αποκλεισμού που επηρεάζει και πλήττει μεγάλα τμήματα της μειονότητας αυτής. Ο αντισημιτισμός και ο αντιαθηγανισμός έχουν βαθιές ρίζες στην ευρωπαϊκή ιστορία. Εμφανίζονται ως προκαταλήψεις στον πληθυσμό, ως ε, στέρηση της ανθρώπινης ιδιότητας από τους ε, ε, Ρωμά, ως δομικές και διαρθρωτικές διακρίσεις εις βάρος των Ρωμά σε πάρα πολλούς θεσμούς. Αυτή η μορφή του, των διακρίσεων εμποδίζει την ίση συμμετοχή των Ρωμά σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής. Αν μιλήσουμε για την απελπιστική κατάσταση στη στέγαση ή την απελπιστική κατάσταση στην παιδεία, τον διαχωρισμό και τις διακρίσεις που υφίστανται σε αυτούς τους τομείς οι Ρωμά, πραγματικά πρέπει να κατανοήσουμε ότι, αυτά αυτή, ε, ότι αυτές οι διακρίσεις, αυτά τα προβλήματα είναι αντικειμενοποιημένος ρατσισμός. Για πάρα πολλά χρόνια οι Ρωμά ε, αντιμετωπίζονταν ως κοινωνικό πρόβλημα που προσπάθησαν να επιλύσουν οι κυβερνήσεις με στρατηγικές κατεπολέμησης της φτώχειας. Όμως αυτές οι στρατηγικές αγνοούν πολλές φορές τον υποβόσκοντα αντιαθηγανισμό που συμβάλλει στην συνέχιση αυτού του φαύλου κύκλου του αποκλεισμού και της περιθωριοποίησης. Στην ουσία είχαμε την, ε, ε, τα θύματα να είναι εκείνα που κατηγοριούνται για την ε, απελπιστική τους κατάσταση. Τα τελευταία στοιχεία λοιπόν δείχνουν ότι χρειάζεται για την κοινωνική ένταξη να υπάρξουν ε, πολύπλευρα και πολύμορφα μέτρα ο, η καταπολέμηση του αντιαθηκανισμού δεν είναι πρώτα και κύρια ευθύνη της ίδιας της μειονότητας, αλλά ολόκληρης κοινωνίας και των θεσμικών της οργάνων. Είναι ε, καθήκον των ευρωπαϊκών κρατών και των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, γιατί οι Ρωμά είναι ισότιμοι πολίτες των κρατών μελών. Βλέπουμε σημαντική πρόοδο στην πολιτική συζήτηση όσον αφορά τον αντιαθηκανισμό. Ταυτόχρονα η απόρριψη Ρωμά και Σύντη μεταξύ του γενικού πληθυσμού είναι ακραία υψηλή, όπως δείχνουν και τα στοιχεία που μας παρουσίασε ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Αυτή η τάση, σε συνδυασμό με τον ε, ε, ε, ολοένα και αυξανόμενο εθνικισμό τα τελευταία χρόνια, αποτελεί μεγάλη απειλή για τις κοινότητες των Ρωμά σε, σχεδόν σε όλες τις χώρες. Στη Γερμανία και σε ολόκληρη την Ευρώπη, οι Σύντη και η Ρώμα αντιμετωπίζουν προκαταλήψεις, επιθέσεις και βία πριν από μία εβδομάδα δολοφονήθηκε ένας 17χρονος ε, Ρωμά καθώς ε, μάζευε άχυρο σε χωράφι. Αντίστοιχη επίθεση έγινε στο Βερολίνο πριν από λίγο καιρό. Η βία είναι ε, παρούσα διαρκώς στις κοινότητες των Ρωμά. Πρέπει λοιπόν οι αρχές να μπορέσουν να εντοπίζουν με μεγαλύτερη σαφήνεια της, ε, τον αντιαθηγανισμό ως πηγή, ως κίνητρο των, ε, ε, των εγκλημάτων εις βάρος των Ρωμά. Σημειώνουμε εδώ τον, την πρόταση του, του Πρωθυπουργού της Ιταλίας Σαλβίνη να δημιουργηθεί ειδικό μητρό στο οποίο θα πρέπει να καταχωρίζονται όλοι οι Ρωμά. Αυτό είναι πλήγμα στο κράτος δικαίου στην Ιταλία. Δυστυχώς ε, αυτή είναι η κατεύθυνση που έχει χαράξει το Υπουργείο Εσωτερικών της Ιταλίας. Πριν από λίγες εβδομάδες, ο δήμαρχος του Ντουίσμπουργκ ε, ξεκίνησε μια ρατσιστική συζήτηση για την, για την κατάχρηση των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Είπε ότι τράφικερ φέρνουν Ρωμά από τη Ρουμανία στη Γερμανία ε, και στη συνέχεια είπε ότι πρέπει να αντιμετωπίσω ανθρώπους που βρωμίζουν δρόμους και που ενισχύουν το πρόβλημα που έχουμε με τους αρουραίους. Όποιος ξέρει ιστορική Γερμανία, ε, ιστορία της Γερμανίας, ξέρει πολύ καλά ποιο είναι ο παραλληλισμό μεταξύ Εβραίων και Αρουραίων και πώς έχει χρησιμοποιηθεί από την ακροδεξιά στη Γερμανία. Αυτά συμβάλλουν στην ενίσχυση του μίσου, στην κοινωνία μας και καθιστούν θύματα τους Ρωμά επιθέσεων και μίσους. Δεν μπορούμε να μιλάμε για τον αντιαθηγανισμό όταν ταυτόχρονα δεν βάζουμε στο επίκεντρο της προσοχής μας την πιο ακραία και ριζοσπαστική μορφή τους. Την, ε, την ε, εξόντωση μισού εκατομμυρίου Ρωμά, Ρωμά στο πλαίσιο του ολοκαυτώματος. Και αυτό στη βάση μιας απάνθρωπης ιδεολογίας. Εξοντώθηκαν γιατί γεννήθηκαν Σύντι και Ρωμά. Οι νόμοι του 1935 αφορούσαν τόσο τους Εβραίους όσο και τους Ρωμά και ξεκίνησαν μια διαδικασία στέρησης δικαιωμάτων και διώξεων που τελικά κατέληξαν στην εξόντωση όλων των, που είχαν ως σκοπό την τελική εξόντωση όλων των Εβραίων και των Ρωμά σε όλη την Ευρώπη. Χρειάστηκαν δεκαετίες μέχρι να αναγνωριστούν τα εγκλήματα κατά των Ρωμά το 1982 έπειτα από ακούραστες προσπάθειες των ε, απογόνων των Ρωμά θυμάτων των Ναζί. Το 2015 αποτέλεσε και το ψήφισμα που ενέκρινε το Γερμανικό Κοινοβούλιο αποτέλεσε ιστορικό ορόσημο, γιατί έκτοτε αναγνωρίζεται ρητό πλέον η γενοκτονία κατά τον Ρωμά στη Γερμανία. Υπήρχαν και άλλες σημαντικές ε, θετικέ εξελίξεις. Στη βάση ενός ε, σχεδίου ψηφίσματος του Bundestag η γερμανική κυβέρνηση ε, σύντομα θα συγκαλέσει ανεξάρτητη συνδιάσκεψη για την καταπολέμηση του αντιαθηγανισμού έτοιμά μα εδώ και πάρα πολλά χρόνια που θα έχει ε, ως σκοπό να καταγράψει τον αντιαθηγανισμό και, τις, ε, και, τις, ε, τους τρόπους εκδήλωσής τους στην ε, ολόκληρη Γερμανία. Ταυτόχρονα θα υποβληθεί στο Κοινοβούλιο έκθεση από, τον, ε, από την συνδιάσκεψη αυτή και στην βάση αυτής της έκθεσης θα χαρακτεί μια νέα στρατηγική. 800.000 ευρώ έχουν ήδη ε, προσημειωθεί για την σύνταξη αυτή τη έκθεση και χαιρετίζουμε το γεγονός ότι η γερμανική ομοσπονδιακή κυβέρνηση έχει επενδύσει αρκετά εκατομμύρια τα τελευταία χρόνια στην εκπαίδευση για την καταπολέμηση του αντιαθηκανισμού. Επίσης, δημιουργήθηκε πρόσφατα ερευνητικό κέντρο στο Πανεπιστήμιο τη Χαϊδελβέργη με αντικείμενο την διερεύνηση του αντιαθηκανισμού. Το ευρωπαϊκό ψήφισμα του 2017 προτείνει να δημιουργηθούν σε εθνικό επίπεδο ομάδες εμπειρογνωμόνων ε, με τον τίτλο «Ομάδες αλήθειας και ε, συμφιλίωσης». Σας καλώ να μεταφέρετε αυτό το αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα εθνικά σας κοινοβούλια. Επιτέλους, λοιπόν, ο αντιαθηγανισμός αποτελεί κεντρικό σύστημα... στην κεντρική πολιτική ε, σκηνή. Σε αυτό το πλαίσιο έγινε και η συνδιάσκεψή μας στο Βερολίνο το 2016 σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με τον ΟΣΑ και με το Συμβούλιο της Ευρώπης. Η συνδιάσκεψη εκείνη απάντησε στο σημαντικό ερώτημα που πρέπει να διαδραματίσουν οι πολιτικοί ηγέτες στην καταπολέμηση του αντιαθηγανισμού. Στόχος ήταν να δημιουργηθεί μια διεθνής ε, κοινοβουλευτική συμμαχία κατά του, αντι... αντιαθηγανισμού. Θα ήταν πολύ σημαντικό αν σήμερα μπορούσαμε να αναβαθμίσουμε αυτή τη συμμαχία μας προκειμένου να υπάρξει συνεργασία μεταξύ Εθνικών Κοινοβουλίων της Διακοινοβουλευτικής Διάσκεψης ε, του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κυρίες και κύριοι, η μετεξέλιξη και η πορεία προς μια πιο δημοκρατική Ευρώπη δεν ήταν μια πορεία ε, αυτονόητη, αλλά χρειάστηκε πολλές προσπάθειες. Ο αντιαθηγανισμός είναι ευθεία επίθεση κατά των ευρωπαϊκών αξιών και των δικαιωμάτων. Γι' αυτόν τον λόγο ο αντιαθηγανισμός θα πρέπει να απαγορευτεί και να επιβάλλονται κυρώσεις σε όλες αυτές τις περιπτώσεις. Αυτό χρειάζεται την προσήλωσή μας, όλων μας, και την δέσμευση από τα κράτη-μέλη και από τα, θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι ο θα αποτελέσει, η καταπολέμηση του αντιαθηγανισμού θα αποτελέσει βασικό και θεμελιώδες στοιχείο όλων των εθνικών στρατηγικών που θα καταρτιστούν από το 2020 και έπειτα. Ευχαριστούμε κύριε Μακ. Τώρα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε τις απόψεις των μελών των Εθνικών Κοινοβουλίων, των Εθνικών Βουλευτών. Ο Τόμας Χάμαρμπεργκ, που είναι Σουηδός ε, βουλευτής. Θα μας ε, μιλήσει. Έχει 10 λεπτά. Εν συνεχεία θα δώσω το λόγο στους υπόλοιπους. Στους υπόλοιπους εθνικούς βουλευτές που θέλουν να πάρουν το λόγο. Ακόμα υπάρχει δυνατότητα, εφόσον το επιθυμείτε, να μιλήσετε στο πρώτο πάνελ ή στο δεύτερο πάνελ, να συμπληρώσετε αυτό το έντυπο. Ευχαριστώ. Δεν ε, ισχύζομαι ότι εκπροσωπώ όλα τα κοινοβούλια της Ευρώπης. αλλά αυτή η διάσκεψη πιστεύω ότι είναι σημαντική. Είναι σημαντικό να έχει το προβάδισμα η Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση του αθηγανισμού. Γιατί σε μεγάλο βαθμό είναι ευρωπαϊκό αυτό το πρόβλημα. Η πραγματική δράση όμως γίνεται σε τοπικό επίπεδο επί κάποια χρόνια, πριν κάποια χρόνια μάλλον, ήμουν επίτροπο ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Συμβούλιο τη Ευρώπη και δου... ταξίδεψα σε όλε τι ευρωπαϊκέ χώρε, μερικέ φορέ ε, κατ' επανάληψη. Και μία από τι ε, βασικέ μου εντυπώσει ήταν ότι αυτό το θέμα δεν έχει λυθεί στις ευρωπαϊκές χώρες και κοινωνίες. Ε, για να μην πω ότι στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες ε, είχαμε σοβαρές αποτυχίες για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος του αθηγανισμού. Νομίζω ότι είναι και καινή ώρα να αντιμετωπίσουμε πλέον αυτό το πρόβλημα. Ακούσαμε τις στατιστικές, ακούσαμε διάφορες υποθέσεις που παρουσιάστηκαν. Δυστυχώς, αυτή είναι η πραγματική κατάσταση. Θα προσπαθήσω να αναφερθώ σε κάποιες δράσεις που ελπίζω ότι θα αναλυφθούν από τα εθνικά κοινοβούλια σε αυτή την προσπάθεια να καθαρίσουμε την Ευρώπη από αυτό το επονίδιστο πρόβλημα διάκρισης, όπου ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού στην Ήπειρό μας ε, έχει πρόβλημα. Μιλάμε για 800 εκατομμύρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγγνώμη, 12 εκατομμύρια συνολικά στην Ευρώπη λοιπόν και είναι πρόβλημα. Πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Θα πρέπει κάπου να μπει στην πολιτική συζήτηση και μάλιστα να ανέβει ως προτεραιότητα. Επίσης δεν μπορούμε να κάνουμε νυφάλια συζήτηση χωρίς να ξεκαθαρίσουμε τα ιστορικά στοιχεία. Νομίζω λοιπόν ότι ε, εξεταστικές επιτροπές πρέπει να συσταθούν. Καταφέραμε να πείσουμε τις Σουηδικές Αρχές να κάνουν κάτι τέτοιο και σας καταμαρτυρώ ότι η επίπτωση στις σχέσεις μεταξύ της πλειονότητας του πληθυσμού και των Ρωμά στη Σουηδία βελτιώθηκε. Ε, υπάρχουν ακόμα προβλήματα σε ό,τι αφορά την εμπιστοσύνη που έχουν οι μέσα τους ΔΕ. Αλλά ξεκίνησε ένας διάλογος μεταξύ των Ρωμά και των ΜΗ που είναι σημαντικό. Το επόμενο βήμα στη Σουηδία ήταν να δημιουργηθεί μια επιτροπή η οποία δεν θα ασχοληθεί με ιστορικά θέματα και παρελθόντα εγκλήματα, και παραβιάσει τον εναντίον των Ρωμά, αλλά θα κοιτάξει και τη σημερινή κατάσταση. Δημιουργήθηκε με νέα μέλη η Επιτροπή αυτή, έξι ήταν Ρωμά, έξι μέλη τη επιτροπή ε, ήταν Ρωμά και οι υπόλοιποι ήταν εμπειρογνώμονε από άλλα στρώματα τη κοινωνία. Αυτοί οι εννέα άνθρωποι ετοίμασαν μια έκθεση για το τι θα πρέπει να γίνει τώρα, τι δράσει θα πρέπει να προαχθούν ούτω ώστε να εξασφαλίσουμε ότι ο αθηγανισμό θα εξαλειφθεί. ότι ο ανδιαθηνικανισμός θα εξαλειφθεί. Συγγνώμη. Πρέπει να δούμε τι πρέπει να κάνουμε. Ε, είναι, ήταν θετική εμπειρία μας και νομίζω ότι θα μπορούσαν να εμπνευστούν και άλλες χώρες από εμά, από αυτό το μοντέλο. Είναι σημαντικό να δούμε τι μπορεί να γίνει συγκεκριμένα, με συγκεκριμένες υποθέσεις. Είχαμε μια σοβαρότατη υπόθεση όπου αποκάλυψαν τα μέσα ενημέρωσης ότι η αστυνομία κάπου στη Σουηδία είχε ένα μητρό και το οποίο το επικαιροποιούσε κάθε τόσο με τους Ρωμ και κατέγραφε ποιος Ρωμά ζούσε στην περιοχή εκεί, ποιες οικογένειες ε, και κάλυπτε ε, και είχε εκεί πέρα καταχωρημένους πάρα πολλούς Ρωμά. Μη, σου πω το, μεγαλύτερο αριθμό του, του πληθυσμού Ρωμά της Σουηδίας. Ε, προκάλεσε κατακραυγή στους Ρωμά. Ε, το γεγονός δηλαδή ότι η αστυνομία τους κατέγραφε σε ένα μητρό μόνο και μόνο γιατί ήταν Ρωμά, αλλά το κάνανε. Το στο αστυνομικοί αυτό. Χρειάστηκε μια πολιτική δράση για να εξασφαλίσουμε ότι θα σταματούσε αυτό και ότι άλλου τύπου καταχωρήσεις δεν θα συνεχιζόταν και στο μέλλον. Είναι σημαντικό να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα. Θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα επίσης και στη δράση που κάνουν οι διαμεσολαβητές. Έχουμε παντού σε όλη την Ευρώπη ε, διαμεσολαβητές. Τα θέματα των διακρίσεων κατά τον Ρωμά θα πρέπει να τα λαμβάνουν υπόψη πολύ σοβαρά. Σε ορισμένε χώρε ασχολούνται πραγματικά σοβαρά με το πρόβλημα των διακρίσεων κατά τον Ρωμά. Σε άλλε χώρε όμω όχι. Είναι πολύ σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε ότι σε ό,τι αφορά τι διακρίσει και τις δράσεις κατά του πληθυσμού των Ρωμά ότι θα σταματήσουν αυτές οι δράσεις. Να είναι σίγουροι οι Ρωμά ότι τα παράπονά τους ε, θα αντιμετωπίζονται σαν σοβαρά για να μπορούν να υποβάλουν ε, παράπονα. Επίσης, ε, υπήρχαν προκαταλήψεις τους δικαστές στη δικαιοσύνη κατά τον Ρωμά. Και όταν τα θέματα πηγαίναν στην αστυνομία, ας και έλεγαν «Μου συνέβη το και το», έβλεπαν ότι ποτέ η αστυνομία δεν ερευνούσε τα καταγγελόμενα. Και ελάχιστες περιπτώσεις φτάθηκαν στο δικαστήριο Για... Και σε ελάχιστες περιπτώσει οι υπεύθυνοι τιμωρήθηκαν. Συχνά λοιπόν η Ρωμά συμπέρναν ότι δεν έχει νόημα κα, κανείς να φύγει στην αστυνομία και να καταγγείλει διάφορα κακοσκήμενα. Άρα αυτό δεν ήταν υπέρ της εμπιστοσύνης, αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Το γεγονός ότι ασχοληθήκαμε αυτά τα θέματα άλλαξε την κουλτούρα. Επίσης κάποιοι επαγγελματίες οι οποίοι είναι σε μεγαλύτερη επαφή με τον πληθυσμό των Ρωμά θα πρέπει να έχουν κάποιες πληροφορίες, να είναι κάπως εκπαιδευμένοι για την κουλτούρα των Ρωμά, για τους ανθρώπους αυτούς. Ειδικά σε ό,τι αφορά τους αστυνομικούς, τους δασκάλους, διάφορους ε, κοινωνικούς λειτουργούς και άλλους λειτουργούς στα πλαίσια της κοινότητας, είναι σημαντικό ότι αυτοί που εκπροσωπούν ε, την κοινωνία και έρχονται σε επαφή με Ρωμά, ε, να γνωρίζουν κάπως την κουλτούρα των Ρωμά, να ξέρουν τι εργαλεία πρέπει να έχουν για να κάνουν τη δουλειά τους, ούτω ώστε να μην βαθύνουν αυτό το χάσμα που υπάρχει αυτή, την έλλειψη εμπιστοσύνη ανάμεσα στις δύο κοινότητες, του Ρώμα και του ΜΗ. Επίσης, κάποια προφανή που μπορούμε να κάνουμε, να εξασφαλίσουμε ότι το κενό που έχουμε στις κοινωνίες μας, σε ό,τι αφορά την ηθαγένεια, ακόμα και τις ταυτότητες και επίσημα έγγραφα, ας πούμε, που θα δίνουν δυνατότητα στους Ρωμά να ταυτοποιούνται, να, να αποδεικνύουν ποιοι είναι. Μερικές φορές βέβαια το πρόβλημα είναι αμοιβαίο γιατί δεν έχουν ήδη πάει ε, στα ληξιαρχεία κτλ. Έχουμε δηλαδή ε, απάτριδες ανθρώπους στην Ευρώπη. Είναι σκανδαλώδες αυτό. Ε, υπάρχουν άνθρωποι στην Ευρώπη που ζουν ε, στην Ευρώπη, δεν έχουν ηθαγένεια, είναι απάτριδες και άρα δεν έχουν και τα δικαιώματα που συνοδεύουν την ηθαγένεια. Πρέπει να εξετάσουμε περαιτέρω την κατάσταση επίση τη εκπαίδευση και των σχολείων σε πολλέ χώρε. Έχουμε πολλά προβλήματα με τους Ρωμά, ε, γιατί θα τους βάζουμε σε ειδικά σχολεία, ειδικέ τάξεις, γιατί είναι Ρωμά, μόνο και μόνο γι' αυτό. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι και οι μαθητές Ρωμά θα έχουν το δικαίωμα να πάνε στα κανονικά σχολεία, στο κανονικό εκπαιδευτικό σύστημα, να φοιτήσουν σε κανονικά σχολεία. Η πολιτική εκπροσώπηση είναι ένα άλλο θέμα. Ελάχιστοι Ρωμά εκπροσωπούνται ε, στο Κοινοβούλιο ή έχουν έδρα στο Κοινοβούλιο. Και αυτό δείχνει το κενό ανάμεσα στην πολιτική και στην ε, καθημερινότητα των Ρωμά. Και υπάρχει ανάγκη να ξανασκεφτούμε το θέμα αυτό. Εδώ το στέλνω αυτό το μήνυμα προς τα πολιτικά κόμματα, τα οποία θα πρέπει να προσπαθήσουν να εξασφαλίσουν ότι οι Ρωμά αποκτούν δεξιότητες για κατάλληλες για την άσκηση της πολιτικής, για την πολιτική ζωή στις χώρες τους. Όλα αυτά τα βήματα όμως θα πρέπει να γίνουν ε, σε συνεργασία με τις κοινότητε των Ρωμά, όχι για αυτούς υπέρ αυτών λοιπά, αλλά μαζί με αυτούς. Στο παρελθόν κάναμε λάθη γιατί αποφασίζαμε κάποια πράγματα να τα κάνουμε για αυτούς και αυτό δεν είναι δημοκρατικό. Ευχαριστώ. Thank you very much, Mr. Was thinking... Ευχαριστούμε πολύ. Και είπα κάπου το ξέρω αυτό το όνομα, το Χάμαρμπεργκ, αλλά δεν είχα καταλάβει ότι ξεκινήσετε μια δεύτερη σταδιοδρομία ω ε, βουλευτή. Χαιρόμαστε που σα έχουμε μαζί μα σήμερα. Λοιπόν, α περάσουμε τώρα σε μια ανοιχτή συζήτηση με τα μέλη των Εθνικών ε, Κοινοβουλίων, αλλά και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στρέφαμε προ του ε, συναδέλφου Ευρωβουλευτέ. Θα θέλατε μήπω να πάρετε το λόγο? Ωραία. Θα ξεκινήσουμε όμως πρώτα με δύο μέλη ο κύριος Μοντσίλο Μαρτίνοβιτς πρώτος, βουλευτής από το Μαυροβούνιο. Θα μιλήσετε τη μητρική σας, η οποία δεν καλύπτεται επισήμως από το λογικό καθεστώς. Έχουμε μετάφραση βέβαια προς τα κροατικά. Κάπως έτσι θα γίνει λοιπόν. Θα δούμε μέχρι πού θα φτάσουμε με αυτή την πρόκληση η ισχύ βρίσκεται στην πολυμορφία μας. Βέβαια, θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Κύριο Μαρτίνοβιτ. Το πιο σημαντικό όμω σε αυτή την πρόκληση είναι να ανάψετε το μικρόφωνο σα. Right. Σας ευχαριστώ. για την πρόσκληση που απευθύνατε προς εμάς. Ήρθα εδώ να ακούσω τις ευέρτιστες πρακτικές που ε, μπορούμε να αντλήσουμε και να ελοποιήσουμε και στις χώρες μας. Εδώ έχουμε έρθει ως καλεσμένοι της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ που συνεργάζεται στενά ε, με την κοινότητα Ρωμά στο Μαυροβούνιο. Το Μαυροβούνιο είναι μια πολύ μικρή χώρα, υποψήφια προσέγγιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με κάτι πάνω από 600.000 ε, κατοίκους, το 1% των οποίων είναι Ρωμά. Σε ό,τι αφορά τις ευάλωτες ε, ομάδες στην κοινωνία μας, και πιο συγκεκριμένα τους Ρωμά, μπορώ να σας πω τα εξής από τη δική μας ε, εμπειρία, η οποία είναι μακρά, γιατί τα τελευταία δέκα χρόνια, η παλοπλούσια, γιατί τα τελευταία δέκα χρόνια έχουμε αναλάβει μία σειρά πρωτοβουλίες. Ε, καθώς υπήρξε και μία μαζική εισρωή Ρωμά από γειτονικέ χώρες. Ε, πολλοί από αυτούς είναι αναλφάβητοι πολύ φτωχοί που παρόλα αυτά ήθελαν να ενταχθούν στην κοινωνία μας. Γι' αυτό και εμείς ε, ακολουθήσαμε μια ολιστική προσέγγιση, τους βοηθήσαμε όπως μπορούσαμε με στέγαση, τροφή και προσπαθήσαμε να τους εντάξουμε στην κοινωνία μας με πολλές ε, ενέργειες στοχευμένες προς εκείνους, ε, κυρίως ό,τι έχει να κάνει με την ε, εκπαίδευση, από νηπιαγωγία μέχρι γυμνάσια, λύκεια και ακαδημαϊκή κατάρτιση. Μέχρι πριν από μερικά χρόνια δεν είχαμε καθόλου φοιτητές Ρωμά στα πανεπιστήμια. Σήμερα έχουμε 24. Η ίδια κατάσταση ισχύει και στην εκπροσώπηση των Ρωμά ε, στους δημόσιους θεσμούς ε, που βλέπουμε ότι η συμμετοχή τους αυξάνεται συνεχώς. Και προσπαθούμε να τους ε, επιτρέπουμε να συμμετέχουν και να τους εμπλέκουμε σε όλες τις δραστηριότητες του δημόσιου βίου και της κοινωνίας. Κάτι που είναι σημαντικό να σημειώσουμε εδώ είναι η υγειονομική περίθαλψη και φυσικά και η απασχόληση. Εργαζόμαστε με όποιο τρόπο μπορούμε για να εμπλέξουμε τους ε, Ρωμά και στην αγορά εργασίας και, αλλά και στον πολιτικό στίβο. Σε οποιαδήποτε μορφή ε, της ε, κοινωνίας μας. Σε πολιτικό επίπεδο λοιπόν προσπαθούμε να αναδείξουμε ε, πολιτικές προσωπικότητες από την κοινότητα Ρωμά και σε τοπικά, στο τοπικό επίπεδο και στο εθνικό. Ε, πολλοί έχουν ε, εντάξει Ρωμά στα ψηφοδέλτιά τους. Έχω πολλά ακόμα να σας πω, αλλά θα σταματήσω εδώ γιατί δεν έχω πολύ χρόνο στη διάθεσή μου. Όμως έχουμε προετοιμάσει υλικό, το οποίο μπορείτε να δείτε και να δείτε την εμπειρία που έχουμε αποκομίσει εμείς, που μπορεί να αποτελέσει και παράδειγμα προς προς, ε, για άλλους. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ήταν μεγάλη μου τιμή να συμμετάσχω στη σημερινή συζήτηση και ελπίζουμε να ε, εφαρμόσουμε στο Μαυροβούνιο τις βέλτιες πρακτικές που είδαμε εδώ σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Μαρτίνοβιτς. Ξέχασα να πω, να δώσω στους αδέλφους ένα χρονικό περιθώριο. Έχετε τρία λεπτά στη διάθεσή σας, δεν χρειάζεται να τα εξαντλήσετε, αλλά μετά τα τρία λεπτά θα έχω εδώ το σφυράκι μου. Να σας πω ποιος είναι στο κατάλογο μιλητών για να προετοιμάζεστε. Η κυρία Μαρσελίνη θα πάρει το λόγο σε λίγο. Μετά, Ρωμαίο Φράντς από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Ιβαν Μπάιτσκάι, Πρέντερακ Μπάκοβιτς, μετά η Τζούλι Βόρτ, Ευρωβουλευτής, και μετά βουλευτές Φέλσκο, Καστάζη και στο τέλος θα πάρω το λόγο εγώ και θα περάσουμε τώρα στο επόμενο πάνελ. Κατρίνα Μαρσελίνο από την Πορτογαλία. Obrigada, senhora Presidente. Ah, Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Καλό απόγευμα σε όλους. Θα ήθελα πολύ απλά Παρότι ήθελα να πάρω το λόγο στο δεύτερο πάνελ, αλλά δεν πειράζει. Ήθελα λοιπόν να σας πω ότι η Πορτογαλία εργάζεται άοκνα για την ε, κοινωνική ενσωμάτωση ε, των Ρωμά στην Πορτογαλία. Βέβαια, ο πληθυσμός Ρωμά στην Πορτογαλία είναι μικρότερος από ό,τι σε άλλες χώρες που εκπροσωπούνται εδώ. 50.000 άτομα περίπου στη χώρα μας. Είναι μια κοινότητα η οποία υφίσταται ε, σοβαρές διακρίσεις, όπως και σε άλλα κράτη-μέλη. Και αυτό Εντάξει, η κατάσταση μπορεί να είναι διαφορετική στην Ιβηρική Χερσόνησο σε σχέση με άλλε ευρωπαϊκέ χώρε, αλλά και πάλι υπάρχει κοινωνικό αποκλεισμό. Ε, υπάρχει εθνική στρατηγική, θέλουμε να εξετάσουμε αυτή την αναθεώρηση που υιοθετήθηκε. Η νέα στρατηγική είναι πιο φιλόδοξη, με στόχο ε, να επικεντρωθεί στην παιδεία, που είναι κέρια σημασία στοιχείο για τους ε, Αθήγανου. Πάνω από το ίμιση των ονομά στη χώρα μας είναι παιδιά. Οπότε, αν επικεντρωθούμε στον τομέα της εκπαίδευσης, είμαστε πεπισμένοι ότι θα υπάρξει πλήρης ενσωμάτωσή του στην κοινότητά μας στο μέλλον, στην κοινωνία μας. Ε, όλο ένα και περισσότερα παιδιά Ρωμά πηγαίνουν σχολείο κανονικά και είναι κάτι το οποίο θέλουμε πολύ σημαντικό ε, και σημαντική είναι και η συμμετοχή τους ε, στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση να πηγαίνουν όλα τα παιδιά σχολείο. Και έχουμε καταβάλει προσπάθειες και για την ε, ανώτατη εκπαίδευση, το λεγόμενο πρόγραμμα ΟΠΡΕ. Κλείνοντας, για την απασχόληση. Πρέπει να επενδύσουμε και στην απασχόληση, να ε, εμπνεύσουμε εμπιστοσύνη και στη στέγαση βέβαια, πρέπει να σταθούμε και με τα κονδύλια μας να δημιουργήσουμε και νέες ε, κατοικίες. Ιδάλλως δεν θα λυθεί καθόλου το πρόβλημα της στέγασης ε, των αθήγκανων Αυτά από μένα και μια τελευταία πρόταση, το ζήτημα της συμμετοχής των Ρωμά. Η εξέλιξη αυτή, εμείς, ε, αυτή που βλέπουμε εμείς δεν θα μπορούσε να σημειωθεί χωρίς τους Ρωμά. Πρέπει να τους εμπνεύσουμε και την επιθυμία να συμμετάσχουν ε, στα κοινά. Είναι θέμα λοιπόν και πολιτικής βούλησης προκειμένου οι Ρωμά να συμμετέχουν πλήρως ε, σε ό,τι έχει να κάνει με την κοινότητά τους. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστούμε κυρία Μαρσελίνο. Όσο εσείς μιλούσατε, λάβαμε και άλλα αιτήματα για ένταξη στο κατάλογο μελητών. Ο κύριος Ρώμιο Φράνς έχει το λόγο. Αγαπητοί συνάδελφοι. Ρώμεο Φράνς. Ονομάζομαι και προέρχομαι από την κοινότητα των Σύντη. Χαίρομαι πάρα πολύ που εδώ στο Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ συζητείτε το θέμα των θεμελιωδών δικαιωμάτων της ε, κοινωνικής ένταξης των Ρωμά και της καταπολέμησης του αντιαθήκανισμού. Λίγο κρίμα βρίσκω το γεγονός ότι η συνεδρία αυτή γίνεται πέμπτη απόγευμα που πολλοί ευρωβουλευτές πλέον λείπουν, έχουν φύγει. Είναι πολύ κρίμα που ε, προσκλήθηκαν λίγοι άνθρωποι με ε, καταγωγή από τις κοινότητες των ε, Ρωμά και των Σύντη. Διότι για εκείνους ε, πρόκειται άλλωστε. Αυτούς αφορά αυτή η συζήτηση. Θέλω να σας μιλήσω για το ποια είναι η κατάσταση στις χώρες μας. Ο αντιαθηγανισμός εμποδίζει την ίση πρόσβαση στην εργασία, στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και στη στέγαση. Ο αντιαθηγανισμός είναι είναι η ισχυρότερη ε, και πλέον ε, και καλυμμένη μορφή ρατσισμού στην Ευρώπη. Θα έπρεπε η καταπολέμηση του αντιαθηγανισμού να αποτελεί βασικό στοιχείο των στρατηγικών για την ε, κοινωνική ένταξη των Ρωμά. Γιατί δεν έχουν επιτευχθεί μέχρι στιγμής τα επιδιωκόμενα, γιατί δεν έχουν επιληθεί τα προβλήματα. Διότι δεν ε, έχουν ίδια, ίσα δικαιώματα οι Ρωμά. Ας πάρουμε ως παράδειγμα τη Γερμανία. Η γερμανική κυβέρνηση αποφάσισε ότι δεν απαιτείται εθνική στρατηγική για την κοινωνική ένταξη των Ρωμά, ενώ υπάρχουν μελέτες που αποδεικνύουν ότι τόσο στην εκπαίδευση όσο και στην αποδοχή ε, ε, των Ρωμά ως ισότιμων μελών της κοινωνίας υπάρχουν σοβαρότατα εμπόδια και προβλήματα. Αυτό αποτελεί σοβαρότατο εμπόδιο για τη συμμετοχή των ε, Ρωμά στην κοινωνική και πολιτική ζωή. Ας πάρουμε την, την περίπτωση της Ουγγαρία. Το ψήφισμα που εγκρίθηκε το 2018 εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με μεγάλη πλειοψηφία αποδεικνύει ότι τα παιδιά των Ρωμά δεν έχουν ίση πρόσβαση στην παιδεία. Και έτσι πάνω ε, από το μέσο όρο ε, βρίσκουμε παιδιά των ε, Ρωμά σε ειδικά σχολεία και μάλιστα ε, τους αποδίδονται ε, πνευματικές και ε, διανοητικές περιπτώσεις καθυστέρησης. Αυτό θυμίζει ναζισμό, θυμίζει περιθωριοποίηση κοινωνική. Μπορώ να σας δώσω πολλά παραδείγματα, αλλά το κοινό στοιχείο όλων των παραδειγμάτων είναι το εξής. Οι άνθρωποι που προέρχονται από τις κοινότητες των Ρωμά δεν λαμβάνονται σοβαρά υπόψη, δεν τους παίρνουν στα σοβαρά. Αν όμως δεν μεταχειριστούμε, δεν ε, αντιμετωπίσουμε ως ίσους τους Ρωμά, διατρέχουμε τον κίνδυνο σε 20 χρόνια να ξαναβερθούμε εδώ σε αυτή την αίθουσα και να συζητούμε και πάλι τα ίδια προβλήματα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ρώμεο. Ο κύριος Ιστφαν Πάσκαη από την Ουγγαρία έχει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί ευρωβουλευτές, κυρίες και κύριοι. Θέλω να αναφερθώ στη Γενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Στον ευρωπαϊκό πολιτισμό είναι μια έννοια γνωστή η μη διακριτική μεχείριση. Ακόμη και η χριστιανοσύνη ορίζει ότι όλοι οι άνθρωποι πρέπει να ζουν ίσοι ενώπιον του Θεού. Αν δεν χάσουμε αυτές τις δύο αρχές από την, από την προσοχή μας, τότε ξέρουμε πολύ καλά τι πρέπει να κάνουμε. Γνωρίζουμε πολύ καλά τι παίρνει από μας η Ρωμά. Τι είναι σημαντικό λοιπόν για τη συνεργασία μας. Όπως είπε και ο βουλευτής πριν από εμένα, αν τα παιδιά των Ρωμά που γεννιούνται σήμερα σε 10 ή 20 χρόνια μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να μην τους αντιμετωπίζουν σαν παιδιά με ειδικέ ανάγκες που χρειάζονται ειδική στήριξη, τότε θα έχουμε επιτύχει το στόχο μας. Εμείς στην Ουγγαρία θέλουμε να προχωρήσουμε με απτά μέτρα, πραγματικά και γνήσια. Και έχω και να το αποδείξω αυτό. Το 2011 ξεκινήσαμε μια πολύ σημαντική διαδικασία με τον τίτλο «Εθνική στρατηγική για την κοινωνική ένταξη των Ρωμά». Η στρατηγική αυτή είχε ως στόχο την ε, κοινωνική ένταξη των Ρωμά και στο πλαίσιο αυτής εγκρίναμε και μια διακήρυξη, ένα πολύ σημαντικό έγγραφο, στο οποίο καθορίζεται ο στόχος της συνεργασίας για την βελτίωση της κατάστασης διαβίωσης της μεγαλύτερης μειονοτικής ομάδας στην Ευρώπη. Στην Ουγγαρία λοιπόν έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο. Βεβαίως και υπάρχουν προβλήματα, είναι γνωστά, Πρέπει ακόμα να γίνουν πάρα πολλά προκειμένου να επιτύχουμε όλους μας τους στόχους. Μεταξύ 2011 και 2017 ο κίνδυνος που αντιμετωπίζουν ε, οι Ρωμά να ε, ζουν σε συνθήκες φτώχειας έχει μειωθεί από 34% στο 25%. Βελτιώθηκε η κατάσταση στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των Ρωμά. Έχουν καλύτερη πρόσβαση στη στέγαση, σε κοινωνικέ παροχές. Τα παιδιά των Ρωμά όλο ένα και περισσότερο εντάσσονται στους παιδικούς σταθμούς, τους παρακολουθούν, είναι δωρεάν, δεν, δεν υπάρχουν δίδακτρα ούτε τροφία. που αυτό ήταν ένα διαχρονικό πρόβλημα στην Ουγγαρία για τις κοινότητες των Ρωμά που ε, έχουμε αρχίσει και το ε, αντιμετωπίζουμε. από την Σλοβενία. Είναι ο επόμενος ομιλητής. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, είμαι Σλοβενός, Είμαι εθνικός βουλευτής και είμαι και αντιπρόεδρος της Επιτροπής Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Με βάση εκτιμήσεις ε, του, της τοπικής αυτοδιοίκησης ε, και διαφόρων άλλων φορέων υπάρχουν περίπου 7 με 10.000 ε, Ρωμά στη Σλοβενία. Η κατάστασή τους ρυθμίζεται από το Σύνταγμα της Σλοβενίας. Επίσης, Υπάρχει και μια συγκεκριμένη πράξη της κοινότητας στο Ρωμά ε, για τις δικές τους υποθέσεις, η οποία είναι υπό αναθεώρηση. Κανένα από τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχει ρυθμίσει την, ε, τα της κοινότητα των Ρωμά με δική τους πράξη. Ε, με βάση αυτή την πράξη γίνεται μια ετήσια έκθεση ε, προς την Βουλή μας, ε, κυρίως στην Επιτροπή Εσωτερικών. Η Επιτροπή συζήτησε αυτή την έκθεση στις 27 ε, Σεπτεμβρίου του 2018 και σύστησε η, η Βουλή, το Κοινοβούλιο να υιοθετήσει στην ολομέλειά της πριν το 2018 την έκθεση αυτή. Η κυβέρνηση υιοθέτησε και το Εθνικό Πρόγραμμα Μέτρων για τους Ρωμά από το 2017 μέχρι το 2021 με στρατηγικό στόχο την αύξηση της ένταξης του πληθυσμού των Ρωμά και της εξομοίωσης του κοινωνικό πληθυσμού. Έχουμε μια επιτροπή για την προστασία των Ρωμά και έχουμε και μια ειδική task force που αντιμετωπίζει τις προκλήσεις, που εξετάζει τις ιδιαίτερες προκλήσεις της κοινότητας αυτής και ετοιμάζει συστάσεις. Εγώ γνωρίζω πολύ προσεκτικά όλα τα προβλήματα και τις προκλήσεις της κοινωνίας, της κοινότητας μάλλον των Ρωμά. Ε, υπάρχουν πολλές προκλήσεις για την κοινότητα των Ρωμά. Τέσσερα βασικά προβλήματα είναι η εκπαίδευση, εργασία, συνθήκες διαβίωσης και η ασφάλεια των Ρωμά. Και τα τέσσερα αυτά πεδία, οι τέσσερις αυτοί άξονες είναι αλληλένδετοι. Η αντιμετώπιση των προκλήσεων πρέπει να γίνει λαμβάνοντας υπόψη το πλαίσιο, το γενικό, μέσα στο οποίο διαβίουν. Πρέπει να ξεκινήσουμε την εφαρμογή μέτρων πάρα αυτά. Αλλιώς χάνουμε την ευκαιρία που μας παρουσιάζεται. Έχουμε ένα όραμα για το πώς θα λύσουμε αυτά τα προβλήματα στη Σλοβενία. Καθορίζουμε τα προβλήματα, όταν τα εντοπίσουμε είναι πολύ πιο εύκολο να βρούμε και τη λύση τους. Δυστυχώς σήμερα δεν έχω αρκετό χρόνο για να μπω σε λεπτομέρειες και να σας παρουσιάσω τις πιθανές λύσεις σε όλα τα προβλήματα. Ίσως κάποια άλλη στιγμή μέσα στη μερινή συνεδρία θα μου δοθεί ευκαιρία. Η Julie Ward έχει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ πολύ τους συναδέλφους και το Κοινοβούλιο που οργανώνει αυτή τη σημαντική διάσκεψη. Από την αρχή που ανέλαβα εδώ, ε, ασχολούμαι άοκνα με το θέμα αυτό. Προσπαθώ να υπερασπίσω τα δικαιώματα όλων και παρεμπιπτόντως και μάλλον και όλους ιδιαίτερος για τους Ρωμά. Ζω σε μια περιοχή όπου έχουμε τη μεγαλύτερη εθνική μειονότητα των Ρωμά ε, σε μια ορεινή βόρεια περιοχή της Αγγλίας. Ε, έχουμε πολλούς Ρωμά εγώ δούλευα στον τομέα των τεχνών. Ετοιμάσαμε μια ταινία με παιδιά Ρωμά, όπου μας ε, μάθαιναν ε, τη γουλτούρα τους και μας, ε, εμείς, παίζαμε το ρόλο των γιαγιάδων τους. Ε, με εμπλούτησε αυτή η επαφή μου με την κουλτούρα των Ρωμά. Δεν είναι κάτι που κάνουμε για το καλό των Ρωμά. Νομίζω ότι μαθαίνουμε και οι δύο, κερδίζουμε και οι δύο με αυτό το διάλογο. Ε, είναι πολύ σημαντικό να μιλάς με τον άλλο, να έχεις αυτή τη διαπολιτιστική συνεργασία, να μοιράζεσαι πράγματα για την κουλτούρα σου και την κουλτούρα τους. Εάν δεν τους εντάξουμε πραγματικά, ε, θα χάσουμε ως ευρωπαϊκές κοινωνίες. Εγώ εκπροσωπώ την ε, βορειοδυτική Αγγλία. Από εκείνη την περιοχή προέρχεται. Και είμαστε σε μια ειδική ιστορική στιγμή, όπου έχουμε τεράστια ξενοφοβία, ρατσισμό, ισλαμοφοβία, όλες τις μορφές της φοβίας του άλλου. Όλες τις έχουμε. Και, ενώψη, και μάλλον πριν την, το δημοψήφισμα τον Ιούνιο του 2016 υπήρχαν ε, κάποια παιδιά Ρωμά που παίζανε στο δρόμο έξω. Συνηθισμένα είναι. Ούτω ή άλλω συνηθισμένο για οποιοδήποτε παιδί να βγαίνει στον δρόμο και να παίζει. Να ασκεί αυτό το δικαίωμα να, να παίζει έξω, στην Ήπεθρο. Και οι γονεί του φοβόταν τόσο πολύ, γιατί έχει αυξηθεί τόσο πολύ ο ρατσισμός σε αυτή τη χώρα λόγω της, του ακροδεξιού τύπου. Και αυτά τα παιδιά, επειδή υπάρχει αυτό το εχθρικό περιβάλλον, έκτοτε δεν ξανά ποτέ στον δρόμο. Το ξέρω πάρα πολύ καλά, γιατί ε, ασχολούμαι με τις... Ε, και συνεργάζομαι με ακτιβιστές που δουλεύουν στον χώρο της οργανώσης νεολαίας. Χρειάστηκε να δημιουργήσουμε ειδικό χώρο ε, στην κοινότητά μας για να μπορούν να παίζουν αυτά τα παιδιά. Και καλό είναι αυτό, αλλά είναι παράδεκτο το γεγονός ότι παιδιά, μικρά παιδιά δεν έχουν την ελευθερία να παίξουν δημιουργικά έξω στον δρόμο, στην πόλη που μένουν. Ήθελα να το πω αυτό, γιατί νομίζω ότι αυτό που συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη είναι ότι δεν υπάρχει καμία ανοχή για τον άλλο, πουθενά. Και το βλέπουμε ειδικά απέναντι στους Ρωμά. Εγώ έχω δουλέψει με το δίκτυο εγώ και με, με το, κίνημα, το μαζικό κίνημα κατά του ρατσισμού της στην Ευρώπη και βλέπω νέα παιδιά από άλλες κουλτούρες που συνεργάζονται μεταξύ τους γιατί θέλουν μια άλλη Ευρώπη ε, νομίζω ότι αν επενδύσουμε στην ε, εκπαίδευση, υψηλή ποιότητα εκπαίδευση με ένταξη των Ρωμά, δημιουργία χώρου για να ανταλλάξουμε εμπειρίε που προέρχονται από τι δικέ μα παραδόσει και κουλτούρε, θα έχουμε μια καλύτερη Ευρώπη. Σας ευχαριστούμε. Ας μην δίνουμε κι εμείς όμως ε, το κακό παράδειγμα, ε, τον χρόνο ομιλία. Ο κύριος Βέρσκο Κατσχάζη από την Κροατία. Ευχαριστώ πολύ. Βέρκο Καζάζη ονομάζομαι. Εκασωπώ 12 μειονότητες ε, στο Κροατικό Κοινοβούλιο. Μία από αυτές είναι και η κοινότητα Ρωμά. τα όσα ακούσαμε δεν προκαλούν έκπληξη, αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν ε, οι Ρωμά. Λυπηροί μεν, αλλά αληθινοί. Μας λένε ότι είμαστε τεμπέληδε, ότι δεν θέλουμε να δουλέψουμε, αυτά τα ακούμε εδώ και δεκαετίες. Η βελτίωση σε ό,τι αφορά τη στέγαση και την εκπαίδευσή μας ε, δεν είναι και τόσο σημαντική. Και όπου υπάρχει μάλιστα βελτίωση, αυτή δεν είναι λίγο οριακή. Οι καταστάσεις και συνθήκες διαβίωσης είναι αυτές περίπου που ήταν και τον 17ο-18ο αιώνα. Είναι πολύ άσχημα τα πράγματα. Σε ό,τι αφορά την απασχόληση, να σας πω το εξή. Μπορείτε να φανταστείτε να ζείτε σε μια διαρκή ύφεση, γιατί κάπως έτσι γεννιούνται και πεθαίνουν οι Ρωμά. Σε μία μόνιμη κατάσταση ύφεση. Ακούσαμε εδώ μια συζήτηση για την αξιολόγηση και εγώ θέτω το εξής ερώτημα. Έχετε στοιχεία για το πόσες ε, συστάσεις του ψηφίσματος έγιναν δεκτές από τα κράτη-μέλη και οδήγησαν τελικά σε συγκεκριμένα προγράμματα που να προκύπτουν απευθείας από το ψήφισμα και να μην προϋπήρχαν δηλαδή. Ευχαριστώ. Σωράγια, μπορείς να απαντήσεις στη συνέχεια σε αυτό το ερώτημα. Τελαρίτη Μαρία από την Ελλάδα. Ευχαριστώ θερμά την ε, Επιτροπή για την πρόσκληση για μια τόσο σημαντική διακοινοβουλευτική συνάντηση. Αναφέρθηκαν οι διακρίσεις που υφίστανται οι Ρωμά και μάλιστα στους περισσότερους τομείς, από τη μη συμμετοχή τους ή την πρόσβασή τους στις υπηρεσίες, μέχρι και τη μη συμμετοχή τους στα κοινά ή σε θέσεις ευθύνης. Ε, γνωρίζουμε όμως ότι η αντιμετώπιση εγνωριζουμε γνωριζουμε ομως ακραίων συνθήκων διαβίωσης που ζουν οι Ρωμά και αναφέρομαι στους καταβλισμούς που έχουν στις παρυφές συνήθω των πόλεων και τη διαβίωση φτώχεια που έχουν και κοινωνικού αποκλεισμού και ιδιαίτερα αυτή η περιθωριοποίηση είναι διαγενακή θα λέγαμε και ως εκ τούτου απαιτεί και σταθερή πολιτική βούληση από τα κράτη-μέλη, στρατηγικό σχεδιασμό, ικανό διοικητικό μηχανισμό, δέσμευση αναγκαίων πόρων και φυσικά και βέβαια την ενεργητική συμμετοχή του ίδιου του πληθυσμού. Εδώ θα συμφωνήσω με τον εισηγητή που είπε ότι οι πολιτικές που είχαμε μέχρι τώρα ένταξης για τους Ρωμά ε, ε, ε, ε, γινόταν μέσα από τα προγράμματα της στόχιας και αυτό παρέλειπε βασικά στοιχεία από την ίδια την ομάδα έως και τον ε, ε, έως και την αθηναγκονοφοβία θα λέγαμε, τη φοβία δηλαδή προς τους τυγκάνους. Εγώ από την εμπειρία μου 10 χρόνια στο, το τερέν παρέμβαση στην αξιοποίηση πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους Ρωμά θα ήθελα να εντοπίσω ότι αυτό που λείπει πάρα πολύ είναι ο συντονισμός και ολοκληρωμένος χαρακτήρας αυτών των παρεμβάσεων από το εθνικό στο τοπικό επίπεδο και γι' αυτό χαίρομαι που αυτό έχει εντοπιστεί και εκφράζεται μέσω μια στρατηγική που πρέπει να έχει κάθε χώρα, να την εξειδικεύει και να πηγαίνει στο περιφερειακό και στο τοπικό επίπεδο, που είναι πολύ σημαντικό, γιατί ακριβώ στο τοπικό επίπεδο έχουμε και τι πολλέ διακρίσει με τη σύγκρουση αυτών των δύο κοινοτήτων. Και νομίζω ότι εκεί πρέπει να δώσουμε ένα ιδιαίτερο βάρο, γιατί εκεί πρέπει να χτυπήσουμε πάρα πολύ αυτή την αυτόν τον αντιθυγκανισμό. Τέλος, θα ήθελα να εντοπίσω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτές οι ετήσιες ε, εκθέσεις πεπραγμένων, γιατί μας δίνει τη δυνατότητα να δούμε ότι προγράμματα ευρωπαϊκά κατά πόσο φτάνουν στον τελικό δικαιούχο, όπως λέμε. Δηλαδή, ο ίδιος ο πληθυσμός κατά πόσο ωφελείται από αυτά τα προγράμματα και όχι η ενδιάμεση. Τέλος, θα ήθελα να πω ότι για μένα είναι επίσης σημαντικό να γίνει πιο, με μεγαλύτερη σαφήνεια και να φύγει αυτό που λέτε οι εθνικές επιτροπές συμφιλίωσης και δεν θυμάμαι ακριβώς πώς το είπατε, που ε, περιγράφεται μέσα στις κατευθύνσεις ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ νομίζω ότι ε, πολύ σημαντικό παίζει ρόλο αυτό που είπατε, τα σημεία που, κινούν όλα και εμεί στη χώρα μας το διαπιστώνουμε αυτό γιατί μετά την σύσταση της ειδική γραμματείας για, την, ε, για τα θέματα των Ρωμά βλέπουμε ότι εκπορεύονται από ένα όργανο όλες αυτές οι πολιτικές και έτσι έχουμε τη δυνατότητα να τις παρακολουθήσουμε. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και νομίζω πρέπει να το δούμε, δηλαδή το συντονισμό, ε, τις στρατηγικές αλλά και τα, την υλοποίηση μέσω της κινητοποίησης των αρχών έτσι ώστε να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η κυρία Εύα Μαϊταϊσόφα από την Τσεχία έχει το λόγο. Ε, Ευχαριστώ κυρίε και κύριοι. Από την Επιτροπή Οικογενειών και μειονοτήτων του Τσεχικού Κοινοβουλίου. Θα ήθελα να μου δώσετε περισσότερε πληροφορίε σχετικά με βέλτιστε πρακτικέ που ακολουθούνται σε άλλα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την κοινωνική ένταξη των Ρωμά και άλλων μειονοτήτων. Πιστεύω ότι φυσικά η αθηγανοφοβία είναι ένα εξαιρετικά αρνητικό φαινόμενο, δεν έχει καμία δουλειά στην κοινωνία μας και πρέπει να καταπολεμηθεί. Από την άλλη πλευρά όμως θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να λαμβάνετε υπόψη και το υπόβαθρο, το ιστορικό, τα, τα, τα αίτια που έχουν οδηγήσει στον αντιαθηγανισμό. Αυτά πρέπει να καταπολεμηθούν. Πρέπει να ενισχύσουμε την ε, κατανόηση και να φωτίσουμε αυτή τη διάσταση που επηρεάζει την ε, καθημερινότητα των πολιτών μας. Νομίζω ότι επίσης πρέπει να αναδειχθεί το θέμα της γλώσσας. Πρέπει να υπάρξει κοινή ε, γλώσσα επικοινωνίας. Πολλές φορές οι Ρωμά δεν μιλούν τη γλώσσα της χώρας στην οποία διαμένουν. Ούτε από την άλλη μεριά βέβαια ξέρω κάποιους από το γενικό πληθυσμό που, να, που θα μπορούσαν να, να, μιλάνε τη, τη γλώσσα των Ρωμά ώστε να διευκολυνθεί η επικοινωνία. Όλα αυτά πρέπει να τα πάρουμε υπόψη μας. Μιλάμε για σχολικά εγχειρίδια για παράδειγμα τα οποία θα μπορούσαν να μεταφραστούν για να ενισχυθεί η συμμετοχή των Ρωμά στην κοινωνική ζωή των τοπικών κοινωνιών στις οποίες ζουν. Ξέρετε μέλη του γενικού πληθυσμού που ξέρουν τη γλώσσα των Ρωμά, που κατέχουν τη γλώσσα των Ρωμά διότι τέτοιοι άνθρωποι ενδεχομένως θα ήταν πιο κατάλληλοι ώστε να έρθουν σε μια πρώτη επαφή με τις ε, κοινότητες των, των Ρωμά. Θα μπορούσαν να γίνουν ε, πιο πολύ δεκτοί, αν θέλετε, από τις κοινότητες των Ρωμά. Τέτοιες επιτροπές θα μπορούσαν ε, θα μπορούσαν να διευκολύνουν το επιτόπου έργο που διεξάγεται. Ενδιαφέρουσα ερώτηση, λέει η Πρόεδρο. Ελπίζω να απαντήσει κάποιο. Τελευταία ομιλήτρια, εγώ. Θυμάμαι πολύ καλά ότι είχαμε διεξαγάγει μια συζήτηση, συναισθηματικά φορτισμένη θα πω, εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η οποία και μας οδήγησε να ζητήσουμε την θέσπιση εθνικών στρατηγικών για την ένταξη των Ρωμά στις κοινωνίες των κρατών μελών. Αυτό, μάλιστα, είχε γίνει έπειτα από ένα σκάνδαλο στην Γαλλία όπου Ρώμα που δεν κατήχαν ε, τη γαλλική υπηκότητα εξορίστηκαν με έναν μαζικό συλλογικό τρόπο χωρίς να εξετάζεται η, κάθε περίπτωση ξεχωριστά ως μαζικό μέτρο το οποίο οδήγησε σε κατακραυγή σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση για τον τρόπο με τον οποίο μια κυβέρνηση εκείνη την εποχή προσέγγισε το θέμα φαινόταν να έχει ξεχάσει τα ατομικά δικαιώματα. Αυτή, αυτό το περιστατικό οδήγησε το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στο να συμφωνήσουν για την ανάγκη ενίσχυση των προσπαθειών όσον αφορά την κοινωνική ένταξη των Ρωμά. Και εδώ θέλω να σταθώ σε αυτό που είπε ο Ρέο Φραντς για την ε, γερμανική ομοσπονδική κυβέρνηση, η οποία αποφάσισε να μην καταρτήσει εθνική στρατηγική για την ένταξη των Ρωμά. Και νομίζω ότι αυτό το ε, ερώτημα θα μπορούσε να μας το απαντήσει ο κύριος Μακ. Πράγματι ισχύει αυτό. Και αν ισχύει, για ποιο λόγο ελήφθη αυτή η απόφαση. Και αν όντω ισχύει, πιστεύετε ότι ήταν σωστή αυτή η κίνηση, αυτή η απόφαση της γερμανικής κυβέρνησης. Και επίση να απευθύνω ένα ερώτημα στο, στους ομιλητές του πάνελ. Πώς, παρά το γεγονός ε, ότι κύριε Μακ, κάνατε μια ιστορική ανασκόπηση και συγκρίνατε την μεταχείριση των ε, ε, Εβραίων από τους Ναζί με, με που επεφύλαξαν στους Ρωμά, πώς δεν καταδικάζεται στη σημερινή κοινωνία ο αντιαθηγανισμός με τον ίδιο τρόπο που ε, καταδικάζεται ο αντισημιτισμός. Λοιπόν, να ξαναδώσω το λόγο στους ομιλητές μας, σοράγια post και μετά με την ίδια σειρά με την οποία τοποθετήθηκαν και στην πρώτη φάση της συζήτησης. Ευχαριστώ. Να σχολιάσω καταρχήν τα όσα είπατε εσείς πρώτα. Η εκπαίδευση, νομίζω, είναι βασικό εργαλείο για την ένταξη, μια επιτυχή ένταξη, προφανώς. Υπάρχει ειδική εκπαίδευση Πρέπει να εκπαιδευτούν και οι μη για την ιστορία τους και την πολιτιστική κληρονομιά των πολιτών. Είτε είναι Ρωμά είτε δεν είναι Ρωμά. Γιατί επί αιώνες οι Ρωμά στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες διαβιούσαν δίπλα μας. Υπάρχει μια κοινή πολιτιστική κληρονομιά και το γεγονός ότι οι υπόλοιποι πολίτες δεν γνωρίζουν ε, τα αρνητικά βιώματα των Ρωμά και τις ε, δυσκολίες που πέρασαν επί αιώνες, ε, είναι προβληματική. Πρέπει να εκπαιδευτούν και οι δύο, και οι Ρωμά και οι μη Ρωμά. Είναι σημαντικό για να υπάρξει εμπιστοσύνη αυτό. Γιατί αν είσαι αποκλεισμένο, αν είσαι μειονότητα και αν έχεις αρνητικές εμπειρίες επί αιώνες όπως έχουν οι Ρωμά, δεν είναι εύκολο να πιστέψεις είναι εμπιστευθείς κάποιους και να πιστέψεις ότι αυτά τα project που ετοιμάζουν άλλοι, ας πούμε για λογαριασμό σου, θα έχουν καλά αποτελέσματα. Ήδη από τη φάση του σχεδιασμού ενός project και ενός προγράμματος θα πρέπει με τη συμμετοχή των Ρωμά και με κοινή πορεία να προχωρήσουμε. Γι' αυτό μίλησα για τις Επιτροπές ε, Συμφιλίωσης στην ε, Σουηδία, το κάναμε αυτό στη Σουηδία, δημιουργήσαμε και μία λευκή βίβλο, ετοιμάσαμε μια λευκή βίβλο από την, όπου απαριθμούσαμε την ιστορία ε, όλου του 20ου αιώνα και ετοιμάσαμε και ε, ένα μάθημα ειδικό για τους μαθητές δημοτικών, για να καταλάβουν όλοι Πώ φτάσαμε στη σημερινή κατάσταση. Όλοι πρέπει να το, να το καταλάβουν. Πώ αυτέ τι ε, πλούσιε και πολιτισμένε κοινωνίε, πώ γίνεται στην Ευρώπη ακόμα να έχουμε 12 εκατομμύρια ανθρώπου οι οποίοι ζουν έτσι. Εγκαταλελειμμένοι. Πρέπει να καταλάβουμε την ιστορία. Πρέπει να καθαρίσουμε την ιστορία, να την αναγνωρίσουμε την ιστορία και να, και, να ε, δημιουργήσουμε ένα νέο κεφάλαιο ισότητας με την ένταξη στο μυαλό και την ισότητα στο μυαλό. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ίδια την έκθεση, κοιτάξτε την, έχω βάλει και κάποια αντίτυπα. Έχουμε 12 σελίδες σε αυτή την έκθεση με συστάσεις και προτάσεις. Πώς ξεκίνησε αυτό? Αλλά σύντομα, λέει η Πρόεδρος. Σύντομα, ναι. Ήμουνα ακτιβίστρια για 40 χρόνια. Ποτέ δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε για την αθηγανοφοβία. Ποτέ δεν μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ειδική μορφή α, ρατσισμού πάντα θεωρούνταν κοινωνικό πρόβλημα. Γιατί? Γιατί κανείς δεν αναγνώριζε ότι υπήρχε ο αθηγαν, αντιαθηγανισμός και αθηγανοφοβία. Το 2000, ή μάλλον με την πρώτη έκθεση, τον Απρίλιο του 2015, αναγνωρίζουμε για πρώτη φορά την αθηγανοφοβία. Και έκτοτε όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα χρησιμοποιούν αυτό τον ορισμό και καταλαβαίνουν ότι αυτό είναι η αιτία όλων των υπόλοιπων κοινωνικών προβλημάτων για τους Ρωμά. Αυτή ήταν η απαρχή. Στο ίδιο ψήφισμα επίσης αναγνωρίσουμε και το ολοκαύτωμα των Ρωμά, το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Ξεκινήσαμε σιγά σιγά, αλλά ήταν πολύ σημαντικό να δημιουργήσουμε μια πλατφόρμα για να υπάρξει αναγνώριση αυτής της ειδική μορφής ρατσισμού. Όσο πιο γρήγορα αναγνωρίζουμε το πρόβλημα, τόσο πιο εύκολα ε, το επιλύουμε. Επίσης, για το θέμα της γλώσσας. Υπάρχουν μη Ρωμά που μιλάνε τη γλώσσα των Ρωμά. Είναι περίεργο και νομίζω ότι είναι αποτυχία της χώρας. Εάν α, οι Ρωμά, ας πούμε, οι ίδιοι δεν μιλάνε τη γλώσσα της χώρας στην οποία ζουν. Είναι λόγω απομόνωσης στο σχολείο, ας πούμε. Μήπως επειδή ζούμε σε απομονωμένα μέρη, αν δεν είσαι ενταγμένος. Ας πούμε, αν μιλάτε εσείς ελληνικά μαζί μου, ε, εάν ζω μαζί σου στην Ελλάδα, ας πούμε, και τα λοιπά, λογικά θα πρέπει να έχω μάθει ελληνικά. Μήπως αυτό είναι το, το μήνυμα που στέλνει στον επόμενο μιλητή για να πάρει τη σκητάλη από σένα. Ναι, ναι, ναι, θα του δώσω το λόγο. Μάλιστα, κύριε Δημητρακόπουλε, ε, μιλήστε για αυτά που θεωρείτε ότι σας αφορούν και σας παρακαλώ λακωνικά όμως. Ναι, θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομο και να κάνω το εξή σχόλιο. Πολύ συχνά η δουλειά για την ένταξη των Ρωμά γίνεται ή σχεδιάζεται ε, υπό φιλανθρωπικούς όρους. Είναι φτωχοί καημένοι, υποφέρουν, πρέπει να τους βοηθήσουμε. Είμαστε χριστιανοί και με βάση τη θρησκεία μας πρέπει να βοηθήσουμε τους άλλους. Ε, μπράβο, αξιέπαινο είναι αυτό και καλό. Όμως, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι το θέμα αυτό είναι θέμα διαχείρισης και κυβερνήσεων. Ε, οι κυβερνήσεις έχουν υποχρεώσει απέναντι στους πολίτες να τους αντιμετωπίζουν ισότιμα, ανεξάρτητα από το αν είναι άντρες ή γυναίκες, ανεξάρτητα από τη θρησκεία τους, ανεξάρτητα από την πιθανή ας πούμε, αναπηρία τους ή από τις διαφορές τους. Λοιπόν, τώρα, από τη σκοπιά του οργανισμού μου, πολύ σύντομα τέλη Νοεμβρίου θα ετοιμάσουμε μια έκθεση για ό,τι σημαίνει ε, να είσαι μαύρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είτε σας αρέσει είτε όχι, δυστυχώς ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση το χρώμα του δέρματός σου μετράει ακόμα. Είναι μια πραγματικότητα. Πρέπει να την μετωπίσουμε και επηρεάζει και τους μαύρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους Ρωμά και οποιονδήποτε μοιάζει διαφορετικός. Είναι ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με τους παλιούς εφιάλτες στο Μεσοπόλεμο και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πρέπει να το αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα γιατί δεν το έχουμε ξεπεράσει. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μάκ. Ευχαριστώ. Πράγματι στη Γερμανία υπάρχει ένα τέτοιο σύνολο μέτρων και η δική μας οργάνωση επέκρινε το ενδεχόμενο μια κυβέρνηση απλώς να επιβάλλει μια ε, κοινωνική πολιτική κατά της φτώχειας που δεν θα κατανομάζει όμως τον αντιαθεγγενισμό. Μια εθνική μειονότητα που είναι πολίτες με χώρες εδώ και αιώνες δεν γίνεται να... Ε, ξεχωρίζει και να τη δείχνουμε το δάχτυλο ως μία μειονότητα που θα πρέπει κάπως να ενταχθεί στην κοινωνία. Επομένως είναι σημαντική βελτίωση τα τελευταία χρόνια που κατονομάζουμε το φαινόμενο του αντιαθηγανισμού και δεν κοιτάζουμε μόνο τους Ρωμά, κοιτάζουμε πλέον την κοινωνία. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι πάντα η αντίσταση και ο ακτιβισμός των Σύντη και των Ρωμά ήταν εκείνη που ανέδειξε το ζήτημα αυτό. Ε, όπως και με την αναγνώριση του ολοκαυτώματος. Εμεί γι' αυτό κατακρίνουμε το γεγονό ότι πολλές φορές κυβερνήσει λένε αυτό ανήκει σε αυτό το τομέα και σε αυτό το Υπουργείο, αυτό το, στο άλλο. Αλλά δεν τα κοιτάζουμε σφαιρικά και συνολικά τα πράγματα. Εμεί τώρα συνομιλούμε με την κυβέρνηση για να φροντίσουμε η Γερμανία να αναλάβει ηγετικό ρόλο και στο πλαίσιο τη υπερχόμενη Προεδρία τη το 2020. Θα πρέπει να συνεργαστούμε σε αυτό το τομέα, λοιπόν. Για το δεύτερο ερώτημα. Γιατί υπάρχει τόσος αντιαθηγανισμός ε, στην κοινωνία μας και γιατί δεν υπάρχουν κυρώσεις, γιατί δεν υπάρχει αντίδραση, κοινωνική κατακραυγή. Έχουμε ουσιαστικά κάτι το οποίο είναι κοινωνικά αποδεκτό και όλοι εμείς Έχουμε πολύ σημαντικό ρόλο να παίξουμε. Δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε ω ένα ζήτημα που θα αναλάβουν ε, ή τα Υπουργεία σε πλαίσιο προγραμμάτων. Χρειαζόμαστε πολιτική βούληση και έναν διάλογο που δεν θα κοιτάζει μόνο του Ρωμά, αλλά την κοινωνία εν γέννη με όλε τι ευθύνε τη. Και χαίρομαι που τουλάχιστον στη Γερμανία δημιουργήσαμε και καταλήξαμε σε μια συνένεση μεταξύ δημοκρατικών κομμάτων για μια αλλαγή νοοτροπία για επιβολή πλέον κυρώσεων ε, για τον αντιαθηγανισμό. Και έχουμε πλέον και την Ειδική Επιτροπή. Με ικανοποίηση είδα ότι και ε, γενικά την, στην Ευρώπη όλο είναι και περισσότεροι Ρωμά συμμετέχουν και στα εθνικά κοινοβούλια. Αυτό είναι κάτι το πολύ, πολύ θετικό και ελπίζω να συμβεί και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο μέλλον. Ευχαριστώ κύριο Χάμαμπεργκ. Ευχαριστώ. Συμφωνώ με όσα υπόθηκαν, παρότι είναι πολύ λίγοι ακόμα οι βουλευτές Ρωμά ε, στην Ευρώπη. Πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Υποεκπροσωπούνται οι Ρωμά σε σχέση με το μέγεθος ε, της κοινότητάς τους στις επιμέρους χώρες. Μία σημαντική αλλαγή που έχει γίνει εδώ στις Βρυξέλλες όμως σε αυτή τη συζήτηση παλιότερα, απλώς διαπιστώναμε τα προβλήματα σε ό,τι έχει να κάνει με την εκπαίδευση, τη γενομική περίθαλψη, την απασχόληση και τα βλέπουμε μόνο ως ένα κοινωνικό πρόβλημα. Φυσικά και είναι κοινωνικά προβλήματα, αλλά κάτι το οποίο αναφέρθηκε πολύ σωστά σε αυτή τη συνεδρίαση είναι ότι πλέον εξετάζουμε την αιτία αυτών των προβλημάτων που είναι ο αντιαθηγανισμός. Πρέπει λοιπόν να αρχίσουμε μία σοβαρή ενημέρωση και του γενικότερου πληθυσμού για το ζήτημα, για το θέμα δηλαδή της ε, κουλτούρας και των δικαιωμάτων των Ρωμά. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να περάσει στα κοινοβούλια ανά την Ευρώπη. Γιατί υπάρχει στήριξη ενεργειών κατά του αντισηματισμού και όχι αντίστοιχη στήριξη για ενέργειες κατά του αντιαθηγανισμού. Η εξήγηση πιστεύω ότι είναι ότι υπάρχει τέτοια καταπίεση προς τις ε, κοινότητε Ρωμά που είναι πολύ δύσκολο για εκείνες να οργανωθούν ε, όπως έχει κάνει η εβραϊκή κοινότητα ευτυχώς. Επομένως, ε, η έλλειψη κατανόησης είναι αυτό που προκύπτει από την γενικότερη κουλτούρα του γενικού πληθυσμού. Ποιο δημιουργεί το πρόβλημα. Φυσικά και υπάρχουν και προβλήματα από την πλευρά των ε, Ρωμά, αλλά το βασικό πρόβλημα είναι ε, η αντίδραση του γενικού πληθυσμού. Αυτό πρέπει να αναγνωρίσουμε για να σημειώσουμε πρόοδο. Κλείνουμε δυναμικά το πρώτο πάνελ. Θα έχουμε τώρα μια αλλαγή φρουράς. Ευχαριστώ τους καλεσμένους του πρώτου πάνελ. Θα συνεχίσουμε εντός ολίγων λεπτών με το δεύτερο. Όποιος θέλει να πάρει το λόγο μπορεί να μας δώσει τα δελτία του. Έχουμε την κυρία Παστουτσόβα από την ε, Τσεχική Δημοκρατία. Σας έχω σημειώσει ήδη ως πρώτη ομιλήτρια του δεύτερου πάνελ. Επιστρέφουμε. Okay, I do understand it's Thursday afternoon and we're not going to go a minute over time. Λοιπόν, λοιπόν δεν θα περβούμε το χρονικό όριο ούτε κατά ένα λεπτό. Πρέπει να κλείσουμε στις 6 ακριβώς. Επίση, καταλαβαίνω ότι θέλετε και λίγο να περπατήσετε και κάποιοι θέλουν και να καπνίσουν, που είναι πολύ δύσκολο σε αυτό το κτίριο, γι' αυτό κάποιοι έχουν βγει εκτός. Εγώ βέβαια δεν καπνίζω, οπότε συνεχίζω απευθείας. Ε, δεύτερο πάνελ για την κλιμάκωση των στρατηγικών Ρωμά και καταπολέμηση του αντιαθηγανισμού. Και στρέφαμε τώρα στις σημειώσεις μου. Στη δεύτερη συνεδρίαση τη Δικοινοβουλευτική Επιτροπή. θα συζητήσουμε πιθανέ λύσει για την περαιτέρω ανάδειξη των στρατηγικών ε, για τους Ρωμά, όπως ε, ανέφερε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισμα που υιοθετήθηκε πέρυσι. Ω συνέχεια, ως προς αυτό το ψήφισμα, η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ έχει ε, παραγγείλει μία μελέτη σε αυτό το τομέα για να έχουμε και τα στοιχεία από εμπειρογνώμονες που θα τροφοδοτήσουν τις μελλοντικέ μας εργασίες. Η μελέτη θα δημοσιοποιηθεί στη συνέχεια της χρονιάς και θα έχουμε και τα πρώτα πορίσματα και ευρήματα που θα μας δώσουν τροφή για τις περαιτέρω ενεργές μας. Λοιπόν, θα σας ε, αναφέρω και πάλι τη δομή της συζήτησης. Έχουμε κάποια γαλάζια έντυπα. Αν κάποιος θέλει να πάρει το λόγο πρέπει να συμπληρώσει αυτό το έγγραφο για όποιον προέρχεται από Εθνικά Κοινοβούλιο. Ε, οι ευρωβουλευτές ε, τα γνωρίζουν, απλώς ε, μου κάνουν ένα νεύμα, σας βάζω στον κατάλογο μελετών και θα υπάρχει και πάλι αυτή η αναλλαγή μεταξύ ευρωβουλευτών και βουλευτών. Θα δούμε και πώς θα ζητήσουν το λόγο τελικά, αλλά θα σας επισημάνω πόσο χρόνο έχετε στη διάθεσή σα. Με δεδομένο πρέπει να κλείσουμε μέχρι τι 6. Το λόγο τώρα θα πάρει η κυρία Λίνα Βοσιλιούτε. Αυτή είναι η πρόκληση στο κοινοβούλιο με τα δύσκολα ονόματα. Είναι ανώτερη ερευνήτρια στο Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών, το ΣΕΠΣ, πολύ γνωστό εδώ στις Βρυξέλλες και είναι μία εκ των συντακτών ε, που... της έκθεσης που ζήτησε το Κοινοβούλιο. Κυρία Βοσλιούτε, έχετε το λόγο για 10 λεπτά. Παρακαλώ. Thank you. And I will have a power... Ευχαριστώ. Έχουμε και μια παρουσίαση PowerPoint, την οποία μπορείτε να παρακολουθήσετε στις οθόνες. Uh, λοιπόν, καταρχάς θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση που μας απευθύνατε και που ζητήσατε την εκπόνηση αυτής της μελέτης. Ευχαριστούμε την ε, Γενική Διεύθυνση IPOL για το γεγονός ότι μας βοήθησε με όλα τα πρακτικά και οργανωτικά θέματα. Βασικά πορίσματα της μελέτης. Βρισκόμαστε εδώ στην αρχή της ε, ερευνητικής μας διαδικασίας. Βλέπετε εδώ το το χρονοδιάγραμμα της μελέτης. Η μελέτη θα εκπονείται και θα ολοκληρωθεί το Νοέμβριο το 2018. Είναι μια πολυεπίπεδη και πολυτομιακή μελέτη, στην οποία συμμετέχουν εθνικοί εμπειρογνώμονες, συντάκτες. Στην προσπάθεια να την ολοκληρώσουμε έχουμε καλύψει 7 κράτη-μέλη προκειμένου να δούμε ποιες είναι οι εμπειρίες που συλλέγονται σε εθνικό επίπεδο. Έχουμε έρθει σε επαφή με εθνικά υπουργεία, με οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών, για να δούμε τι έχει γίνει και τι πρέπει να γίνει στο μέλλον. Όπως βλέπουμε εδώ στους μηχανισμούς ε, κατανομής εξουσιών, αυτή τη στιγμή εμείς επικεντρωθήκαμε στον οικονομικό ε, αποκλεισμό και συζητήθηκε και στην προηγούμενη συζήτηση πώς οι πληθυσμοί των Ρωμά έχουν ε, 17 χρόνια μικρότερο προσδόκιμο ζωή από ότι ο γενικό πληθυσμό, ή πώ είναι δυνατόν ακόμη να μην έχουν πρόσβαση σε καθαρό νερό, σε εγκαταστάσει προσωπικής υγιεινής που θεωρούνται πλέον αυτονόητε για τον γενικό πληθυσμό. Λόγος ε, αυτής της κατάστασης, μεταξύ άλλων, είναι βεβαίως η έλλειψη πολιτικής εκπροσώπησης, ο αντιαθυγκανισμός και η θεσμική διακριτική μεταχείριση. Παρά το γεγονό λοιπόν ότι έχουν ε, δοθεί 9 δισεκατομμύρια ευρώ για την αντιμετώπιση και την άρση του αποκλεισμού, εξακολουθούμε να διαπιστώνουμε ότι τα θετικά αποτελέσματα είναι πάρα πάρα πολύ περιορισμένα. Μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις γίνονται και βήματα προς τα πίσω όσον αφορά τη ρητορική μίσους για παράδειγμα ή τα εγκλήματα μίσους που διαπράττονται στην Ευρώπη. Κάτρα τη γνώμη μας αυτά είναι τα κενά που υπάρχουν ακόμη σε, αυτό το, σε αυτή την τελευταία κοινωνικά αποδεκτή μορφή του ρατσισμού που πρέπει άμεσα να αντιμετωπιστεί. Κοιτάζοντας λοιπόν και στρέφοντας το, μέλλον, το, το βλέμμα μας στο μέλλον για το πώς θα ενισχύσουμε την ένταξη των Ρωμά και θα καταπολεμήσουμε τον αντικαθηγενισμό, καταφέραμε και καταλήξαμε σε, βασικές, σε βασικές δομικές μονάδες που θα μας οδηγήσουν σε αυτό. Πρώτον, Καλύτερη διακυβέρνηση, ισότητα και μη διαχείριση. Δεύτερον, χρειάζεται να οικοδομηθεί εμπιστοσύνη. Αυτό θα μπορούσαν να, ε, αυτόν τον ρόλο θα μπορούσαν να, επιτελέσουν αυτές οι ομάδες αλήθειας και συμφιλίωσης που θα αναγνωρίζουν τον ιστορικά βαθιά ριζωμένο αντιανθηγανισμό στον πληθυσμό. Τρίτο δομικό στοιχείο, κράτος δικαίου γιατί οι διακρίσεις πλήττουν όχι μόνο τους Ρωμά, αλλά την ίδια τη δημοκρατική νομιμοποίηση, τα εχέγγυα, τις εξασφαλίσεις του δημοκρατικού πολιτεύματος και την αντιμετώπιση εγκλημάτων μίσους. Πρέπει να εξασφαλιστεί ότι η δημοκρατία και το κράτο δικαίου θα εφαρμόζονται σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση με ομοιόμορφο και ίσο τρόπο. Και αυτό είναι και πάγιο αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πολιτική συμμετοχή των ε, Ρωμά. Εδώ έχουν γίνει πολλά. Αλλά το στοιχείο αυτό πρέπει να αποτελέσει στοιχείο και των μελλοντικών εθνικών στρατηγικών. Η αυτοεκπροσώπηση και η ενίσχυση των κοινοτήτων των ΟΜΑ πρέπει να ληφθεί σοβαρότερα υπόψη. Επίσης, λάβαμε υπόψη μας τοπικά σχέδια κοινωνικής ένταξης των Ρωμά. Έχει υποθεί. Χρειαζόμαστε πιο ολοκληρωμένες, πιο ολιστικές, αν θέλετε, ε, προσεγγίσεις ε, που θα αντιμετωπίζουν βασικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι Ρωμά στις τοπικές τους κοινωνίες. Λοιπόν, γιατί υπάρχουν προκλήσεις όσον αφορά την αρχή του κράτους δικαίου. Αυτή τη στιγμή η Ευρώπη είναι η πιο πλούσια ήπειρο στον κόσμο με το πιο προηγμένο νομικό και πολιτικό σύστημα. Παρ' όλα αυτά δεν έχει τα εργαλεία για την άρση και την αντιμετώπιση συστηματικών και θεσμικών παραβιάσεων των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ε, Ρωμά. Οι φορείς ε, του μίσους, όλο ένα και περισσότερο διαπιστώνουμε ότι δεν καταλήγουν στη δικαιοσύνη. Τι μπορεί να κάνει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση Θα μπορούσε για παράδειγμα να ε, εξετάσει ορισμένες υποθέσεις από κοινού προκειμένου να καταλήξει και το δικαστήριο σε νομολογία. Θα μπορούσε επίσης να ενισχύσει την παρακολούθηση ε, των, ε, της αξιοποίησης των ε, ευρωπαϊκών κονδυλίων που δίνονται. Αυτή η διαδικασία βεβαίως ήδη υπάρχει, αλλά θα πρέπει να ενισχυθεί. Επόμενη. Εδώ βλέπετε ποια είναι τα κενά που υπάρχουν στο συντονισμό και συνεργασία μεταξύ των εθνικών φορέων με, το, με τους ευρωπαϊκούς φορείς. Αυτά τα κενά μπορούν και πρέπει να ε, καλυφθούν. When we speak about uh, truth and reconciliation... Μιλήσαμε λοιπόν για τη διαδικασία αλήθεια και συμφιλίωση σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει έλλειψη κατανόηση για το τι έχει συμβεί στι κοινότητε των Ρωμά. Άρα, έχουμε πρώτον το δικαίωμα γνώση των θυμάτων και τη κοινωνία εν γέννη τι έχει γίνει στι χώρε του. Δεύτερον, πρόσβαση στη δικαιοσύνη στους πληθυσμούς των Ρωμά και παροχή ένδικων μέσων προσφυγής, αλλά και αποζημιώσεις είτε συμβολικές ή και ε, νομικές αποζημιώσεις. Αυτό μπορεί να ενισχύσει το αφήγημα του, της, της εφαρμογής του κράτου δικαίου. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Θα μπορούσε για παράδειγμα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δημιουργήσει, να συστήσει μια δική του εξεταστική επιτροπή ή θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα υψηλό επίπεδο διάλογο, ε, όπως έχει γίνει από την Κομισιόν σε άλλους τομείς και σε άλλα θέματα. Ακόμα το συζητάμε τι μορφή θα μπορούσε να πάρει μια τέτοια διαδικασία. Υπάρχουν πάντως πολλές εναλλακτικέ, όλες, όλες τους θετικές. Θα μπορούσε να ληφθεί υπόψη και η εμπειρία στη Σουηδία και στη Γερμανία. Αυτά είναι παραδείγματα τα οποία πραγματικά μπορούσαν να αξιοποιηθούν και από άλλα κράτη-μέλη. Γιατί φαίνεται ότι σε αυτέ τι δύο χώρε υπάρχει μια ε, ενισχυμένη ευαισθητοποίηση και έχουν ε, υπάρξει και απτά αποτελέσματα όσον αφορά τη μείωση της αποδοχής του αντιαθηκανισμού. Περνάμε τώρα στη συμμετοχή των Ρωμά. Έχουν με βάση το τελευταίο ενωσιακό πλαίσιο δημιουργηθεί κάποιες δομές για τη συμμετοχή των Ρωμά, ωστόσο η κοινωνία των πολιτών μπορεί να παίξει ενισχυμένο ρόλο όσον αφορά την καλύτερη εφαρμογή, παρακολούθηση, επισκόπηση του σχεδιασμού, της χρηματοδότησης και της εφαρμογής των τοπικών δράσεων. Βλέπουμε ότι οι αυτοοργανωμένες δομές των Ρωμά που είναι πολύ συχνά μικρής κλίμακας, κοινοτικέ πρωτοβουλίες, δεν έχουν τη δυνατότητα ε, πρόσβασης ε, στη χρηματοδότηση από τα ε, ενωσιακά κονδύλια. Πρέπει να βελτιωθεί αυτό, πρέπει να ενισχυθεί για να ενισχυθεί η δυνατότητα των, ε, των ίδιων των οργανώσεων των Ρωμά να χρηματοδοτούνται από στρατηγικές και καθεστώτα για την αντιμετώπιση της φτώχειας. Αυτά είναι, αυτές είναι κάποιες πρώτες σκέψεις, κάποια πρω, καταρκτικά πορίσματα στα οποία έχουμε καταλήξει. Η συνολική έκθεσή μας, όπως είπα, θα δημοσιευθεί τον Νοέμβριο. Στο τελικό γύρο θα απαντήσουμε σε διάφορες σχετικές ερωτήσεις. Ο Κλοντ Καν από το γραφείο του ΟΗΕ, που είναι η παρτιαμοστία του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, θα σας παρουσιάσει κάποια διδάγματα από την εφαρμογή του ενωσιακού πλαισίου για τους Ρωμά ούτω ώστε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα των Ρωμά και να σχεδιάσουμε πιο αποτελεσματικά μέτρα για την περίοδο μέχρι, μετά το 2020. Έχετε 10 λεπτά για να παρουσιάσετε τις σκέψεις σας. Σας ακούμε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τους συναδέλφους που εξακολουθούν να παραμένουν στην αίθουσα. Εμείς λέμε κάποια πράγματα από τη δική μας τη σκοπιά. Κάποια τα ακούσατε. Θα προσπαθήσω να προσθέσω και κάποια νέα πράγματα. Δεν θέλω να επαναλάβω ιδέε που ακούσατε, αλλά το βασικό είναι να προκύψει μια συνένεση από τη δική μας ομάδα και να προσθέσουμε και τη φωνή του ΟΗΕ τους φορεί που εκφράστηκαν. Σύντομα, για την ενδιάμεση έκθεση του ενωσιακού πλαισίου, ε, έχουμε την ίδια ερμηνεία με εσά. Και καταρχάς τα δεδομένα του Οργανισμού για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα ε, για την περίοδο 11 έως 16 και το πώς πάνε τα πράγματα ε, με βάση τις πρώτες πολιτικές της Ευρώπης για τους Ρωμά. Τα συμπεράσματά μας ε, τα συνόψε πολύ εύγλωτα ο εκπρόσωπος του οργανισμού αυτού του ΦΡΑ. Ορισμένες περιοχές είναι πιο καλές και είμαστε πιο αισιόδοξοι, ορισμένοι τομείς, δηλαδή, παραδείγματος χάρη, Έχουμε αυξήσει την εγγραφή στα σχολεία των ε, παιδιών ε, δημοτικού. Θετικό είναι αυτό. Υπάρχουν θετικές εξελίξεις και σε άλλους τομείς, αλλά υπάρχουν και αρνητικές εξελίξεις, οι οποίες είναι πολύ πιο έντονες σε ό,τι αφορά την απομόνωση. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε και να αναγνωρίσουμε ότι στα περισσότερα κράτη-μέλη υπάρχει απομόνωση των Ρωμά από του υπόλοιπου πληθυσμού για την περίοδο 2011 2016. Είναι ανησυχητικό κατά την άποψή μου δεν είναι κάτι που μας εκπλήσει, αντίθετα είναι αναμενόμενο και αντικατοπτρίζει μία αύξηση ε, της ε, πίεσης ε, των Ρωμά για να ενταχθούν στην κοινωνία, μεγαλύτερη ζήτηση για ένταξή τους στο εκπαιδευτικό σύστημα κτλ. Τις αντιστάσεις που αυτό δημιουργεί. Είπαμε πέρυσι τον Οκτώβριο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα σχόλιά μας και απαντήσεις μας, είναι σημαντικό να έχουμε και μια στρατηγική follow-up ε, συνέχειας μετά το 2020 και ελπίζουμε ότι θα υπάρξει. Υπάρχει μια θετική ορμή προς αυτήν την κατεύθυνση. Θέλουμε να πούμε όμως ε, βοερά ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για τη συνέχεια μετά το 2020 για την ένταξη των ΟΜΑ και θα πρέπει να τονίζει περισσότερο την ένταξη των Ρωμά και όχι την απομόνωσή του στην κοινωνία και την αντιμετώπιση της αθηνικανοφοβίας. Φυσικά και εμείς θεωρούμε ότι αυτά τα νούμερα σημαίνουν ότι θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στην ένταξη των Ρωμά στο πολιετές ε, δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο μετά το 2020. Διαβάζουμε τα ίδια έγγραφα, κυρίως τις προτάσεις Κομισιόν ε, από τον Ιούνιο. Κάποια πράγματα είναι θετικά. Σε ένα πιο δύσκολο περιβάλλον όμως, όπου γίνονται αιτήματα για περικοπές και απλουστεύσει από διάφορες φωνέ και τομείς, αυτά που έχουν μπει στην πρόταση της Κομισιόν δεν είναι τόσο λεπτομερή ή τόσο φιλόδοξα όσα με αυτά που υπάρχουν στην τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού. Το αντίθετο θα έπρεπε να συμβαίνει. Θα έπρεπε να δοθεί μεγαλύτερη ακόμα έμφαση στην αντιμετώπιση τη αντικανοφοβία και την αντιμετώπιση της του αποπονοτισμού εναντίον του. Μεγαλύτερη έμφαση στους κανονισμούς επίσης, ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να δώσουν δεδομένα για να δείξουν τι συμβαίνει ε, και το κατά πόσον εντάσσουν πραγματικά τους εντα, τους ε, απομονωμένους ας πούμε, στις κοινωνίες τους. Ε, τις επόμενες εβδομάδες και μήνες όλα αυτά τα θέματα θα ξανασυζητηθούν και μπορούν να μπουν στα σχέδια κανονισμών. Μιλάω για τα, τους κανονισμούς ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, αυτό είναι το πρώτο κομμάτι. Δεύτερον, και εμείς ζητούμε αλήθεια και συμφιλίωση. Συμφωνούμε με αυτούς που ζητάνε κάτι τέτοιο. Ε, συμφωνούμε με τα πορίσματα του Γενικού Συμβουλίου της Γερμανίας για τους Σύντι και τους ε, Ρωμά. Ε, όλο και περισσότεροι άνθρωποι λένε ότι αυτό είναι κανός ε, μηχανισμό, οι επιτροπέ δηλαδή και συμφιλίωσης για να αντιμετωπιστούν τα βαθιά ριζωμένα στερεότυπα, η παρανόηση, παρεξηγήσει, οι ασάφειες που υπάρχουν στην κοινωνία μα ε, για τα ιστορικά θέματα που, από τα οποία απορρέουν ε, οι τάσεις αποκλεισμού. Όλα αυτά που ακούσαμε από τη Σουηδία, την Νορβηγία και από άλλες χώρες που λένε ότι έχει νόημα να το κάνουμε αυτό για να αντιμετωπίσουμε ή τουλάχιστον να προσπαθούμε να, προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε την, τις παρεξηγήσεις, την κοινή γνώμη, τους, τις τρευλώσεις κτλ. Οι επιτροπές αλήθειας και Συμφιλίωση σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο είναι σημαντικέ. και οι επόμενοι 12 μήνε είναι σημαντικοί για το θα γίνει σε εθνικό επίπεδο. Όταν έχουμε προ τα τέλη του επόμενου έτου την ΕΕ Επιτροπή, θα επανέλθουμε εδώ για να σα πούμε, κοιτάξτε τι κάνουν τα κράτη-μέλη, έχουμε μια Ευρωπαϊκή Συνένωση, Α προσπαθήσουμε λοιπόν την επόμενη χρονιά να κάνουμε κάτι επιτέλου αυτό. Τέλο. Αυτά τα δύο που σας είπα τώρα τα έχουν ήδη καλύψει οι άλλοι συνάδελφοι. Επομένως θέλω να μιλήσω και για άλλα πράγματα σημαντικά και πιο λεπτομερή. Καταρχάς, κάναμε μια πολύ σημαντική παρουσίαση, ακούσαμε μια σημαντική παρουσίαση της, ε, του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Κομισιόν αυτή τη βδομάδα όπου παρουσιάστηκε το εξής, ότι 80% των ε, ατόμων ε, που αποκλείονται και απελάβνονται από την Ευρώπη προς τη Σερβία είναι Ρωμά. Ορισμένοι λένε ότι είναι τυχαίο αυτό. Ε, δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι πιστευτό κάτι τέτοιο. Επίσης, το να απελάσουμε, κάποιον και να τον διώξουμε προς μια άλλη χώρα είναι μια απίστευτα βίαιη πράξη και σε καμία περίπτωση δεν συντείνει στην κοινωνική ένταξη, δεν βοηθάει το άτομο αυτό και έχει βαθύτατες συνέπειες. Γιατί ξέρουμε διάφορες υποθέσεις. Δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι φτάσανε εχθέ αυτοί που απελάφνονται. Συχνά μιλάμε για ανθρώπους που γεννήθηκαν στη Γερμανία, Αυστρία, Ιταλία ή άλλες χώρες ε, και που αναγκάστηκαν να φύγουν για να πάνε στην Βοσνία, Σερβία, Κοσφοπέδιο, Αυτά είναι πολύ ευάλωτα άτομα και στέλνουμε και ένα απίστευτο μήνυμα σε αυτές τις ε, υποψήφιες χώρες. Γιατί τους λέμε πάρτε λίγα λεφτά, οι χώρες μας δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτά τα θέματα, παρότι ο αριθμός των ε, ανθρώπων αυτών είναι μικρός. Ασχοληθείτε εσείς. Εσείς ασχοληθείτε, εσείς αντιμετωπίστε το πρόβλημα. Και παρότι σε ένα επίπεδο οι υποψήφιες χώρες ε, ακούνε να τους λέμε αντιμετωπίσετε και εντάξτε τους Ρωμά, και τους δίνουμε και πακέτα χρηματοδότηση για να το κάνουν. Από την άλλη, στο άλλο επίπεδο τους λέμε εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε. Δεν μπορούμε να το κάνουμε και αφού δεν μπορούμε εμείς, γιατί να μπορείτε κι εσείς. Η ένταξη απαιτεί διακοπή αυτών των πολιτικών απέλασης, εκδίωξης χωρών από τη μία και απέλασή τους προς μια άλλη. Στη Σλοβακία έγινε μια ε, αστυνομική, ας πούμε, ένα μπλοκ της αστυνομίας ε, το 2013 με 60 αστυνομικούς οι οποίοι ε, προέβησαν σε φοβερές παραβιάσεις ε, ανθρωπινών δικαιωμάτων. Ξεκίνησε μια έρευνα στην αστυνομία, επειδή δύο χρόνια τελικά έκλεισε χωρίς καθόλου απαγγελία ε, κατηγοριών αντίον αστυνομικών. Και από τι αρχέ του περασμένου έτους οι μάρτυρε κατηγορήθηκαν για διάφορα αδικήματα ή διάφορα εγκλήματα. Για μας οι μάρτυρε, έτσι. Αυτό δείχνει ε, ρατσισμό, διακρίσεις, έλλειψη λογοδοσία αστυνομία, ανησυχίες για τα δικαιώματα του πολίτη για το ότι υπάρχει ατιμορρησία για αυτούς που παραβίασαν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ελπίζουμε ότι αυτή η έρευνα και η δίωξη, θα, ή μάλλον αυτή η δίωξη αυτών των ανθρώπων θα σταματήσει. Γιατί όταν δεν διώκουμε, ή μάλλον όταν διώκουμε ανθρώπους που έχουν την α, γενναιότητα να μιλήσουν αντίον αστυνομικών, τους τιμωρούμε τελικά η Σλοβακία θα πρέπει να αναγνωρίσει το ρόλο τους και θα πρέπει να αποζημιώσει τους Ρωμά άντρες και γυναίκες, θύματα στη Ρωσία και τα λοιπά, αλλά και άλλους ανθρώπους. Ε, αυτό το έχει πει ο ΙΕ από τις αρχές του 2000 ε, και από το 1977 στη Σλοβακία θεωρείται στόχος και θα πρέπει οι κυβερνήσεις της Σλοβακίας να κάνουν κάτι επιτέλους γι' αυτό. Σταματώ εδώ. Ευχαριστούμε πολύ. βλέπουμε κάτι που συμβαίνει συχνά ότι έχουμε ομιλητέ εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που μιλούν συγκεκριμένα για κράτη-μέλη, ενώ αυτοί που είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν λένε συγκεκριμένα σε ποιον αναφέρονται, οπότε εκτιμώ την ειλικρινιά σας. Επόμενη ομιλήτρια η κυρία Γελένα Γιωβάνοβιτς. λένε δε μου, ότι είναι η φωνή της κοινωνίας των πολιτών. Εντυπωσιακός ε, τίτλος. Αλλά όπως και να έχει είναι πολύ σημαντικό να ακούσουμε και την κοινωνία των πολιτών γιατί παίζεται πολύ σημαντικό ρόλο στην ενσωμάτωση των Ρωμά, εκπροσωπείται το δίκτυο έργο και θα παρουσιάσετε ορισμένες βέλτιστες πρακτικές από τη σκοπιά των ΜΚΟ με πανευρωπαϊκή εμπειρία. Και εσείς 10 λεπτά έχετε στη διάθεσή σας, παρακαλώ. Thank you very much. Uh, I would like to say at the very beginning that uh, I am sorry that the director of Ergo Network... Αρχικά, ε, να πω μεταλήψω ότι δεν είναι εδώ η Διευθύντρια, κυρία Γαμπριέλα Χαμάνοβα, που βρίσκεται αυτή στιγμή σε πολύ σημαντική αποστολή στην Ουκρανία ε, και κάνει ό,τι μπορεί για να δει Πώ μπορούμε να υποστηρίξουμε τους Ρωμά στην Ουκρανία που συχνά έρχονται αντιμέτωποι με φαινόμενα βία και ε, εγκλημάτων μίσου. Θα κάνω λοιπόν ό,τι μπορώ για να την βγάλω πρόσωπη. Και εκείνη και την οργάνωσή μου και την κοινωνία των πολιτών με την οποία συνεργαζόμαστε στενά. Να πω επίσης αυτής εξ αρχής ότι με μεγάλη προσοχή χρησιμοποιούμε τον όρο βέλτιστες πρακτικές. Με κάθε ειλικρίνη, λοιπόν, μπορώ να σας πω ότι δεν πιστεύουμε ότι εμείς είμαστε οι βέλτιστοι, οι καλύτεροι, αλλά θα σας παρουσιάσω τρεις πρωτοβουλίες που θεωρούμε ότι είναι τουλάχιστον πολλά υποσχόμενες. Ακόμα παρότι βλέπουμε κάποια πρώτα άμεσα αποτελέσματα, δεν γνωρίζουμε ποιος θα είναι ο μακροπρόθεσμος αντίκτυπος και αν θα πετύχουμε τον τελικό μας στόχο. Το δίκτυο έργο με προσήλωση εργάζεται κατά ε, του αντιαθηγανισμού εδώ και πολλά χρόνια. Και σε αυτή την παρουσίαση θα ήθελα να σας μιλήσω για τις ε, ανάγκες και τα κενά που εντοπίζει η κοινωνία των πολιτών και οι φορείς της σε ό,τι αφορά τη θεσμική ανταπόκριση ως προς την ε, καταπολέμηση του αντιαθηγανισμού σε εθνικό επίπεδο. Εδώ καλό είναι να πούμε ότι συνεργαζόμαστε με την κοινότητα των πολιτών σε όλα τα κρατημέλη. Αλλά και στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Θα σα παρουσιάσω λοιπόν αυτά τα βασικά κενά και στη συνέχεια ε, θα αναφερθώ και σε ορισμένες βασικές ε, προκλήσεις Πριν περάσω ε, στη συνέχεια της παρουσίασης, θα ήθελα να σας πω αρχικά από πού προέρχονται όλες αυτές οι πληροφορίες. Και θα σας αναφέρω και τα ονόματα των πρωτοβουλειών. Ένα είναι ένα πρόγραμμα που λέγεται Κοινή Πρωτοβουλία για την Ενδυνάμωση της Κοινωνίας των Πολιτών Ρωμά στις, ε, στα Δυτικά Βαλκάνια και στην Τουρκία, ε, που διακονώνεται από την DG και άλλους φορείς. Εδώ συνεργαζόμαστε με φορεί τη κοινωνία των πολιτών από έξι χώρε των Δυτικών βρακανίων και από την Τουρκία. Η επόμενη σημαντική πρωτοβουλία είναι το Roma Civil Monitoring. Μπορείτε να βρείτε στοιχεία στο διαδίκτυο. Ξεκίνησε με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πιλωτικό πρόγραμμα. Ε, το διαχειρίζεται η DG Justice. Μέσω αυτού του προγράμματος ε, ανταλλάσσουμε πληροφορίες με περίπου 90 φορείς της κοινωνίας των πολιτών και εμπειρογνώμονες από 27 κράτη-μέλη. Το κοινό στοιχείο σε αυτές τις δύο πρωτοβουλίες είναι μια ενέργεια που αναλαμβάνει η κοινωνία των πολιτών, πιο συγκεκριμένα η αναφορά περιστατικών αντιαθηγανισμού και καταπολέμηση του φαινομένου αυτού αυτή η ενέργεια υπάρχει και, στις, και στα δύο προγράμματα. Τρίτο πρόγραμμα που ήθελα να αναφερθώ είναι άτυπο, αλλά σημαντικό για μας, γιατί θεωρούμε ότι πρέπει να δημιουργήσουμε συνασπισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι η συμμαχία κατά του αντιαθηγανισμού. Βασικά μέλη είναι το δίκτυο Έργο, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά του Ρατσισμού και το Γερμανικό Δίκτυο Σύντη και Ρωμά. Η συμμαχία αυτή δημοσιοποίησε ένα έγγραφο αναφοράς για τον αντιαθηγανισμό, γιατί τα μέλη είδαν ότι είναι δύσκολο να δημιουργήσουμε και να καταλήξουμε σε έναν ορισμό του φαινομένου για να το κατανοήσουμε καλύτερα. Και θέλουν και να αυξήσουν ευαισθητοποίηση για όλες τις διαστάσεις του φαινομένου. Αυτό είναι σημαντικό γιατί είχαμε τη στήριξη εκατοντάδων φορέων από την κοινωνία των πολιτών που κατανοούν ότι έχει έρθει η ώρα να εμπλουτίσουμε ε, τη θέση των εμπλεκομένων ε, φορέων που έχουν να κάνουν ε, με ε, τις αντιλήψεις που κυριαρχούν για τους Ρωμά, τους και άλλες τέτοιες ομάδες. Πρώτα απ' όλα, πολλοί φορείς κοινωνίας των πολιτών και κάποιοι θεσμικοί φορείς αναγνωρίζουν την, ε, την μακραίωνη ε, διάκριση την οποία εφίστανται οι Ρωμά, αλλά πολλοί άλλοι δεν το αναγνωρίζουν. Μετά έχουν εντοπιστεί σημαντικά ανά, όχι σε ό,τι αφορά την αναγνώριση και κατανόηση του φαινομένου, αλλά και από πλευρά έλλειψη θεσμικών δομών και επιδόσεων για την καταπολέμηση του φαινομένου. Είναι αλληλένδετα βέβαια αυτά τα δύο, γιατί αν οι φορεί δεν κατανοούν τι είναι αυτό το φαινόμενο και δεν μπορούν να το αναγνωρίσουν, φυσικά και δεν μπορούν να το καταπολεμήσουν. η έλλειψη ρητής αναγνώρισης του αντιαθηγανισμού δεν επιτρέπει την ανάπτυξη ειδικών δικτών ε, ή την χορήγηση χρηματοδότησης για την καταβολή του φαινομένου. Επίσης, η έλλειψη αναγνώρισης, ρητής αναγνώρισης του φαινομένου οδηγεί σε έλλειψη ικανότητας παρακολούθησης των ενεργειών αντιαθυγενισμού και δεν μας επιτρέπει να αξιολογήσουμε και τον αντίκτυπο των ε, δημοσίων πολιτικών. Τέλος, είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε τις ε, διάφορες διαστάσεις ε, του φαινομένου. Μεγάλη πρόκληση εδώ είναι ο θεσμικός αντιαθηγανισμός. Για παράδειγμα, η αστυνομία ορισμένες φορές επιτρέπει τον αντιθυγανισμό γιατί δεν ανταποκρίνεται σε φαινόμενα βίας κατά τον Ρωμά ή κάποιες φορές ε, διαπράττουν και οι ίδιοι ε, εγκλήματα κατά τον Ρωμά. Είδαμε ότι ο αντιθυγανισμός υπάρχει σε πολλούς τομείς ε, της κοινωνικής ζωής, από το πολιτικό βίο, την εκπαίδευση, την υγεία, μέχρι τα ΜΜΕ. 70 χρόνια και έχουν περάσει από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν εγκλήματα μίσου κατά τον Ρωμά και εναντίον άλλων ε, ε, ομάδων που ε, για κάποιο λόγο εκλαμβάνονται ως Ρωμά και δεν καταγράφονται πολλά τέτοια περιστατικά. Ο ρατσιστικός χαρακτήρας παραγνωρίζεται και τα εγκλήματα κατά των Ρωμάτων, Σύντη και λοιπόν τέτοιων ομάδων δεν ε, αναδεικνύονται γενικά από την κοινωνία. Καταλήξαμε και σε μία σειρά συστάσεων που θα θέλουμε να σας παρουσιάσουμε σήμερα. Κάποια προκύπτουν από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και κάποια από εθνικού φορεί. Είναι σε όλα σημαντικά να τα εντάξουμε ε, στο νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο, το οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνει και συγκεκριμένα μέτρα για την ε, ανταπόκριση ε, και καταπολέμηση του αντιαθηγανισμού με όλες τις προεκτάσεις και να αποτελέσει και μια εγκάρση προτεραιότητα και ως δίκτυο έργων και ευρύτερα στηρίζουμε την πρωτοβουλία της κυρίας Post ε, για τη θέσπιση αυτής της σύσταση αλήθειας και ε, συμφιλίωσης ε, σε όλα τα κρατημέλη. Και τέλος πιστεύουμε ότι το έργο σε ευρωπαϊκό επίπεδο κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, όμως δεν έχει κανένα νόημα εάν οι εθνικές αρχές δεν αναλάβουν τη δέσμευση να καταπολεμήσουν τον αντιαθηγανισμό. Τα κράτη-μέλη λοιπόν και, και άλλες χώρες θα πρέπει να αναγνωρίσουν τον αντιαθηγανισμό ως ε, μορφή ρατσισμού. Και πώς θα γίνει αυτό. Πρέπει να ιεραρχήσουν ως προτεραιότητα την καταπολέμηση του αντιαθηγανισμού στο πλαίσιο των ε, δικών τους ε, στρατηγικών εγγράφων και νομικά. Δεύτερον, θα πρέπει να ενσωματώσουν αυτό το στοιχείο σε όλες τις πολιτικές, όπως για παράδειγμα τα εθνικά σχέδια δράσης κατά του ρατσισμού. Τρίτον, η χρηματοδότηση είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση των πολιτικών. Φαντάζομαι ότι αυτό είναι κατανοητό για όλους, ούτως ώστε ο αντιθυγανισμός να μην ε, μείνει κενό γράμμα. Τέταρτον, οι θεσμικοί φορείς, οι αρμόδιες αρχές, θα πρέπει να αρχίσουν ε, να παρακολουθούν και να καταγράφουν και να ανταποκρίνονται σε ε, ενέργειες αντιθυγανισμού, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει τώρα. Και τέλος, οι θεσμοί θα πρέπει να αναλάβουν δράση για να προστατεύσουν τα δικαιώματα ε, όσων ε, ε, βιώνουν τον αντιεθνικανισμό σε καθημερινή βάση και οι κρατικοί φορείς και θεσμοί θα πρέπει να διασφαλίσουν την πρόσβαση αυτών των ανθρώπων στη δικαιοσύνη. Τέλος, ελπίζουμε ότι θα αυξηθεί κατά αυτόν τον τρόπο η πολιτική βούληση σε όλες τις χώρες για την καταπολέμηση του φαινομένου και προκειμένου να οικοδομήσουμε μία ε, κοινωνία χωρίς ρατσισμό. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. That, uh, the European Parliament also... Έχουμε απευθυνθεί και στη ΣΕΠΟΛ, τον Οργανισμό για την Εκπαίδευση των Αστυνομικών Αρχών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, ώστε να παρέχει εκπαίδευση και γύρω από αυτό που αποκαλέσατε εσείς σε ε, θεσμικό αντιαθηγανισμό. Λοιπόν, έχουμε τώρα δύο βουλευτές Εθνικών Κοινοβουλίων, την, ε, τον κύριο Καταλήν Δημήτριο Τόμα που είναι γερουσιαστής από την ε, Ρουμανία και έχουμε μαζί μας και τον κύριο Βέλσκο Καστάζη που είναι μέλος της Κροατικής Βουλής. Ξεκινάμε με τον κύριο Τόμα, μετά θα έχει το λόγο ο κύριος Καστάζη. Έχετε αμφότεροι περίπου 8 λεπτά στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ πολύ, μεγάλη μου τιμή που βρίσκομαι εδώ. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, όπως είπα είναι μεγάλη μου τιμή που έχω την ευκαιρία να συμμετέχω σε μια τόσο ενδιαφέρουσα συζήτηση για ένα θέμα που έχει τόσες πολλές φορές συζητηθεί. Υπάρχει εμπειρία σε όλα τα κράτη-μέλη από τη συνύπαρξη με τις κοινότητες των Ρωμά. Η στρατηγική της ρουμανικής κυβέρνησης όχι μόνο δεν απέφερε ε, θετικά αποτελέσματα, αλλά έχει ενισχύσει και τις ε, διακρίσεις και, την, και το άνοιγμα της ε, ψαλίδας, καθώς και την ενίσχυση των προκα, προκαταλήψεων. Αποτέλεσμα, μαζικό κύμα μετανάστασης των Ρωμά προς δυτικές χώρες της, Ευ της Ευρώπης. Ο αντιαθηκανισμός πλέον αναφέρεται ως επίσημη επίσημος όρος για, σε έγγραφα που αφορούν την καταπολέμηση του ρατσισμού και των διακρίσεων. on all of the EC. Υπάρχει πλέον ε, ως ε, όρος ε, που αναφέρεται σε επίσημα έγγραφα και πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ανάγκη μιας ε, νέας ισορροπημένης και επανασυμφιλωτικής προσέγγισης για όλα τα ζητήματα που αφορούν την, την ε, κοινωνική ένταξη μέσω ολοκληρωμένων μέτρων αναδεικνύεται ως βασικό συμπέρασμα της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου μας. Οι νομικές τροποποιήσεις προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι σύγχρονε συνθήκε αποτελούν σημαντικό στοιχείο τη μελλοντική μα προσέγγιση. Η ανάγκη λοιπόν μια προσαρμοσμένη και συντονισμένη προσέγγιση για τον αντιαθυγιανισμό πρέπει να ε, συμπεριλάβουν στι δικέ μας, ε, στις δικές μας περιστάσεις και άλλα δύο στερεότυπα. Η συμμετοχή των Ρωμά στην διαδικασία λήψη αποφάσεων για τις πολιτικές που έχουν ως ε, στόχο τους ίδιους πρέπει να ε, αντιμετωπιστεί μέσω της υποστήριξης ε, της συλλογικής ευθύνης και της αρχής της αλληλεγγύης. Η ηγεσία από το ίδιο τους Ρωμά ως φάρος ακαιρεότητας, ικανότητας και ανταγωνιστικότητας είναι απαραίτητο στοιχείο προκειμένου να προωθήσει η κοινότητα τον εαυτό της και για να αναπτύξει τις δυνατότητές της. Η, η, η ιδιαιτερότητα ορισμένων ευρωπαϊκών χωρών, όπως είναι η ισορροπία εξωτερικής και εσωτερικής μετανάστευσης, η, ε, βελτιωμένη αποτελεσματικότητα ε, όσον αφορά συγκεκριμένες ε, κοινωνικές ομάδες στις οποίες έχουν παρουσία η Ρωμά, όπως είναι η πλανοδή μουσική, η Ζητιάνη αποτελεί ένα στοιχείο που πρέπει να αντικατοπτρίζεται στις ε, δημόσιες πολιτικές για τους Ρωμά. Αυτό απαιτεί συγκεκριμένους κανόνες που θα ισχύουν τόσο για τις κοινωνίες των Ρωμά όσο και για τα θεσμικά όργανα. Η έναρξη λοιπόν μιας δημόσιας αντιρατσιστικής εκστρατείας για την προστασία των ε, γυναικών και των παιδιών των Ρωμά πρέπει να είναι μία από τις εκφράσεις εθνικής και ευρωπαϊκής πολιτικής για την διαρθρωμένη αντιμετώπιση του αντιαθηγανισμού και των διακρίσεων. Η Ρουμανία είναι υπέρ ε, της ανάπτυξης δημόσιων πολιτικών που θα καταλήγουν στην καταπολέμηση του αθιαδικανισμού και θα συμβάλλουν σε μια προοδευτική τυποποίηση των πολιτικών στα κράτη-μέλη και στους, στις τοπικές κοινωνίες των Ρωμά. Η ένταξη στο Ρωμά δεν είναι ένα εθνικό πρόβλημα, αλλά πανευρωπαϊκό. Και γι' αυτό χρειάζεται ευρωπαϊκή λύση. Θέλω να επισημάνω ότι η υπεράσπιση τη ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ο αγώνα κατά των διακρίσεων και κατά του αντιαθηγανισμού είναι ρουμανικέ προτεραιότητε. Γι' αυτό με μεγάλη μου χαρά μπορώ να σα προσκαλέσω να συμμετάσχετε στη συζήτηση που γίνεται στη χώρα μου ε, και που θα γίνει στο πλαίσιο της επικείμενης Ρουμανικής Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριο Καστάζη. Πρόβλημα τεχνικό gleda i kako je pripremljen. Πρόεδρε, πρέπει να, θα ήθελα να σας μιλήσω λιγάκι για το, την εμπειρία ενός ε, παιδιού που πάει στο σχολείο για πρώτη φορά στο δημοτικό ε, και είναι Ρωμά. Καταρχάς θέλω να σας ευχαριστήσω όλους και που συμμετέχετε σε αυτή τη συζήτηση για την ένταξη των Ρωμά. Είμαι Κροάτης. Ε, για τρίτη φορά έχω εκλεγεί στο Κροατικό Κοινοβούλιο και εκπροσωπώ όλες τις ε, μειονότητες που υπάρχουν στην ε, Κροατία και είναι πολλές. Τούρκοι, ε, Βούλγαροι, Ουγγροί κτλ. κτλ. Δεν είχα πολλές ευκαιρίες να έρθω εδώ στο Κοινοβούλιο. Ε, και δεν έχω πολλές πληροφορίες για την κατάσταση άλλων μειονοτήτων. Δεν ξέρω πολύ καλά πώς ζουν οι Ρωμά. Ε, το, δουλεύω σε τοπικό επίπεδο και συνεργάζομαι με διάφορες οργανώσεις που εκπροσωπούν τους Ρωμά, ε, συμβούλια των Ρωμά και τόπους, πόλους έλξης των Ρωμά στην χώρα μου, στην Κροατία. Το θέμα μου είναι οι εθνικές στρατηγικές για την ένταξη των Ρωμά. Και πρέπει να σας πω ότι είμαι δυσαρεστημένος με την κατάσταση εφαρμογής τους. Παρότι τα έγγραφα είναι φανταστικά, γιατί εντοπίζουν τα προβλήματα που ζουν οι Ρωμά, αυτό που δεν έχουμε είναι σωστή εφαρμογή και θεσμική λογοδοσία. Μπορούμε να υιοθετούμε υπέροχα έγγραφα πλαίσιο και στρατηγικές. Αυτό είναι εύκολο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε όμως το πώς λειτουργούν τα Υπουργεία και πώς λειτουργούν ε, τα δημοτικά και κοινοτικά συμβούλια. Το κάνουν με βάση την εθνική νομοθεσία και την εθνική ενωμένη τάξη. Αυτό που προσπαθώ να κάνω σε αυτή τη θητεία είναι να μεταφέρω τα στρατηγικά έγγραφα στο εθνικό, στην Εθνική Ενωμή Τάξη και στην, στο νομοθετικό μας πλαίσιο. Η τρέχουσα κυβέρνηση, η σημερινή κυβέρνηση στην Κροατία, έχει μια εθνική στρατηγική και έχει και επιχειρησιακά προγράμματα. Πολύ ωραίος τρόπος αυτός είναι για να προχωρήσουμε. Και είναι και κάτι το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρότυπο ε, όμως η φάση της ε, εφαρμογής, η διαδικασία της εφαρμογής δεν είναι εξίσου ικανοποιητική ή αρκετά γρήγορη. Για την εφαρμογή θα ήθελα να σας πω ότι στην Κροατία δεν είχαμε βασικά δεδομένα για τους Ρωμά, βασικά δεδομένα, βασικά στατιστικά στοιχεία για τους Ρωμά, για, τις, για τους τέσσερις τομείς προτεραιότητας που αφορούν την εκπαίδευση, την απασχόληση, την υγεία και τη σταγή. Ξοδέψαμε χρόνια ατελείωτα να εκπονούμε μέτρα χωρίς να έχουμε βασικά στοιχεία για τους Ρωμά. Νομίζω ότι το ίδιο συμβαίνει σε όλα τα κράτη-μέλη. Πολύ συχνά ο κόσμος έχει τα μάτια του στραμμένα στα ευρωπαϊκά project που κάνουν ε, μη κυβερνητικέ οργανώσεις και που δεν συμπεριλαμβάνουν αρκετά τους Ρωμά. Συχνά ε, με τη συνεργασία των τοπικών αρχών. Αλλά δεν είμαστε ικανοποιημένοι ούτε με αυτό. Θα ήθελα να σας τονίσω λοιπόν ότι τα ευρωπαϊκά project αναγνωρίζουν το πρόβλημα που ζουν οι Ρωμά. Αλλά οι συνθήκες υποβολής των υποψηφιωτήτων, οι διαγωνισμοί δηλαδή και τα λοιπά, δεν λαμβάνουν υπόψη τις φοβερές δυσκολίες μέσα στις οποίες ζουν οι Ρωμά. Εγώ νομίζω ότι κάποια από τα ευρωπαϊκά project θα πρέπει να εστιάζουν απόλυτα στα πραγματικά προβλήματα της κοινότητας στο Ρώμα και θα πρέπει ε, αυτά τα project να έχουν ειδικό καθεστώς και ειδικό μηχανισμό παρακολούθησης σε σχέση με τα υπόλοιπα project της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, νομίζω ότι αυτά τα ευρωπαϊκά ε, project είναι ήπια, soft ας πούμε, που αντιμετωπίζουν την άτυπη και μη τυπική εκπαίδευση και κατάρτιση. Ε, και πολύ σπάνια αφορούν την ένταξη των Ρωμά στην αγορά τελικά. Η κοινότητα των Ρωμά στην Κροατία θα ήθελε να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στην ένταξη των Ρωμά σε, προγράμματα και έργα υποδομών, σε προγράμματα άμεσης βοήθειας που θα δίδεται σε άτομα, συγκεκριμένα άτομα, νέους ειδικά, για να έχουν καλύτερη ευκαιρία ένταξη στη ζωή τους μετά. Λαμβάνοντα υπόψη την κατάσταση λοιπόν στην οποία ζουν οι Ρωμά, λαμβάνοντα υπόψη τι πολύ δύσκολε συνθήκε διαβίωσή του και το βιωτικό του επίπεδο, θα ήθελα να σα πω ότι οι προσπάθειε ένταξή του μέχρι στιγμή ήταν α, αποτυχημένες. Το βασικό πρόβλημα είναι η έλλειψη λογοδοσίας και ανάληψη ευθυνών των κρατών μελών σε ό,τι αφορά την εφαρμογή συγκεκριμένων πολιτικών οι οποίες θα μπορούσαν να λύσουν το πρόβλημα. Από τις δηλώσει και τα έγγραφα πώς θα περάσουμε στις πράξεις. Δεν αρκούν τα στρατηγικά πλαίσια αν δεν υπάρχει καμία υποχρέωση να λογοδοτήσει κανείς για το επίπεδο εφαρμογής, για την κατάσταση εφαρμογής αυτών των εγγράφων. Εάν δεν εστιάσουμε επίση στις συνθήκες διαβίωσης των Ρωμά, και, όχι, και να μην μιλάμε μόνο για βραχυπρόθεσμα, ήπια προγράμματα και project. Εγώ ξέρω ότι οι δικοί μας οι Ρωμά στην ζουν σε ιδιαίτερες συνθήκες. Σε συγκεκριμένες ε, τοποθεσίες, σε συγκεκριμένους χώρους, μακριά από τις βασικές υποδομές, βασικές πόλεις, κοινότητες, ε, σε απομονωμένοι, όχι σε επαφή με τον γενικό πληθυσμό. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να εφαρμόσουμε πολιτικές ένταξης. Όχι όμως ε, για να του κοινωνικοποιήσουμε και όχι μόνο στον τομέα τη εκπαίδευση. αλλά επίσης να υπάρξει φυσική επαφή, φυσική ένταξη των Ρωμά στην ε, πραγματική κοινωνία, στην κοινωνία, την κανονική. Να χρησιμοποιήσουμε την εκπαίδευση ως μέσο για να προσφέρουμε εκπαίδευση στους Ρωμά, εκπαίδευση που θα τους χρησιμεύσει μετά στην αγορά εργασίας. Επίσης, θα ήθελα να σας πω ότι οι Ρωμά στην Κροατία δεν είναι ικανοποιημένοι με την εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής για την ένταξή τους, που τους αφορά, και είμαστε πολύ δυσαρεστημένοι με το γεγονός ότι δεν υπάρχει πολιτική λογοδοσία για την έλλειψη εφαρμογή. Επίσης πιστεύουμε ότι τα ευρωπαϊκά έργα και προγράμματα που χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι αρκετά ευέλικτα και δεν εστιάζουν σε θέματα προτεραιότητας. Τέλος, θα πρέπει να προσφέρουμε συγκεκριμένες λύσεις σε αναγνωρισμένα προβλήματα, με προθεσμίες, χρονοδιαγράμματα, με πολιτική και οικονομική λογοδοσία. Αλλιώς δεν υπάρχει καμία ανάγκη να έχουμε στρατηγικά πλαίσια. Ευχαριστώ. Φανταστικά μας τα είπατε. Και από πλευρά χρόνου. Τον σεβαστήκατε, ήσασταν στο τσακ. Ανοίγω τώρα το λόγο για τους βουλευτές. Έχουμε πέντε, πέντε ομιλητές από εθνικά κοινοβούλια και έχω και ευρωβουλευτές, τον κύριο Ένστα και τον κύριο Φρανς και άλλον έναν ευρωβουλευτή. Γιάννα Παστούτσοβα από την Τσεχική Δημοκρατία, δύο λεπτά παρακαλώ. Στο πρώτο πάνελ ήμουν πολύ χαλαρή. Και τώρα μας πιέζει ο χρόνος. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Με μικρόφωνο κατά προτίμηση. Δεν θα επαναλάβω πράγματα που ακούσαμε. Σας ευχαριστώ που μας προσκαλέσατε. Ε, είμαι από τη Τσεχική Δημοκρατία και είμαι πρόεδρος της Επιτροπής εθνικών μειονοτήτων, οικογένειας και ισότητα φύλων. Η τσεχική δημοκρατία περιγράφηκε με αρνητικές αποχρώσεις και όρους ε, και από τους πρώτους πανελίστες και από τους δεύτερους. Έχουμε κάνει όμως πολλά πράγματα στην τελευταία μας ε, κοινοβουλευτική θητεία ε, για το, την κουλτούρα και τον πολιτισμό και, τον, και την εκπαίδευση. στο πρώτο πάνελ δεν μπόρεσα να μιλήσω, Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα τώρα να σας μιλήσω για το εξής πράγμα. Δεν ξέρω για το, την κατάσταση στα άλλα κράτη-μέλη, αλλά τα μέσα ενημέρωσης δεν μιλάνε ε, και δεν δίνουν τα καλά παραδείγματα επιτυχημένης προσπάθειας υπέρ των Ρωμά. Ε, νομίζω ότι τις καλές πρακτικές θα πρέπει να τις διαδίδουμε στον τομέα της απασχόλησης, στις κοινωνικές επιχειρήσεις, ε, επιτυχημένες επιχειρήσεις, ας πούμε, που προσλαμβάνουν Ρωμά, γιατί τουλάχιστον στην τσεχική δημοκρατία τα ΜΜΕ μόνο ε, μιλάνε για τις αρνητικές εμπειρίες, δεν μιλάνε για τις θετικές εμπειρίες. Δεν ξέρω ποια είναι η κατάσταση στα άλλα κράτη-μέλη, αλλά κάνω έκκληση εδώ να γίνεται μια πιο σωστή πληροφόρηση από τα ΜΜΕ. Γιατί πραγματικά τα ΜΜΕ επηρεάζουν τα μυαλά, επηρεάζουν την οροπία του κόσμου. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λάσλο Ήμρα από την Ουγγαρία. Παρακαλώ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ακούσαμε κάτι πολύ ε, ανησυχητικό, θα έλεγα, στην πρώτη ομιλία. Αναφέρομαι στο γεγονός ότι το προσδόκιμο ζωής των Ρωμά είναι 12 χρόνια μικρότερο από 17 χρόνια ε, από το γενικό πληθυσμό. Επιβεβαιώνω αυτήν την πληροφορία και είναι πραγματικά Πάρα πολύ ανησυχητικό το γεγονός αυτό. Διότι αυτό συνδέεται και με την υγειονομική και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη που παρέχεται στους ανθρώπους αυτούς. Όταν δεν υπάρχει οικογενειακός γιατρός, είναι προφανές ότι δεν μπορεί να δοθεί η απαραίτητη ε, ιατρική και φαρμακευτική περίθαλψη. Είναι ένα θέμα που μας απασχολεί πάρα πολύ και στην Ουγγαρία. Και αυτό είναι εξαιρετικά ανησυχητικό, γιατί πρέπει κανεί να συμπολογίσει το γεγονό ότι έτσι και αλλιώ το προσδόκιμο ζωή στην Ουγγαρία είναι τέσσερα χρόνια λίγο μικρότερο από ότι ο, μεσ, ο ευρωπαϊκό μέσο όρο. Οπότε μιλάμε για 12 συν, 10, συν 4 χρόνια. Όλα αυτά συνδέονται με την κατάσταση στην, στην κοινωνία, στην αγορά εργασίας, με περιβαλλοντικά θέματα. Νομίζω ότι αυτό, αυτό είναι ένα πραγματικό θέμα που μας απασχολεί όχι μόνο σήμερα, θα, θα συνεχίσει να μας απασχολεί και στο μέλλον. Όσον αφορά την υγειονομική και ιατροφαρμική ε, περίθαλψη που παρέχεται στους Ρωμά, είναι ένα θέμα που θα πρέπει να αποτελέσει, και, να αποτελέσει βασικό θέμα των στρατηγικών που θα αναπτυχθούν σε εθνικό επίπεδο. Θα πρέπει με κάθε ευκαιρία να εξασφαλίζεται η ιατροφαρμακευτική, υγειονομική περίθελψη των ανθρώπων. Πρέπει να πιστούν τα μέλη των κοινοτήτων των Ρωμά ότι η υγεία τους και η προσωπική τους υγιεινή είναι σημαντικότατα θέματα στα οποία θα πρέπει να δοθεί απαραίτητη ε, προσοχή. Σεσίλ Κιέγγι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να θέσω ένα θέμα πολύ συγκεκριμένο για τα στρατόπεδα των Ρωμά. Ε, υπάρχει και σχετικό κοινοβουλευτικό ερώτημα για μια ε, ε, για ένα πρόβλημα ενός καταβλισμού Σίντι στον Καλαράντε ε, το οποίο επισκέφτηκα πριν από λίγο καιρό. Ζουν επί πάρα πολλές γενιές ανθρώπων Ιταλικής Ιθαγένειας με τρόπο έφτακτο και ειρηνικό. Μπορεί να ξε, ξεχαρβαλωθεί αυτός ο καταβλισμός ε, που είναι μακραίωνος. Υπάρχουν εθνικές στρατηγικές για την ένταξη των Ρωμά. Ε, η Κομισιόν στα πλαίσια αυτών ε, λέει ότι δεν θα πρέπει να έχουμε τέτοιες... Ε, δεν θα πρέπει να υπάρχει διάλυση καταβλισμών και αναγκαστική μετακίνηση ε, πληθυσμών. Υπάρχουν ε, κρατικοί και επίσημοι φορεί που δεν είναι υπέρ τη ένταξη. Παραδείγματο χάρη, ο Δήμαρχο του Γκαλαράτε στην Ιταλία. Δεν πρέπει να διαλύσει τον ε, καταβλισμό αυτό, ε, γιατί μιλάμε για οικογένειες Ιταλών, αλλά κυρίως μιλάμε για το μέλλον ευάλωτων ανθρώπων, οι οποίοι ετοιμάζονται να περάσουν το χειμώνα τώρα. Και πού θα τον περάσουν. Ερώτηση προ την Κομισιόν. Πώς θα εξασφαλίσετε ότι οι διαδικασίες αυτές διάλυση του καταβλισμού γίνονται με σεβασμό των δικαιωμάτων όλων και κυρίως των πιο ευάλωτων ανθρώπων. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω και την Σοράγια Πόστ για τη δουλειά που κάνει εδώ και όλους τους συναδέλφους που ασχολήθηκαν με αυτό το θέμα σε αυτή την κοινοβουλευτική θητεία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, Σεσίλη. Δυστυχώ δεν είναι εδώ εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οπότε αν θέλει να απευθύνει κάποιο ερώτημα προ εκείνου να το κάνει γραπτό, πολύ φοβάμαι. Θα δώσουμε το λόγο και πάλι στην κυρία Θελαρίτη από την Ελλάδα. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να τονίσω ότι η κοινωνική ένταξη ε, είναι απαραίτητη για να αμβλύνουμε αυτό που λέμε αντιαθηγανισμό. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά. Σημαίνει ότι πρέπει να ξεκινήσουμε να αντιμετωπίσουμε τις αρνητικές συνθήκες διαβίωσης στο Ρωμά μέσα από μια χαρτογράφηση και μια τυπολογική ανάλυση των οικισμών μπορούμε να αναπτύξουμε στεγαστικές πολιτικές, ε, τέτοιες που να είναι φιλικές ως προς την αντιμετώπιση του προβλήματος, γιατί διαφορετικά δεν μπορούμε να προχωρήσουμε την πρόσβαση στην εκπαίδευση, στην υγεία κτλ. Όσον αφορά την εκπαίδευση, εγώ θα μπορούσα να πω ότι Υπάρχουν, για παράδειγμα, προγράμματα που στηρίζουν ε, τα παιδιά το Ρωμά ως προς τα προβλήματα της γλώσσας. Εμείς έχουμε υποδοχή, τάξη υποδοχής για να μπορούν να στηριχτούν ε, ως προς τη γλώσσα τα παιδιά το Ρωμά. Έχουμε επίσης προγράμματα που αφορά την προσέγγιση των οικογενειών το Ρωμά για να μπορούν να διευκολύνονται στις υπηρεσίες ε, υγειονομικής, ό,τι αφορά δηλαδή για να πηγαίνει το παιδί στο σχολείο. Όμως δεν υπάρχουν προγράμματα ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών για να ε, γίνει όλο αυτό αποδεκτό μέσα σε μια τοπική κοινωνία. Εδώ νομίζω ότι οι επιτροπές συμφιλίωσης θα, θα μπορούσαν να παίξουν ένα πολύ σοβαρό ρόλο ακριβώς για να αμβλύνουν αυτή την αντίθεση που υπάρχει μεταξύ των δύο κοινοτήτων. Το δεύτερο που θα ήθελα να επισημάνω είναι το κομμάτι, στο κομμάτι της απασχόλησης. Στο κομμάτι της απασχόλησης, για παράδειγμα, ε, με μία θεσμοθέτηση ε, ενός ε, άδειας, δηλαδή άσκηση υπαίθριου εμπορίου, ε, είχαμε καλύτερα αποτελέσματα, ώστε επειδή αυτό γινόταν παράνομα από τη μεριά των Ρωμά, έτσι να αντιμετωπίσουμε, ώστε να μην αντιμετωπίζουμε προβλήματα με την αστυνομία. Νομίζω ότι βοηθώντας αυτούς τους ανθρώπους να, να, να ασκήσουν αυτό το επάγγελμα ή για παράδειγμα είναι, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον η δυνατότητα που έχουν να συνδιοργανώνουν ειδικέ υπαίθριες αγορές με δήμους, δηλαδή σωματεία και σύλλογοι Ρωμά με δήμους. Και αυτό πραγματικά δίνει μια άλλη διάσταση στο να βληθεί αυτός ο αντιαθηγανισμός που υπάρχει. Ολοκληρώνοντας θα ήθελα να εντοπίσω ότι ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέμε εμείς η θεσμική η πρόσβαση των Ρωμά σε υπηρεσίες που αντιμετωπίζουν ένα έντονο πρόβλημα και εκεί πραγματικά ο ρόλος του διαμεσολαβητή και τελειώνω έχει να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο και έχει να παίξει αν πιστοποιηθεί και σε μας γίνεται αυτή η προσπάθεια και νομίζω ότι και στις επιτροπές συμφιλίωσης θα μπορούσε ο διαμεσολαβητής να τον δούμε με ένα ρόλο πολύ ενεργό. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστούμε. Ο κύριος Μουρίτς από το Μαυροβούνιο έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας απευθύνω χαιρετισμό εκ μέρους της Εθνοσυνέλευσης του Μαυροβουνίου και της Επιτροπής ε, πολιτικών δικαιωμάτων και να σας ευχαριστήσω για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Θα ήθελα επίσης βεβαίως να σας απευθύνω και προσωπικά χαιρετισμό. Η Επιτροπή Ατομικών Ελευθεριών και Δικαιωμάτων του Μαυροβουνίου αναδεικνύει την ανάγκη πολύμορφη συνεργασίας μεταξύ όλων των φορέων εμπλεκόμενων ε, και στο Μαυροβούνιο ε, βρίσκονται σε εφαρμογή μια σειρά από μέτρα για τη βελτίωση της θέσης των Ρωμά. Κατά την σύνταξη του ετήσιου προγράμματος εργασιών μας, βασιζόμαστε πάντοτε στα συμπεράσματα που λαμβάνουμε από την Κομισιόν για το Μαυροβούνιο, ιδίως όσον αφορά τα συμπεράσματα και τις συστάσεις που λαμβάνουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τη θέση των μειονοτήτων. Εμείς λοιπόν υλοποιούμε αυτές τις συστάσεις της Κομισιόν όσον αφορά τη βελτίωση της θέσης των Ρωμά. Αυτό έχει αποφέρει αποτελέσματα και αυτό αναγνωρίζεται ακόμη και από διεθνείς οργανισμούς. Σε ψήφισμα του 2015 του Κοινοβουλίου του Μαυρο... Μαυροβουνίου συμπεριλαμβάνονταν εκείνα τα στοιχεία που ακριβώς μας έδωσαν τη δυνατότητα να βελτιώσουμε τη θέση των ε, ανθρώπων που ζουν στις, το, κοινωνίες, στις κοινότητες των Ρωμά. Τι, για ποιο λόγο. Ήταν ένα πρώτο βήμα να, το να εντοπιστούν τα ακριβή προβλήματα και εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι Ρωμά, κάτι που μας ε, βοήθησε ένα προς ένα να αρχίσουμε να τα αντιμετωπίζουμε. Βεβαίως χρειάζεται να γίνουν πολλά ακόμη, αλλά θέλω να σας δώσω ε, κάποια στοιχεία για, την, ε, για το εκπαιδευτικό σύστημα στο Μαυροβούνιο. Με τη βοήθεια του Υπουργείου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Δικαιωμάτων των Μειονοτήτων, το Μαυροβούνιο χρηματοδότησε την σύνταξη ενός λεξικού μαυροβουνιακού και ρωμανικού, δηλαδή έχουμε πλέον ένα δίγλωσσο λεξικό ε, που καλύπτει τις ε, δύο γλώσσες ε, που θα βοηθήσει και στην περαιτέρω ένταξη αυτών των ομάδων. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Βλέπετε ότι έχει περάσει ο χρόνος. Έχουμε πολύ λίγα λεπτά. Να περάσουμε στην Κορνέλια Έρνστ. Ευχαριστώ πολύ, Γιούντιτ. Πρέπει να πω ότι ότι με εντυπωσίασε ο Κροάτης συνάδελφος με τα όσα μας παρουσίασε. Εγώ πρόσφατα βρέθηκα στην Άπολη, ε, επισκέφθηκα καταβλισμό ε, τσιγκάνων και εκεί πραγματικά ε, η κατάσταση ήταν αποτρόπα, ήταν καταστροφική, δεν υπήρχε ούτε ρεύμα, ούτε νερό, ούτε εγκαταστάσεις ε, υγιεινής και μάλιστα οι αρχές μας είπαν ότι έτσι θέλουν να ζουν αυτοί. Δεν υπήρχε καν η δυνατότητα οι μη κυβερνητικέ οργανώσει να προσεγγίσουν τον καταβλητισμό αυτό. Τι θέλω να πω με όλα αυτά. Κάποιοι από εσά μιλήσατε για θεσμικό, διαρθρωμένο ρατσισμό. Αυτό είναι το πρόβλημα. Μπορούμε να δώσουμε εκατομμύρια, κονδύλια, δισεκατομμύρια που, που τάχα θα καταλήξουν στους Ρωμά. Όλα αυτά μπορείς να το κάνεις. Ξέρω ότι στην Τσεχία έχουν δοθεί εκατομμύρια ευρώ, τα οποία μάλιστα δεν αξιοποιήθηκαν. Γιατί, γιατί δεν θέλουμε να δώσουμε λεφτά στους Ρωμά. Αυτός είναι ε, ο θεσμικός, ε, ο θεσμοθετημένος ρατσισμός που πλήττει τους, ε, τους τσιγκάνους σε όλη την Ευρώπη. Οι απλές μας αρχές, ενώ έχουν δυνατότητες, δεν βοηθάνε τους Ρωμά. Επίσης, μιλήσατε για project. Χρειαζόμαστε εξειδικευμένα project κτλ. κτλ με άμεση πρόσβαση στα Ευρωπαϊ... στην ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Ξέρω ότι στην Ουγγαρία είναι τεράστιο το πρόβλημα Κάποιο Ρωμά να πάρει την οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, οποιαδήποτε οργάνωση ή ομοσπονδία Ρωμά. Δεν μπαίνει ποτέ ούτε φράγκο. Πείτε μας γι' αυτό. Και τέλος, απελάθηκαν χιλιάδες Ρωμά και από την ε, Γερμανία υπό την ε, πρόφαση ότι το Κόσοβο είναι ασφαλής χώρα προέλευσης. Όλα αυτά στο πλαίσιο της προσφυγικής κρίσης. Ε, επιχειρήθηκε να στραφούν Ρωμά εναντίον προσφύγων. Και τι έγινε. Ασχολούμαστε τάχα με τους πρόσφυγες και ξαφνικά ξεχνάμε τους Ρωμά. Και όχι μόνο, όχι μόνο τους ξεχνάμε, γίνονται και θύματα πολλές φορές όλων αυτών των ρατσιστικών συζητήσεων ε, που διεξάγονται στις χώρες μας τα τελευταία χρόνια. Ευχαριστώ πολύ η κυρία Μαρσελίνα από την ε, Πορτογαλία. Ευχαριστώ. Δύο αναφορές, δύο σκέψεις. Θέλω να μιλήσω λιγάκι για τις ε, τσιγκάνες, τις γυναίκες. Ε, μιλήσαμε λιγάκι εδώ, αλλά πρέπει να εντάξουμε βεβαίως τους Ρωμά, κυρίως τις γυναίκες όμως, για να είναι αυτόνομες οι γυναίκες, χειραφετημένες μόνο όταν είναι χειραφετημένες θα έχουν ε, καλύτερα αποτελέσματα και θα βοηθήσουν και τα παιδιά τους να προχωρήσουν. Για να βοηθήσουμε τον πληθυσμό πρέπει πρώτα να βοηθήσουμε τις γυναίκες. Είναι οι γυναίκες, ε, οι τσιγκάνες που πρέπει να κερδίσουν την ισότητα. Πρέπει να τονίσουμε τη σημασία των τσιγκάνων γυναικών στην κοινότητά τους. Θα πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να τις εντάξουμε, κυρίως τις τσιγκάνες, γιατί θα ακολουθήσει και το υπόλοιπο του πληθυσμού. Θα ήθελα να δώσω και μια άλλη σκέψη, μια πληροφορία. Το Κοινοβούλιο της Πορτογαλίας ε, ξεκίνησε μια πρωτοβουλία, δημοσίευσε μια έκθεση για τον ρατσισμό και την ξενοφοβία και τον ε, ρατσισμό. Έτσι. Μέχρι τον Ιούλιο του 19 μέχρι το τέλος δηλαδή της θητείας μας, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, θα συνεργαστούμε με την ε, κοινωνία των πολιτών και με προσώπους ε, των Ρωμά και θα πρέπει όλα τα πολιτικά κόμματα της ε, Πορτογαλίας να δρομολογήσουν δράσεις για να βοηθήσουν τους Ρωμά. Γιατί προς αυτούς πρέπει να στραφούμε γιατί είναι οι πιο ευάλωτοι. Θέλω επίσης να τονίσω την ανάγκη ευρωπαϊκής χρηματοδότησης που θα πρέπει να είναι πολύ πιο σημαντική για τη στέγασή τους. Μιλήσαμε για τους ε, καταβλισμού Ρωμά, που είναι απλώς ε, τέντε μερικές φορές ή παράγκε που, ανθρώπων που ζουν σε άθλιε συνθήκες. Ε, δεν έχει νόημα να μιλάμε για απασχόληση όταν αν δεν ε, κάνουμε επενδύσεις στη στέγαση. Θα πρέπει το επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο να μας βοηθήσει να εστιάσουμε στην ε, πρόσβαση στη στέγη. Ευχαριστώ. Ο τελευταίος ομιλητής στον κατάλογο, ο Ρωμαίο Φρανς. Πριν σου δώσω το λόγο, Ρώμεο, θα ήθελα να σας πω σε όλους ότι θα δώσω ένα λεπτό στον καθένα, δεδομένης της ώρας. Θα είμαι πολύ αυστηρή. Και μετά η πρωταγωνίστρια μας σήμερα θα κλείσει τη σύνοδο την απογευματινή. Ρώμεο, έχεις το λόγο. Στρέφομαι προς τα κράτη-μέλη. Τα κράτη-μέλη πρέπει να θέσουν το, το ερώτημα στον εαυτό τους. Οι προσεγγίσεις μας είναι αντιπατριαρχικές. Έχουμε εμπιστοσύνη στους ίδιους τους Ρωμά και στις κοινότητες των Ρωμά εμπλέκουμε μέλη των κοινοτήτων αυτών στις δράσεις μας, τους αναγνωρίζουμε ως πολίτες. Έχουμε αναγνωρίσει ότι ο αντιαθηκανισμός αποτελεί πλήγμα ε, στα θεμέλια της δημοκρατικής μας κοινωνίας. Αν απαντήσουμε ναι, τότε βρισκόμαστε σε σωστό δρόμο. Αν όχι, τότε πρέπει να τα ξαναδούμε αυτά τα θέματα και να τα επανεπεξεργαστούμε. Η διαφθορά είναι μία από τους, ένας από τους σημαντικότερους λόγους για την μη επιτυχή υλοποίηση των στρατηγικών ένταξης των ε, Ρωμά. Μέσα από αυτήν τη διαδικασία, ωστόσο, ε, παράγονται και ε, σκλάβοι για, με εργαζόμενους που αμείβονται με 1,2 ευρώ την ώρα. Οι Ρωμά αποτελούν τον τελευταίο κρίκο της αλυσίδας της διαφοράς. Πρέπει να σπάσει η αλυσίδα αυτή. Πολλές φορές έχω την αίσθηση ότι όταν μιλάμε για Ρωμά είναι σχεδόν σαν να μιλάμε για άλλο είδος. Όχι, όχι για πολίτες που ζουν εδώ και αιώνες στις χώρες μας. Η, η, η εντύπωση αυτή δημιουργείται διότι η πλειοψηφική ε, κοινωνία κλείνει τα μάτια της στα πραγματικά προβλήματα των Ρωμά. Τα αγνοεί ενεργά, ενώ στην πραγματικότητα θα έπρεπε οι στρατηγικές από το στάδιο της θέσπισής τους, της εκπόνησής τους να είναι υποδειγμετικές και να λαμβάνουν υπόψη και να εμπλέκουν τους ίδιους τους δικαιούχους και τους αποδέκτες. Κρατήδια στη Γερμανία έχουν συνάψει συμβάσεις με οργανώσεις Σύντη και Ρωμά. Αυτό σημαίνει ότι πλέον είναι αναγκαίο στα αναλυτικά σχολικά προγράμματα να λαμβάνονται υπόψη και να διδάσκεται και η ιστορία των Ρωμά. Αυτό είναι ένα θετικό παράδειγμα. Εγώ, ξέρετε, έχω πάει και εγώ στην Κανεράτα και το, το επιβεβαιώνω. Οι Σύντι που ζουν εκεί στον καταβλισμό στην Ιταλία ε, έρχονται αντιμέτωποι με πραγματικό θεσμοθετημένο, θεσμοποιημένο ρατσισμό. Ευχαριστώ Ρώμεο. Επανέρχομαι στην, ε, στον κατάλογό μου η κυρία Βουσιλιούτε. Ένα λεπτό. Αν θέλετε να απαντήσετε μάλιστα σε κάτι, έχετε την ευκαιρία να το κάνετε. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Με μεγάλη χαρά ακούσαμε την ικανοποίηση, τη στήριξη που απευθύνεται προς ε, την ιδέα των Επιτροπών Αλήθειας και Συμφιλίωσης να επισημάνω δύο στοιχεία. Κάποιες φορές ο τρόπος με τον οποίο έχουν υλοποιηθεί οι στρατηγικές για τους Ρωμά μας δείχνουν ότι έχουν εφαρμόσει κάποια κράτη-μέλη ενδιαφέρουσες πολιτικές, όπως τα δημόσια έργα. Οπότε υπήρξε αυξημένη απασχόληση, αλλά με πολύ χαμηλέ ε, αμοιβέ. Ούτε καν τον κατώτατο δεν παίρνανε. Αυτό είναι ανησυχητικό. Δεύτερον, η συλλογή στοιχείων είναι νευραλική σημασίας. Ο Φρά ξέρει λοιπόν πώς να το κάνει αυτό, αλλά καλό θα ήταν να γίνουν όλα αυτά και σε εθνικό επίπεδο. Σαλβίνη στο BBC έλεγε ότι πρέπει να γίνει αυτό και ότι το ζητούν και τα κράτη-μέλη. Πρέπει λοιπόν να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε ό,τι αφορά τα στοιχεία και τα δεδομένα για του Ρωμά και για τη διασφαλίσεις. Πρέπει να δούμε κατά πόσο παρέχονται ποιοτικέ υπηρεσίε. Να παρακολουθούμε την κατάσταση και να υπάρχει λογοδοσία σε περίπτωση όπου δεν παρέχονται οι απαραίτητε υπηρεσίε. Ευχαριστώ, κύριο Σκάν. Ευχαριστώ. Έχουν φύγει οι συνάδελφοι από την Τσεχία, αλλά επισημαίνω να πω κάτι. είχαμε εξαιρετική ε, δραστηριοποίηση για τη στήρωση από πολλούς φορείς ε, στην Τσεχία ε, και κυβερνητικούς φορείς και μη. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να αναφέρουμε ανοιχτά. Όμως η εκπρόσωπος μίλησε για θετικά παραδείγματα στα μέσα ενημέρωσης. Εγώ το καλύτερο παράδειγμα που σας φέρω είναι αυτό της Τσεχίας, όπου ο πρόεδρος έκανε αρνητικές παρατηρήσεις για τους Ρωμά ε, οι Ρωμά ανταποκρίθηκαν, είπαν όχι εμείς εδώ είμαστε και δουλεύουμε. Μετά ε, το Ρωμαία που είναι ένα τσεχικό δίκτυο ενημέρωσης Ρωμά το ε, ανέδειξε. Υπάρχουν λοιπόν θετικά παραδείγματα. Συνήθως είναι κοντά μας, κάτω από τη μύτη μας και δεν τα βλέπουμε. Μπορούμε λοιπόν να τα βρούμε αν ψάξουμε λίγο καλύτερα. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε η κυρία Γιωβανόβιτς, παρακαλώ. Ευχαριστώ που μου, το συνάδελφο που μου δίνετε το λόγο. Όχι, παρότι δείχνετε ότι είστε έτοιμοι για πολιτικός, η πρόεδρος σας δίνει το ένα λεπτό. Ευχαριστώ, αστείευουμε φυσικά. Ευχαριστώ, ε, Κλοντ, που ανέφερε σε αυτό το επιχείρημα για τα μέσα ενημέρωση και έτσι μπορώ εγώ να σταθώ στην ισότητα των φίλων, γιατί είναι κάτι το οποίο με προβληματίζει ε, ιδιαίτερα τελευταία. Βλέπουμε ότι το πολιτικό αφήγημα ε, για τον αντιαθηγενισμό σπάνια στέκεται στην ισότητα των φίλων. Και όταν μιλούμε για φύλλα, δεν πρέπει να μιλούμε μόνο για τις γυναίκες. Φανταστείτε πώς είναι η κατάσταση για έναν Ρωμά ε, που ταυτόχρονα είναι λεσβή ομοφιλόφιλος ή ομοφιλόφιλοι. Επομένως και έτσι δημιουργείται ένα επιπρόσθετο επίπεδο δυσκολίας ε, στο πλαίσιο της κοινωνίας. Οι αναγκαστικές θυρώσεις δεν στόχευαν ε, άντρες Ρωμά, αλλά γυναίκες Ρωμά. για να μην ε, αναπαράγεται ο πληθυσμός ε, των Ρωμά. Πρέπει λοιπόν να δούμε πώς ε, μπορούμε να ενσωματώσουμε και αυτή τη διάσταση στην χάραξη και υλοποίηση πολιτικής. Αυτό είναι πολύ σημαντικό καθήκον. Ευχαριστώ. Προς τους διερμηνείς μια έκκληση. Ένα λεπτό ακόμα για τον κύριο Κατσαϊσή και μετά Ξέρω ήδη ότι έχουμε ξεπεράσει το χρόνο. Ένα λεπτό και μετά οι υπόλοιποι στα αγγλικά. Παρακαλώ κύριε Κατσάηση. Ευχαριστώ. Φέτος συμπληρώσαμε χίλια χρόνια μετανάστευσης των Ρωμά. Η Ρωμά είναι μειονότητα σε διάφορες χώρες. Και μέχρι να φτάσουμε να έχουμε ποσοστώσεις για έδρες στα εθνικά κοινοβούλια, μέχρι να εκπαιδευτούν ε, όλος ο πληθυ... να εκπαιδευτεί όλος ο πληθυσμός, θα πρέπει να έχουμε ποσοστώσεις. Γιατί αλλιώς δεν θα αλλάξει τίποτα. 15 χρόνια συζητάμε εθνικές στρατηγικές, εθνικά προγράμματα, στρατηγικές πλαίσιο, αλλά τίποτα δεν έχει αλλάξει, τίποτα δεν έχει γίνει. Θέλουμε να κάνουμε κάτι για τους Ρωμά, αλλά αυτά που έχουμε κάνει είναι πολύ, είναι πολύ λίγα. Πόσους Ρωμά έχουμε εντάξει, ελάχιστους. Σταματούμε εδώ τη διερμηνία. Ε, θα ακούσετε τη για Πόστ χωρίς διερμηνία στα αγγλικά. Post.